10. Dear colleagues, probably we can uh, start. Αγαπητοί συνάδελφοι, μπορούμε να ξεκινήσουμε με κάποια καθυστέρηση. Το πρώτο είναι η έγκριση της ημερήσιας διάταξης. Μετά το αίτημα του εισηγητή και των σκιωδών για να επιτραπεί η τελική επεξεργασία των ε, συμβαστικών τροπολογιών και οι συζήτηση μεταξύ των πολιτικών ομάδων, η ψηφοφορία για το σημείο 14 γενετικά τροποποιημένοι οργανισμοί αναβάλλεται για τις 14 Νοεμβρίου το πρωί. Σύμφωνα με τους εισηγητές, τα 18 και 19 θα αντιστραφούν. Και αν δεν υπάρχουν αντιρρήσεις, μπορούμε τώρα με αυτές τις τροποποιήσεις να εγκρίνουμε το σχέδιο ημερήσιας διάταξης. Εντάξει. Σημείο 2. Ανακοινώσει του Προέδρου. Λοιπόν, για το High Look θα αλλάξει το χρονοδιάγραμμα. Το Συμβούλιο ζήτησε να αναβληθεί η υποβολή της ε, πρότασης του Συμβουλίου για την 1η Ιανουαρίου αντί να μας το στείλουν για την Ολομέλεια του Νοεμβρίου όπως είχε αρχικά προβλεφθεί. Ο λόγος για αυτό το αίτημα είναι ότι το Συμβούλιο θα προτιμούσε η διαδικασία δεύτερης ανάγνωσης να γίνει υπό την επερχόμενη Λετωνική Προεδρία. Ο εισηγητής κ. Στόλτβαλτ δεν ήταν υπέρ αυτή της περαιτέρω καθυστέρησης ε, στη διαδικασία, αλλά μετά από διαβούλευση με τους ε, σκιόδης αποφάσισε να αποδεκτεί αυτό το αίτημα του Συμβουλίου σε ένα πνεύμα καλής ε, διοργανικής συνεργασίας. Το νέο χρονοδιάγραμμα θα έχει ως εξής. Ανακοίνωση της θέσης του Συμβουλίου στην Ολομέλεια, πρώτη Ολομέλεια του Ιανουαρίου. Εξέταση του σχεδίου σύστασης στην ΕΝΒΗ 21-22 Ιανουαρίου. Προθεσμία για τροπολογίες 27 Ιανουαρίου. Ψηφοφορία στην ΕΝΒΗ 23-24 Φεβρουαρίου. Ψηφοφορία στην Ολομέλεια. Στη δεύτερη Ολομέλεια του Απριλίου. Ο εισηγητής ωστόσο έχει ζητήσει το λόγο. Ευχαριστώ. Είμαι κάπως απογοητευμένος γιατί χθες μιλήσαμε με κάποιον που μας είπε ότι το Συμβούλιο είπε ότι αυτή η καθυστέρηση οφείλεται στο Κοινοβούλιο, κάτι που δεν ισχύει. Η πολιτική συμφωνία στο Συμβούλιο έγινε στις 3 Ιουνίου, πριν από πέντε μήνες δηλαδή. Και έκτοτε αυτοί οι εργούν Και αυτό είναι απαράδεκτο. Πρόεδρος, όπως είπα στην ανακοίνωσή μου, είναι έτοιμα από πλευράς του Συμβουλίου πρέπει να είναι σαφές ότι η απόφαση για αναβολή προέρχεται από το Συμβούλιο. Δεύτερη ανακοίνωση. Η επόμενη συνεδρίασή μας θα γίνει τη Δευτέρα 10 Νοεμβρίου το απόγευμα και θα παραταθεί και Τρίτη 11 Νοεμβρίου το πρωί για να ψηφίσουμε την έκθεση της κυρίας Ράις για τους γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς και να κάνουμε ανταλλαγή απόψεων με τον νέο Επίτροπο για την Κλιματική Αλλαγή και την Ενέργεια, κύριο Άρια Κανιέτε. Και καταργείται η συνεδρίασή μας στις 13 Νοεμβρίου 5η το απόγευμα. Και μια έκτακτη συνεδρίαση της Επιτροπής μας προβλέπεται για τη Δευτέρα 24 Νοεμβρίου από τις 7 έως τις 10 στο Στρασβούργο για να ψηφίσουμε την έκθεση Νίκολσον για τα νέα τρόφιμα. Τώρα, ανακοίνωση για το σχέδιο χωρίς γραπτά έγγραφα. Ζητήσαμε από τα πλήρη μέλη, τα τακτικά μέλη της Επιτροπής μας, αν θέλουν να, λαμβάνουν, να συνεχίσουν να λαμβάνουν ένα πλήρη φάκελο γραπτών εγγράφων και λαμβάνουμε υπόψη ότι μόνο τρεις το ζήτησαν αυτό. Οπότε θεωρούμε ότι πρέπει η Επιτροπή μας να παίξει ηγετικό ρόλο για να στη μείωση της χρήσης χαρτιού. Θα μπορούσαμε το 2015 να ξαναδούμε την κατάσταση και να εξετάσουμε αν μπορούμε να καταργήσουμε τα γραπτά έγγραφα όπως έχει κάνει η έμπλα από την αρχή της θητείας. μια συνεδρίαση για τα μέλη και τους βοηθούς για τη χρήση του e-committee θα γίνει σήμερα 2 με 3 σε αυτήν εδώ την αίθουσα. Διερμηνία έχουμε σήμερα μόνο 21 γλώσσες, δεν έχουμε αστωνικά και μαλτέζικα. Ως συνήθως έχετε ηλεκτρονικά τα έγγραφα στο e-committee και η συνεδρίαση μεταδίδεται ζωντανά από το ίντερνετ. Ανακοίνωση των αποφάσεων των συντονιστών 13 Οκτώβρη. Οι συντονιστές απέστειλαν ηλεκτρονικά τις συστάσεις τους, τα αποτελέσματα της συνεδρίασής τους 13 Οκτώβρη. Αν δεν υπάρχουν αντιρρήσεις μπορούμε να θεωρήσουμε ότι εγκρίθηκαν. Ωραία, εντάξει. Έγκριση πρακτικών προηγούμενων συνεδριάσεων. Εάν δεν υπάρχουν αντιρρήσεις, μέχρι τέλους της συνεδρίασης, τα πρακτικά της συνεδρίασης 24, 24 και 25 Σεπτεμβρίου θα θεωρηθεί ότι ενεκρίθησαν. Εντάξει. Λοιπόν, κάτι ακόμη. Να σας ενημερώσω για τις συνεχιζόμενες διοργανικές διαπραγματεύσεις. Λοιπόν, είχαμε τριμερή διάλογο για την παρατήρηση και υποβολή εκθέσεων για την τροποποίηση του κανονισμού για τις εκπομπές οξυδίων του άνθρακα από την αυτιλία. Στην πρώτη συνάντηση εκφράστηκε ετοιμότητα όλων των ε, θεσμών να καταλήξουν σύντομα σε συμφωνία κατά τη δεύτερη ανάγνωση μετά από δύο τριμερείς διαλόγους και δύο τεχνικές συναντήσεις. Υπήρξε ανταλλαγή απόψεων για τα πολιτικά θέματα που εκκρεμούν, το Συμβούλιο αποδέχτηκε μια σειρά τροπολογιών από την πρώτη ανάγνωση του Κοινοβουλίου και ε, για το θέμα των μεταφορών έχουμε ακόμη ανοιχτά θέματα. Η δεύτερη συνάντηση για τον τριμερή διάλογο θα γίνει στις 18 Νοεμβρίου. Δεύτερο θέμα, μείωση κατανάλωσης πλαστικό, για πλαστικές σακούλες. Στον πρώτο τριμερή διάλογο στις 14 Οκτωβρίου όλα τα όργανα εξέφρασαν την ετοιμότητά τους να διαπραγματευτούν και να καταλήξουν σε μια ε, πρόορη ε, συμφωνία στην ε, δεύτερη ανάγνωση. Ζητήσαμε από το Συμβούλιο να μας εξηγήσει τη θέση του και να μας πει σε ποια σημεία υπάρχει ενδεχόμενο συνένεση, ιδιαίτερα όσον αφορά τις εκστρατείες για την ενημέρωση του κοινού. Χρειάζεται επίσης μια ε, ανάλυση σε βάθος των τροπολογιών που έγινε σε έναν τεχνικό διάλογο. Χθες είχαμε την δεύτερη συνεδρίαση όπου είδαμε που μπορούμε να καταλήξουμε σε συμβασμούς. Οι συμβασμοί έγιναν αποδεκτοί και ο συγητής υπέβαλε κάθε συνεδρίαση ορισμένες προτάσεις για να διευκολύνει την ε, διατύπωση περαιτέρω αποδεκτών συμβασμών. Η επόμενη τεχνική συνεδρίαση θα βοηθήσει την προώθηση των προτάσεων για να προσπαθήσουμε να καταλήξουμε σε μια σφαιρική συμφωνία στην τρίτη συνεδρίαση τριμερούς διαλόγου που προβλέπεται στις 13 Νοεμβρίου. Συγγνώμη, 17. 17 Νοεμβρίου. Και τώρα. Επόμενο θέμα. Έκθεση του κυρίου James Nicholson για τα νέα τρόφιμα. Έχουμε λάβει 393 τροπολογίες στην Επιτροπή μας, 276 στην Άγκρη και 96 στην Ίντα. Οπότε έχουμε δουλειά μπροστά μας. Να δώσω πρώτα το λόγο στον εισηγητή κύριο Νίκολσον. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Έχουμε ένα τεράστιο καθήκον ενωπιών μας σε αυτό το συγκεκριμένο φάκελο και φυσικά θα γνωρίζετε το ιστορικό των προτάσεων για τα νέα τρόφιμα. Ήταν ιδιαίτερα πολύπλοκο και πραγματικά ακολούθησε μια δύσκολη πορεία για να φτάσουμε εδώ που είμαστε σήμερα και δεν θα μας εκπλήξει που το επίπεδο της δέσμευσης των συναδέλφων αυτής της Επιτροπής ε, με ε, τόσες πολλές τροπολογίες ε, και θα ψηφίσουμε την άλλη εβδομάδα τις ε, τροπολογίες από την Άγκρα και την ΕΝΤΕ. Εγώ καλωσορίζω την, το επίπεδο της δέσμευσή ε, και είμαι σίγουρος ότι μπορούμε να πετύχουμε συμβιβασμό για τις τροπολογίες. Χθες συναντήθηκα με τους σκιώδεις εισηγητές για συναντήσουμε το πρώτο σύνολο των τροπολογιών που κατέθεσα. Είχα να κάνουν με τα άρθρα 1 και 2 ενώ μπορεί ε, να, εμφανίζονται περιορισμένα και ότι αντιμετωπίζουν μόνο δύο άρθρα. Εγώ νομίζω ότι κάναμε πολύ σημαντική πρόοδο δεδομένου ότι το άρθρο 2 σε σχέση με τον ορισμό του νέου τροφίμου είναι ένα από τα κύρια σημεία της πρότασης αυτής. Ε, βρήκαμε ευρεία συνένεση για την επενσαγωγή των κατηγοριών ε, και στην πλειοψηφία των περιπτώσεων Αυτές οι κατηγορίες ε, θα έπρεπε να προσδιοριστούν πλήρως. Ε, θα πρέπει να υπάρχει μεγαλύτερη σαφήνεια στις κατηγορίες και για τους καταναλωτές και για τους παραγωγούς ε, και πραγματικά με ενθαρρύνει το επίπεδο συμφωνία το οποίο καταλήξαμε χθε. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν και κρεμή ζητήματα, κυρίως ό,τι φορά τα ανανοηλικά, Ξέρω ότι οι συνάδελφοι τουλάχιστον από τέσσερι ομάδε του Κοινοβούλου έχουν ισχυρέ απόψει για τι προτάσει Κομισιόν και θέλω να δράξω την ευκαιρία, ίσω για να ζητήσω από την Κομισιόν κάποιε διευκρινήσει και να μα πει τι σκεφτείτε για τι τροπολογίε που έχουν κατατεθεί για τα νανοηλικά και ιδίω σε σχέση με το να αποσύρουμε το κανονισμό στις αναφορές ε, στο κανονισμό 1196 και 20 του 2011 να μας πούν ε, τι πεδίο προβλέπουν για να καταλήξουμε σε συμβιβασμό. Επίσης ε, πρέπει να δούμε τι συμβαίνει με τις τρίτες χώρες και νομίζω ότι μπορούμε να πούμε ότι όλοι οι σκιώδεις συμφωνούν ότι η διάταξη ότι ένα παραδοσιακό ε, τρόφιμο μιας παραδοσιακής δίαιτας ενός τμήματος του πληθυσμού χρειάζεται να διευκρινιστεί περαιτέρω. Και ενώ συμφωνήσαμε ότι θα πρέπει να υπάρχουν κατευθυντηρίες γραμμές για να βοηθήσουμε τους ενδυνάμει ετούντες, ε, πρέπει ο κανονισμός ρητά να αντιμετωπίσει αυτό το θέμα στο ίδιο το άρθρο 2. Και πάλι θέλω να δράξω την ευκαιρία για να ζητήσω από την Κομισιόν να μας εξηγήσει το σκεπτικό της για ε, τον large or significant και αυτοί οι όροι, οι οποίοι μπορεί να φαίνονται αθώοι, μπορεί να έχουν τεράστιες συνέπειες για τον όρο της ασφαλούς ε, χρήσης, για το ιστορικό ασφαλούς χρήσης. Και σε ό,τι αφορά τα τρόφιμα από τι χώρες. Ε, θα υπάρχουν ε, φυσικά και συζητήσεις ε, για την προστασία των δεδομένων, της της πράξης και τις προθεσμίες για τις διαδικασίες. Νομίζω πάντως ότι μπορούμε να σημειώσουμε πρόοδο σε πολλά θέματα καθώς ε, όπως είπατε και εσείς ε, πρόεδρε έχουμε την ψηφοφορία στις 24 στο Στρασβούργο και εγώ θα διασφαλίσω ότι αυτή η ψηφοφορία θα διέπεται από όσο το δυνατόν περισσότερους συμβιβασμούς μέχρι τότε όμως ε, μην απατάστε έχουμε πάρα πολλή δουλειά μπροστά μας έχουμε κάνει μια καλή αρχή και θέλω να ευχαριστήσω τους σκιώδεις εισηγητές για την επικοδομητική τους δέσμευση χθε και ελπίζω να συνεχίσουμε με από τις επόμενες εβδομάδες. Το μόνο άλλο θέμα ε, έχω μια ανταλλαγή με το, απόψεων με το Συμβούλιο σήμερα και ελπίζω και εκεί να έχουμε επιτυχία έκβαση. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Και τώρα θα ξεκινήσουμε τον πρώτο γύρο με τους σκιώδεις εισηγητές. Η κυρία Γιούσο, παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ και τον εισηγητή για τις εξηγήσει του. Εγώ, κατόπιν αυτών, δεν έχω να προσθέσω πολλά. Πολύ καλά. Πολύ καλή μου φαίνεται η έκθεση του κυρίου Νίκολσον και εγώ δεν παρουσίασα καμία τροπολογία. Παρ' όλα αυτά ε, υπήρχε μια χιονοστιβάδα τροπολογιών, όμως αφορούν όλες ε, τα ίδια θέματα επί των οποίων συζητάμε και είμαι σίγουρη ότι θα φτάσουμε στη συνένεση. Χτες ήδη σημειώσαμε μεγάλη πρόοδο στη συνάντησή μας και όπως είπε και ο κύριος Νίκολσον, και εγώ θα ήθελα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μας εξηγήσει, να μας δώσει περισσότερες πληροφορίες για το θέμα των ανοηλικών. Για το τι είναι το ιστορικό ασφαλούς χρήση, τι είναι η ασφαλής χρήση και μιλάμε και για κάποιες λέξεις, ε, το larger significant είναι λέξεις πάρα πολύ ευρύ και νομίζω ότι θα πρέπει να τι εξηγήσουμε ή να βρούμε άλλε λέξει και για τι εκδοκισιδότηση πράξει και για τι εκτελεστικέ πράξει. Θα ήθελαμε και εκεί κάποιε εξηγήσει. Και να πω και το εξή. Στην νομοθεσία που έχουμε τελευταία, κατά την άποψή μου γίνεται μια κατάχρηση των κατεξοδοτήσεων πράξεων και των εκτελεστικών πράξεων. Και Αυτό μας οδηγεί στο να έχουμε κάποια ανασφάλεια, γιατί εγκρίνουμε μια νομοθεσία και κατόπιν με αυτά τα δύο νομοθετικά μέσα ε, τροποποιεί η Κομισιόν την νομοθεσία πολύ ουσιαστικά. Θα θέλαμε λοιπόν κάποιες εξηγήσει για αυτό το θέμα και επίσης να ζητήσω στο μέλλον τέτοιες νομοθετικές πράξεις ε, να χρησιμοποιούνται μόνο για πράγματα τα οποία είναι απαραίτητα. Και όχι για να αφήνουμε κατά κάποιο τρόπο ανοιχτή την νομοθεσία. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ο Αντιπρόεδρος Πολπότης. Ευχαριστώ. Καταρχήν, να πω ότι μετά τη χθεσινή συγκεντρία των σκηνών συγγητών είμαι σίγουρος ότι μπορούμε να καταλήξουμε σε συμβιβασμούς και ότι μπορούμε να έχουμε μια κοινή θέση. Αλλά θα ήθελα να αναφέρω ορισμένα πράγματα που νομίζω πρέπει να αντιμετωπιστούν στην έκθεση. Ορισμένα είδη βέβαια αντιμετωπίζονται. Καταρχήν πρέπει να δούμε τι γίνεται με τους κλόνους ε, από τα ζώα. Ο στόχος της δουλειάς μας είναι η συγκεκριμένη νομοθεσία για τρόφιμα που προέρχονται από κλωνοποιημένα ζώα και του απαγόνους τους να χρησιμοποιήσουμε συγκεκριμένα μέτρα για να αποφύγουμε οποιοδήποτε ρυθμιστικό κενό. Νομίζω ότι αυτό είναι σαφές, γιατί είχαμε μπροστά μα την TTIP και είναι απολύτω βασικό να αντιμετωπίσουμε αυτό το θέμα. Πριν ε, η όλη διαδικασία διαπραγμάτευσης ε, για το θέμα της κλωνοποίησης ολοκληρωθεί. Ένα δεύτερο θέμα είναι το ιστορικό ασφαλούς χρήσης, όπως αναφέρει και ο συγητής. Συμφωνώ ότι η βάση για το θέμα αυτό είναι να έχουμε και επιστημονικές κατητήρε γραμμές από την Κομισιόν ή από την ΕΦΣΑ. Θα δούμε πώς ε, θα χειριστεί το θέμα η Κομισιόν. Ε, ίσως προετοιμαστούν ε, κάποιες κατηγορίες γραμμές από την Κομισιόν ή από την ΕΦΣΑ αλλά συμφωνώ με τον εισηγητή και τους υπόλοιπους κοιότητες ότι πρέπει να έχουμε τέτοιες κατευθυντήριες γραμμές. Κατόπιν έχουμε το θέμα των ενοηλικών στο τρόφιμα. Είναι κάπως δύσκολο αυτό το θέμα γιατί έχουμε έναν ορισμό που βασίζεται στην επισήμανση στην πρόταση και που λειτουργεί με ένα κατόφυλλο 50% για τα ενοηλικά στα τρόφιμα. Σύμφωνα με τη γνώμη της ΕΦΣΑ από το 2012, κάτι τέτοιο δεν είναι δυνατόν ε, για ε, τα τρόφιμα και προτείνει η ΕΦΣΑ κατόφλι 10%. Όμως ε, δεν έχουμε μεθόδους ανείχνευσης για τέτοια κατόφλια, επομένως είμαι πεπισμένος ότι θα πρέπει να εισαγάγουμε ή εγώ τέλος πάντων έχω παρουσιάσει μια πρόταση να τα βασίσουμε αυτά στις ε, διαδικασίες, ε, τεχνολογικές διαδικασίες ε, οι οποίες μπορεί να αυξήσουν τα νανοηλικά στα τρόφιμα. Δηλαδή πρέπει να επικεντρωθούμε σε κάποιες διαδικασίες που μπορεί να προκαλέσουν ή να εισαγάγουν τέτοια νανοηλικά στα τρόφιμα. Ελπίζω ότι θα μπορέσω να πείσω και τους υπόλοιπους σκιώδεις, συζητητές, και τον εισηγητή να ακολουθήσουμε αυτό το σκεπτικό. Και το όποιο θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Συγητή για την εισαγωγή των κατηγοριών. Είναι πολύ σημαντικό για λόγους και νομίζω ότι και εδώ μπορούμε να φτάσουμε σε μια ισορροπημένη θέση μέχρι να μπορέσουμε να εισαγωγούμε και ποια ίσονοσημασία σημασία ζητήματος, ζητήματα όπως παραδείγματος χάρη το θέμα της καλλιέργειας ιστών που δεν περιλαμβάνεται και ιδιαίτερα τώρα. Ελπίζω λοιπόν ότι θα μπορέσουμε να συζητήσουμε περαιτέρω τις τροπολογίες ε, για τα θέματα αυτά και νομίζω ότι και το κρέας που ε, προέρχεται από τεστ ε, στο Σολίνα θα το συμπεριλάβουμε εκεί, τεστ tube meat. Επίσης, για το θέμα των κατεξουσιοδότηση πράξεων και των εκτελεστικών πράξεων, πάντα υπάρχει σύγκρουση μεταξύ Συμβουλίου και Κοινοβουλίου γι' αυτό. Κατά την άποψή μου, δεν ε, είναι αποδεκτό να έχουμε εκτελεστικές πράξεις ε, για το θέμα του ορισμού του νέου τροφίμου, ούτε για την προσαρμογή του καταλόγου όταν χρειάζεται έγκριση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, παραδείγματο χάρη σε περίπτωση πρόσθετων ε, υλικών, ενζήμων ε, και αρτημάτων. Και νομίζω ότι το ίδιο θα πρέπει να ισχύει όταν μιλάμε για το νέο τρόφιμα. Είναι σαφές ότι θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε το μοντέλο αυτό. Επίσης, είμαι πολύ ικανοποιημένο που κατορθώσαμε να βάλουμε και την έννοια της ευμερίας και της υγείας των ζώων και την αρχή της πρόληψης. Και επίση χαίρομαι που μπορούμε να συνεργαστούμε με τον εισηγητή και του σκιώδες με τον τρόπο αυτό και είμαι πεπισμένος ότι εν τέλει θα μπορέσουμε να φτάσουμε σε μια κοινή θέση. Σα ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Τώρα για τους φιλελεύθερους. Μαρή Πόλτσα. Ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ και τον εισηγητή κύριο Νίκολσον για την θαυμάσια πραγματικά έκθεση. Θαυμάσια δουλειά έκανε και ως Ευρωβουλευτής στη σύνταξη εκθέσεως αλλά και ως διαπραγματευτής πραγματικά επαγγελματι... επαγγελματίας. Χαίρομαι που επανέρχονται οι κατηγορίες στο κείμενο, διότι η πρόταση της Κομισιόν ήταν ασαφής, ήταν αόριστη. Και ήταν δύσκολο να αποκρισταλώσει κανείς, να καταλήξει κάπου, πού πήγαιναν, πού το πήγαιναν δηλαδή. Και αν ήταν κάτι κάτω από το κατόφλι ή πάνω. Και αυτό φαίνεται ωστόσο να εξακολουθεί να είναι το πρόβλημα όταν μιλούμε για εισαγωγές από τρίτες χώρες. Θα επανέλθω σε αυτό. Πάντως είναι καλό που επιτύχαμε την συμπερίληψη σαφών κατηγοριών. Χρειαζόμαστε άραγε περισσότερες. Αυτό είναι ένα ερώτημα και μπορεί να αντεχθεί επιτάπητος για να μπει στο περιεχόμενο ενός συμβιβασμού. Την κλωνοποίηση εγώ δεν θέλω να την περιλάβουμε στον κανονισμό. Αντίθετα από αυτά που ακούσαμε βρίσκω ότι το θέμα αυτό είναι τόσο αμφιλεγόμενο, τόσο εξειδικευμένο, που είναι σημαντικό πρώτα να έχουμε την απαραίτητη σαφήνεια, να μην υπάρξει σύγχυση, να κάνουμε προσπάθεια δηλαδή να επεξεργαστούμε την πρόταση που έχουμε λάβει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή καταρχήν διότι από τα πιο αμφιλεγόμενα θέματα σε όλη την ιστορία και πάντως όλα τα χρόνια που δουλεύω εγώ στο θέμα αυτό δεν έχω δει αντιθέσεις του είδους που βλέπουμε τώρα Ενώ, δηλαδή πάντα γύρω από το θέμα της κλωνοποίησης στον αρχικό συμβασμό που πετύχαμε χθες Υπάρχει και μια διατύπωση που λέει ότι υπό ορισμένε περιστάσεις το νέο τρόφιμο θα πρέπει να δοκιμάζεται και να εξετάζεται και η επίπτωση που μπορεί να έχει στο περιβάλλον. Διότι οι νέες τεχνολογίες δεν έχουν μονάχα επιπτώσεις στη δημόσια υγεία. Οι νέες τεχνολογίες Εγώ τις δέχομαι και θεωρώ ότι τις χρειαζόμαστε και πρέπει να έχουμε την τόλμη να δοκιμάζουμε νέα πράγματα. Ωστόσο, να παρακολουθούμε πάντα προσεκτικά ποιε μπορεί να είναι οι επιπτώσεις και στον οργανισμό μας αλλά και στο περιβάλλον μέσα στο οποίο ζούμε. Άρα, η περιβαλλοντική εξέταση, εν προκειμένου, είναι μια σημαντική πτυχή Σε ό,τι αφορά τώρα τη λήψη αποφάσεω, και εδώ έχουν σχέση και οι εκτελεστικέ ή κατεξουσιοδότηση πράξει, θα πρέπει να προσπαθήσουμε να βασιστούμε σε ανεξάρτητα και μετρήσιμα επιστημονικά αποτελέσματα. Δεν μπορούμε να προχωρήσουμε με μια τυφλή πίστη επιμένοντας σε χωρίς να έχουμε πρώτα όλες τις απαραίτητες εμπειρικές ενδείξεις που είναι απαραίτητες. Και ο, ο ρόλος της ΕΦΣΑ εν προκειμένου θα είναι πολύ σημαντικός. Και αυτό ίσως πρέπει να το τονίσουμε και πάλι. Τώρα, να δούμε ποια θα είναι τα επόμενα βήματα. Ο ορισμός των εισαγωγών από τρίτες χώρες πρέπει να μας απασχολήσει. αφού δεν είναι θέμα μοναχά νέων τροφίμων, είναι νέα τρόφιμα στην ευρωπαϊκή αγορά. Διότι εδώ εμείς απαιτούμε να έχουν χρησιμοποιηθεί αυτά τα τρόφιμα, από, να καταναλωθεί δηλαδή από μεγάλο αριθμό ανθρώπων για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Αυτό τι σημαίνει τώρα, μιλούμε για μια συγκεκριμένη χώρα ή για μια περιφέρεια. Και ποια είναι η διαφορά τώρα μεταξύ μιας μικρής χώρας όπως για παράδειγμα το Λουξεμβούργο και μιας πολύ μεγάλη όπως η Βραζιλία. Καλά, τέλος πάντων το Λουξεμβούργο βεβαίως είναι και μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το γνωρίζω, αλλά βάζω ένα παράδειγμα γιατί ε, αυτή τη στιγμή είναι μια μικρή χώρα που με έρχεται αυτόματα στο μυαλό. Ε, πού βρίσκεται το στοιχείο της ασφάλειας εν προκειμένου. Εξακολουθούν να υπάρχουν αβεβαιότητες και νομίζω ότι αυτές πρέπει να τις αντιμετωπίσουμε. Και επιμένω ότι δεν πρέπει να χρησιμοποιήσουμε οποιοδήποτε εργαλείο για να ορθώσουμε προστατευτικά τείχη. Υπάρχουν ωστόσο δύο, συγκεκριμένες, δύο συγκεκριμένοι στόχοι. Να προχωρήσει η οικονομία δηλαδή, να αρχίσει, να ξαναπάρει μπρος η οικονομία και Αναπόσπαστο μέρος αυτού είναι η μείωση της γραφειοκρατίας και η προσφορά περισσότερων και καλύτερων ευκαιριών, ιδίω για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, ώστε να ξανασταθούν στα πόδια τους, να αρχίσουν να αναπτύσσονται, να μπορέσουν να χρησιμοποιήσουν και να υιοθετήσουν νέες τεχνολογίες, μεθόδους παραγωγής κ.ο.κ. Σας παρακαλώ λοιπόν, όταν θα διεξέλθουμε την πρόταση αυτή κανονισμού, να μην λησμονούμε ότι χρειάζεται σαφήνεια, και απλές διατυπώσεις. Αυτά είναι απαραίτητο να τα έχουμε πάντα υπόψη ότι απότερο στόχος μας είναι η διευκόλυνση της ζωής των πολιτών. Λίγα σχόλια κύριε Πρόεδρε, αφού υποστηρίζω τα πιο πολλά από όσα λέχθηκαν μέχρι τώρα. Αναμένουμε νέα συμβαστική τροπολογία για τις κατεξουσιοδότηση πράξης, γιατί εμείς δεν δεχόμαστε τη λίστα των νέων τροφίμων όπως εφαρμόζεται με τέτοια πράξη. Όπως είπα συμφωνώ με πολλά από αυτά που ακούστηκαν. Πολλές τροπολογίες έχουν κατατεθεί και ζητούν από την ΕΦΣΑ να υποβάλει γνωμοδότηση σε κάθε περίπτωση. Αυτό λοιπόν το ΜΕΙ, τη δυνητική διατύπωση, να την αντικαταστήσουμε με το ΣΑΛ, με οριστική ε, διατύπωση. Σε ό,τι αφορά την επισήμαση δεν αρκεί μονάχα ο σχετικός κανονισμός. Πρέπει να υπάρχει και αξιολόγηση του κινδύνου και να διασφαλίσουμε ότι σημειώνονται όλα τα είδη νανοηλικών. Και τέλος για την κλωνοποίηση θυμούμε τον τριμερή διάλογο στην προηγούμενη κοινοβουλευτική θητεία που είχαμε περάσει όλη τη νύχτα. Και ακόμη και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αλλά και ορισμένες χώρες μέλη επέμεναν ότι πρέπει να απαγορεύεται μονάχα η κατανάλωση κρέατος του κλωνοποιημένου ζώου. Βεβαίω όλοι συμφωνούσαν με αυτό, διότι κάτι τέτοιο είναι εξαιρετικά δαπανηρό πρώτα-πρώτα. Και αυτό ήταν εντελώ γελίο το επιχείρημα όταν μιλούμε για προστασία ζώων κλπ. Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι θα περιληφθούν και οι απόγονοι του κλωνοποιημένου ζώου. Γιατί αν δεν γίνει έτσι τότε ξεχάστε, δεν υπάρχει λόγος να προχωρήσουμε σε κανονισμό. Κυρίως πρόκειται για το offspring, κυρίως πρόκειται για τους απογόνους και όχι για το ίδιο το κλωνοποιημένο ζώο. Βρισκόμαστε μπροστά στον κίνδυνο να υπάρξει ένα κενό και χρειαζόμαστε κάποια νομοθετική ρύθμιση. και υποστηρίζουμε τη θέση σας. Αυτά από την πλευρά μας για να μακρηγορήσουμε και περισσότερο. Σας ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος, για Μπόιλεν της Ενωτικής Αριστεράς. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ και τον εισηγητή. Η χθεσινή συνεδρίαση για τις σημαντικές τροπολογίες ήταν εξαιρετικά επιτυχής. Από τα πιο σημαντικά στοιχεία της εκθέσεως είναι του ορισμού του νέου τροφίμου. Εάν πρόκειται δηλαδή για νανοηλικά τα οποία προέρχονται από engineering, να δούμε που θα πει ο ορισμός. Και η αξιολόγηση κινδύνου, που αυτό πρέπει να είναι το περιεχόμενο του κανονισμού για τα νέα τρόφιμα. Έχουμε κάποιες ανησυχίες λοιπόν προκειμένου. Με ικανοποιούν και οι πολλές τροπολογίες που έχουν υποβληθεί από όλο το φάσμα της ε, Επιτροπής. Όλοι συμφωνούν ότι το 50% του κατοφλίου είναι κατάλληλα και ότι η γνωμοδότηση της ΕΦΣΑ που προβλέπει μόνο 10% κατόφλιο για νανοεφαρμογές δεν καλύπτονται από την αναφορά στο νομοθέτημα περί επισήμανσης. Ε, πολύ χαμηλότερο όριο. Χρειάζεται λοιπόν πολύ χαμηλότερο κατόφλι για να καθορίζονται τα νανοειδικά τα οποία είναι παρόντα μέσα σε νέα τρόφιμα και προέρχονται από engineering. Για αυτούς τους λόγους εμείς έχουμε υποβάλει τροπολογία που λέει ότι σε περίπτωση που υπάρχει αμφιβολία που προκαλείται από έλλειψη βεβαιότητας ή από έλλειψη δεδομένων πρέπει να εφαρμόζεται η αρχή της προφύλαξης και επομένως το νέο τρόφιμο δεν πρέπει να εισέρχεται στην ε, λίστα των εγκεκριμένων νέων τροφίμων. Πρέπει να, δεν μπορούμε να συνεχίσουμε να εγκρίνουμε νέα τρόφιμα εάν δεν είναι εξασφαλισμένο ότι είναι ασφαλή η ανθρώπινη κατανάλωση. Και υπάρχει και ένα άλλο σημαντικό θέμα και στις τροπολογίες που είναι αυτό της κλωνοποίησης. Όπως είπα και πριν, δεν νομίζω ότι μπορούμε να επιτρέψουμε μια κατάσταση όπου θα περάσει η ε, ρύθμιση για τα νέα τρόφιμα, αλλά δεν θα περάσει αυτή για την κλωνοποίηση και επομένως θα μείνουμε με ένα κενό στον νόμο, με ένα παράθυρο στον νόμο. Γι' αυτό πρέπει να πούμε ότι μέχρι ότου αρχίσει να ισχύει η οδηγία για την κλωνοποίηση που να καλύπτει τα κλωνοποιημένα ζώα και τους απογόνους τους δεν πρέπει να ισχύσει ο οργανισμός για τα νέα τρόφιμα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Για το EFTD κυρία Χέιβιν. Ευχαριστώ πολύ. Όταν μιλάμε για τα νέα τρόφιμα, είμαστε μπροστά σε ένα πολύ λεπτό θέμα, πρόκειται για ένα νέο θέμα. Είμαστε σε ένα εξερεύνητο πεδίο ουσιαστικά και επίσης εξελίσσεται συνεχώς. Γνωρίζουμε λοιπόν τι δεν είναι, αλλά δεν ξέρουμε τι ακριβώς είναι. Επομένως, αυτό που λέτε να ορίσουμε για τις κατηγορίες ε, των τροφίμων είναι και αυτό επικίνδυνο, γιατί κινδυνεύουμε να περιορίσουμε το πεδίο και να παρέσχουμε τη δυνατότητα ενταχθούν νέα προϊόντα σε αυτόν τον κατάλογο χωρίς να έχουμε πραγματικό έλεγχο. Πέρα από εκεί έχουμε και πιο τεχνικά θέματα, όπως ε, το θέμα της παρουσίας των ενοηλικών, του καθορισμού των κατηγοριών. Εδώ ε, για το θέμα των ενοηλικών, πρόκειται για εξολόγηση κινδύνου και όχι μόνο θέμα επισήμανσης. Και πρέπει να κατανοήσουμε ότι η αξιολόγηση και η ποσοτικοποίηση των ενοηλικών είναι ζωτική για τον καθορισμό ενός νεοτροφίμου. γιατί κατά την άποψή μας και ένα πολύ μικρό μέρος του ενοηλικού, αν υπάρχει, θα ορίσει το τρόφιμο ως νεοτρόφιμο. Κάτι άλλο πολύ σημαντικό ήταν ε, το θέμα των σημαντικών ε, αλλαγών στη δομή ε, των τροφίμων που τροποποιούν ε, την ε, θρεπτική αξία και υπάρχουν και ανεπιθύμητες ουσίες. Ποιες είναι αυτές οι ανεπιθύμητες ουσίες, υπάρχει κατάλογος και αυτά τα νέα τρόφιμα δεν θα έπρεπε υποτίθεται να είναι καλύτερα και να μην ε, περιέχουν κανένα τέτοιο χειρότερο στοιχείο. Δηλαδή θέλουμε να βελτιώσουμε, να προστατεύσουμε την υγεία και την ποιότητα των τροφίμων. Πραγματική ερώτηση λοιπόν που θα ήθελα να θέσω και κάπως προκλητικά είναι το εξής. Θέλουμε ουσιαστικά ο κανονισμός εδώ να ευνοήσει την λογική της αγοράς ε, και τους επιχειρηματίες ή θέλουμε ένα κανονισμό, μια νομοθεσία πιο σαφή και πιο περιορισμένη για να προστατεύσουμε τα συμφέροντα και την υγεία των καταναλωτών και των περιβάλλον. Αυτή είναι η άποψή μας, έτσι βλέπουμε τα καυτά θέματα και θέλουμε να υπάρχει μεγαλύτερος προβληματισμός γιατί εμείς ε, ουσιαστικά θα θέλουμε πιο συγκεκριμένη πολιτική για τα τρόφιμα και ε, νομίζω ότι πρέπει να όλα αυτά να δείχνουν και προς την κατεύθυνση μιας εκπαίδευσης στον τομέα των τροφίμων, της διατροφής. Κύριε Μπότσα. E, Ευχαριστώ πολύ. Στόχος είναι να εγγυθούμε την διατροφική ασφάλεια, να προστατεύσουμε την υγεία των καταναλωτών και να υποστηρίξουμε την καινοτομία. Και αυτοί οι στόχοι θα επιτευχθούν αν ορίσουμε το πεδίο εφαρμογής, αν επιταχύνουμε τις διαδικασίες και αν λάβουμε αποφάσεις που θα πρέπει να υιοθετηθούν ισότιμα από όλα τα κράτη-μέλη. Μέχρι τώρα έχουμε δει εγγενείς δυσκολίες ε, γιατί οι αιτούντες αδειών για ε, τα νέα τρόφιμα δεν ξέρουν ε, ποια έγγραφα πρέπει να συνοδεύουν την αίτηση. Έτσι λοιπόν οι οργανισμοί ε, λάμβαναν αυτές τις αιτήσει και τις έστειλαν στους αρμόδιους οργανισμούς ε, για να λάβουν ε, την άποψή τους και κατόπιν δεν υπήρχε δυνατότητα να επικοινωνήσουν οι αρμόδιοι με τους ετούντες. Έτσι λοιπόν έστελναν τις αιτήσει στο Υπουργείο και μετά πάλι πίσω στον ετούντα. Υπήρχε πολύ μεγάλη καθυστέρηση λοιπόν για την έκδοση των αδειών και θα έπρεπε λοιπόν να καθορίζουμε στην νομοθεσία ποια είναι τα απαραίτητα έγγραφα που πρέπει να συνοδεύουν την αίτηση για να κυκλοφορήσουν στην αγορά νέα τρόφιμα, έτσι ώστε να αποφύγουμε περαιτέρω καθυστερήσεις. Επίσης, βάση της αρχής της διαφάνειας, θα ήταν καλό να έχουμε έναν κατάλογο των αιτήσεων λαμβάνοντας φυσικά υπόψη και την προστασία των δεδομένων σύμφωνα με το άρθρο 22. Και καθώς η έγκριση αυτή θα ισχύει σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν πρέπει να έχουμε επικαλύψεις ε, και ούτε να ζητάμε από τους ετούντες να στέλνουν ε, τις αιτήσει τους σε διαφορετικούς οργανισμούς και σε διαφορετικά αντίτυπα. Η κυρία Πέτικα είναι τελευταία. Ευχαριστώ πολύ. Συμφωνώ με τα σχόλια που έχουν ήδη γίνει. Να τονίσω ωστόσο ότι είναι πολύ σημαντικό το θέμα αυτό. Ή θα έχουμε μια καλή νομοθεσία, είτε δεν θα έχουμε. Και αν δεν έχουμε καλή νομοθεσία για την κλωνοποίηση, για την ασφάλεια, για την εισαγωγή των νέων νανοηλικών, δεν θα μπορούμε να επανέλθουμε και να διορθώσουμε την κατάσταση. Γι' αυτό κάνω έκκληση προς όλους. Να είμαστε ιδιαίτερα στεναροί, αλλά και αποδοτικοί. Πρώτα απ' όλα πρέπει να εφαρμόσουμε την ε, αρχή της ε, πρόληψης με πολύ αυστηρό τρόπο. Δεν έχει να εισαγάγουμε κάτι και μετά να μην το εφαρμόσουμε. Πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι τα πρόσθετα είναι ασφαλή. Τα πρόσθετα τροφίμων. Δεν είναι μόνο θέμα είναι θέμα διαδικασιών. Κάτι άλλο. Γιατί ήμουν ε, μέλος της διαπραγματευτικής ομάδας την προηγούμενη φορά. Έχουμε πολύ ισχυρέ πιέσεις να μην υπάρξει καθόλου νομοθεσία για τα κλωνοποιημένα σε αυτή τη φάση. Γιατί η επιστήμη προοδεύει πάρα πολύ. Αν περιμένουν δύο-τρία χρόνια, τα κλανοποιημένα ήδη υπάρχουν. Και δεν θα μπορούμε να τα απογορεύσουμε. Γιατί ήδη θα έχουν μπει στην αγορά. Πολύ σημαντικό λοιπόν να συμπεριληφθεί ο τομέας των γενετικά τροποποιημένων σε αυτό τον κανονισμό και να συμπεριλαμβάνονται τρεις γενιές των απογόνων του κλωνοποιημένου και επίσης πρέπει να υπάρχει ίχνη λασιμότητα, ό,τι και να πείτε. Αν μπορεί να γίνει ή όχι. Και το έλεξα, ναι μπορεί να γίνει. Το έλεξα από διάφορους διεθνείς οργανισμούς να έχουμε ε, μία, ε, κωδικούς, να έχουμε μία διαδικασία κωδικών για, τα, για το γονιδίωμα. Αυτά είναι προϋποθέσεις για να έχουμε καλό κανονισμό. Όπως είπαμε και κατά την προηγούμενη θητεία, εάν το Συμβούλιο και η Επιτροπή δεν συμφωνούν, τότε καλύτερα να μην έχουμε κανονισμό. Παρά να καταλήξουμε σε έναν απαράδεκτο κανονισμό που δεν θα μπορούμε να το διορθώσουμε μετά όταν θα έχει αρχίσει να εφαρμόζεται. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. και έχουν υποβληθεί κάποιες ερωτήσεις από συναδέλφους στην Επιτροπή οπότε να ζητήσω από τον κύριο που λέει από την Επιτροπή να απαντήσει στις ερωτήσεις που υπέβαλαν οι συνάδελφοι. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Όντως. Και μας μας εντυπωσίασε ο μεγάλος αριθμός ε, τροπολογιών που υποβλήθηκαν και εδώ και στην Άγκρη να επιχειρήσω να απαντήσω σε ορισμένα θέματα. Πρώτον, η επανεισαγωγή κατηγοριών. Βεβαίως, στην αρχική πρόταση της Επιτροπής δεν ε, περιλαμβάναμε αυτά που υπήρχαν στα προηγούμενα κείμενα. Αλλά αντιλαμβανόμεθα ότι έτσι γίνεται πιο σαφής η συζήτηση και οι προτάσεις και των ετούντων μας πείθουν να μην είμαστε κατά της επανεισαγωγής κατηγοριών για αυτά τα νέα τρόφιμα. Δεύτερον, πολύ το αναφέρατε, κλωνοποίηση. Ξέρετε ότι η Επιτροπή έκανε μια παράλληλη πρόταση για τη συζήτηση για τα κλωνοποιημένα. Είναι δύσκολη, πολύ. Σε αυτό το κείμενο για τα νέα τρόφιμα δεν, αναφερόμε, δεν αναφερόμασταν ε, στους ε, γάμα τάφ αλλά είναι σαφές ότι τουλάχιστον για το κρέας και το γάλα που προέρχονται από κλωνοποιημένα πρέπει να διατηρηθούν οι αναφορές. Γι' αυτό και περιμένοντας το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο να εγκρίνουν αυτό το νέο κείμενο για τα κλωνοποιημένα κάνουμε αυτές τις αναφορές. Είμαστε υπέρ της τροπολογίας 92. Να επανέλθουμε στην ε, προηγούμενη άποψη ότι τα τρόφιμα που προέρχονται από κλωνοποιημένα ζώα πρέπει να θεωρούνται νέα τρόφιμα και να υποβάλλονται σε όλες τις διαδικασίες επιστημονικής εξέτασης και έγκρισης. Για τα νάνο υλικά. Ξέρετε ότι υπάρχει ορισμός. Στο κείμενο ενημέρωση καταναλωτών για τα τρόφιμα. Είναι το κείμενο 69 του 2011. Και με κατεξοδότηση πράξη είχαμε ζητήσει τροποποίηση του ορισμού. Το προηγούμενο κοινοβούλιο απέριψε αυτή την πρότασή μας και πολύ σύντομα θα σας υποβάλουμε ένα νέο κείμενο για αυτήν την κατεξοδότηση πράξη που θα περιλαμβάνει αυτά που ζήτησε το Κοινοβούλιο. Δηλαδή ότι τα παλιά πρόσθετα, αυτά δηλαδή που είναι στην αγορά εδώ και καιρό αλλά περιέχουν λόγω της διαδικασίας ε, κατασκευής τους νανοελικά να περιληφθούν σε αυτή την πρόταση για την ε, ταυτοποίηση και σήμανση. Αυτό που δεν επιθυμούμε για λόγους νομικής σαφήνειας είναι να μην έχουμε δύο διαφορετικούς ορισμούς σε δύο κείμενα. Ένα στη σήμανση και ένα για τα νέα τρόφιμα. Και με δυνατότητα τροποποίησης με κατεξοδότηση πράξη και για τα δύο κείμενα, γιατί φοβόμαστε πολύ, ότι αν υπάρχουν δύο κείμενα, δύο δυνατότητες τροποποίησης, με συμμετοχή εμπειρογνωμών από τα κράτη-μέλη και το Κοινοβούλιο, φοβόμαστε λοιπόν ότι τελικά θα αποκλίνουν οι ορισμοί. Θα θέλαμε να υπάρχει ένας μόνο ορισμός και κυρίως το κείμενο για τη σήμανση που να λαμβάνει υπόψη το θέμα της αποτίμησης της ε, ασφάλειας τροφίμων, όπως ισχύει για τα νέα τρόφιμα. Προφανώς ε, τίθεται επίσης το θέμα του κατοφλίου, αν θα είναι 50% ή 10%. Ο κύριο Πότς έχει δίκιο. Σήμερα είναι αδύνατο να ανοιχνεύσουμε 10% νανοηλικών σε ένα συστατικό στο μέλλον. Σίγουρα θα έχουμε αυτή τη δυνατότητα, αλλά σήμερα ακόμη και αν είναι 50% είναι δύσκολο να ανοιχνευθεί. Αλλά βάλαμε ένα άρθρο που λέει ότι όσο θα προχωράει η επιστημονική γνώση, αυτό το επίπεδο του 50% θα μειωθεί. Στο 40, 30, 20, 10. Νομίζω ότι όλοι το επιθυμούμε τουλάχιστον οι παρόντε εδώ, Κοινοβούλιο, Συμβούλιο, Επιτροπή δηλαδή, όλοι θέλουμε να έχουμε ένα πολύ χαμηλό κατώτατο όριο, αλλά σήμερα δεν είναι εφικτό. Δεν μπορούμε να ελέγξουμε. Ούτε στα εργοστάσια που παράγουν αυτά τα προϊόντα, ούτε όταν εισάγονται από τρίτες χώρες. Είναι αδύνατο, επαναλαμβάνω, να ελέγξουμε ένα 10% αυτά για τα νάνο υλικά θέλουμε να υπάρχει λογική και για τη σήμανση επί των προϊόντων για ενημέρωση του καταναλωτή και για αποτίμηση του επίπεδου ασφάλειας τροφίμων για αυτά τα νέα τρόφιμα και όχι μόνο για αυτά αλλά και αυτά που υπήρχαν πριν το 97 άρα θέλουμε να υπάρχει ένας μόνο ορισμός στο κείμενο για τη σήμανση για το οποίο βεβαίως θα έχετε δυνατότητα να εκφραστείτε. Άλλο θέμα που εφήγει η αναφορά στην αρχή της πρόληψης ή στην αρχή της, ε, του αντικτύπου στο περιβάλλον των νέων τροφίμων. Έχουμε μια ολόκληρη συστοιχεία κειμένων για τους τομείς αυτούς, είτε είναι θέμα προστασίας του περιβάλλοντος, είτε είναι θέμα χρήσης, εφαρμογής της αρχής της πρόληψης και βεβαίως το κείμενο αυτό ισχύει πλήρως και για τα νέα τρόφιμα. Αποτίμησή τους και όταν η ΕΦΣΑ, η αρχή για την ασφάλεια των τροφίμων, θα μελετήσει το επίπεδο ασφαλείας για τα νέα τρόφιμα, εάν δεν έχει όλη την ε, επιστημονική τεκμηρίωση για να αποδείξει ότι είναι αυλαβή, τότε η αρχή της ε, πρόληψης που ισχύει γενικά για τα τρόφιμα θα ισχύσει και εδώ. Αν υπάρχουν αμφιβολίες για το κατά πόσον είναι αυλαβή, αυτή λοιπόν η αρχή της ε, πρόληψης θα έχει ως επίπτωση τη μη χορήγηση έγκρισης κυκλοφορίας. διαφάνεια και αυλαβής χαρακτήρας. Η πρόταση που έχετε υποβάλει είναι να υπάρχει δυνατότητα ενημέρωσης των κρατών μελών και των ετούντων αναλυτικά για να καταλάβουν τι είναι ένα νέο τρόφιμο. Συμφωνούμε. Βεβαίως, θα υπάρξουν κατευθυντήριες γραμμές που θα εκπονηθούν σε συνεργασία με την ΕΦΣΑ για να μπορούν οι επιχειρήσεις και ιδιαίτερα οι μικρομεσαίες να ερμηνεύσουν τα κείμενα. Είναι σαφές ότι αυτές οι κατευθυντήριες γραμμές δεν τροποποιούν την νομοθεσία, απλώς την εξηγούν. Πολλοί επίσης ε, αναφέρθηκαν στο θέμα αυτό κατεξοδότηση ή εκτελεστικές πράξεις. Εδώ υπάρχει διαφωνία μεταξύ Κοινοβουλίου και Συμβουλίου. Οι, οι μεν και οι δε πράξεις δεν έχουν στόχο δεν έχουν δυνατότητα να τροποποιούν το βασικό κείμενο. Όλοι οι νομομαθείς και των δικών σας και των δικών μας νομικών υπηρεσιών επαγρυπνούν ιδιαίτερα από αυτού και δεν είναι δυνατόν με τις πράξεις αυτές να τροποποιηθεί το κείμενο στο οποίο αναφέρονται. Δεν είναι δυνατόν. Και δεν το κάνουμε. Αντίθετα θεωρούμε ότι πρέπει να έχουμε μια κάποια ευελιξία ιδιαίτερα για την εκπόνηση των καταλόγων νέων τροφίμων, για την ε, πορεία μετάβασης από το προηγούμενο στο νέο κείμενο που θα εγκριθεί και γι' αυτό έχουμε ανάγκη την ευελιξία που μας δίνουν οι εκτελεστικές πράξεις για να μην παραλύσει το σύστημα. Η κυρία Πόλσεν το είπε. Πρέπει να απλοποιήσουμε τις διαδικασίες για να επιτρέψουμε στις επιχειρήσεις να παίξουν πλήρως το ρόλο τους ε, καινοτομίας, να μην τις εμποδίζουμε με υπερβολική γραφειοκρατία. Αυτό είναι το μήνυμα και του καινούργιου Προέδρου μας, του κυρίου Γιούνκερ. Γιατί θέλουμε να προωθήσουμε την καινοτομία. Είναι πολύ βασικό, ιδιαίτερα στον τομέα των τροφίμων, όπου συχνά Υπάρχουν φόβοι, αμφιβολίες, άγχη ε, για τα τρόφιμα, κάτι που δεν ισχύει για άλλους ε, βιομηχανικούς κλάδους ή για τα φάρμακα. Και μέσω της επιστημονικής εκτίμησης του ΕΦΣΑ νομίζω ότι έχουμε όλες τις εγγύησεις που δεν θα επιτρέψουν την εισαγωγή μη ασφαλών τροφίμων στην αγορά. Αλλά αυτό για το οποίο μας επικρίνουν οι επιχειρήσεις, ο κλάδος, είναι ότι η διαδικασία εισαγωγής στην αγορά νέων τροφίμων πρέπει να είναι σχετικά ταχεία. Αυτά θέλαμε να τονίσουμε και καταλήγοντας τονίζω ότι φυσικά ε, προσβλέπουμε στη συνεργασία με τον κύριο Νίκολσον και τους Κιώδης για να καταλήξουμε από κοινού και με το Συμβούλιο σε ένα κείμενο για τα νέα τρόφιμα που να είναι θαυμάσιο και να εγκριθεί όσο το δυνατόν ταχύτερα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Και τώρα ο κύριος Νίκολσον για να ολοκληρώσουμε. Ευχαριστώ Πρόεδρε και ευχαριστώ όλους ε, για τα σχόλιά τους. Νομίζω ότι ήταν ε, πάρα πολύ χρήσιμα. Η συζήτηση ήταν πολύ καλή και επέφερε σαφήνεια. Φυσικά υπάρχουν ακρεμή ζητήματα. Υπάρχουν και κάποιες μεγάλες διαφωνίες και αν μπορούμε να ξεπεράσουμε αυτά τα εμπόδια θα το δούμε, αλλά σίγουρα θα εργαστούμε σκληρά για να το πετύχουμε τις επόμενες εβδομάδες. Σας ευχαριστώ όλους και ζητώ συγγνώμη γιατί πρέπει να πάω στην Επιτροπή Γεωργίας γιατί έχω και εκεί μια έκθεση που αναμένει. Ευχαριστώ. Μάλιστα, πριν ολοκληρώσουμε τη συζήτηση, πρέπει να υπενθυμίσουμε ότι η ψηφοφορία θα λάβει χώρα σε μια έκτατη συνεδρίαση στο Στρασβούργο στις 24 Νοεμβρίου για την έκθεση για τα νέα τρόφιμα και τώρα μπορούμε να πάμε στο επόμενο θέμα που είναι η Σύμβαση για το Διεθνές Εμπόριο των Ειδών Άγριας κλωρίδες και Πανίδας που απειλούνται με εξαφάνιση, τη Σύμβαση ΣΥΤΕΣ. Και θα δώσω αμέσως το λόγο στην εισηγήτρια μάλλον πρώτα στην Κομισιόν. Καταρχήν το λόγο στην Κομισιόν επομένως και κατόπιν θα ακούσουμε την εισηγήτρια. Ευχαριστώ Πρόεδρε, καλημέρα σε όλους. Ευχαριστώ την κυρία Αγιούσο για την έκθεσή της και που πρότεινε να συνενέσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στην προσχώρηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Σύμβαση ΣΥΤΕΣ. Όπως ε, ξέρετε, θα ήθελα να πω δύο λόγια για τις συζήτες. Ε, η σύμβαση αυτή γράφτηκε το 1973, μόνο τότε κράτη μπορούσε να είναι μέρη της σύμβασης. Από τότε υπήρξε μετακίνηση και πολλές περιβαλλοντικές συμβάσεις που γνωρίζουμε προβλέπουν δυνατότητα και για τη συμπεριλήψη περιφερειακών οργανώσεων, όπως είναι και η Ευρωπαϊκή Ένωση, να καταστούν μέλη. Αυτό απέτησε μια τροποποίηση της ε, σύμβασης ε, ΣΕΤΕΣ ε, που τέθηκε σε ισχύ το Νοέμβριο 2013 και έτσι κάναμε την αντίστοιχη πρόταση να προσχωρήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση τώρα στην σύμβαση αυτή. Το μόνο που θέλω να πω είναι ότι η ΣΥΤΕΣ είναι μια σύμβαση που αφορά το ε, τα εμπορίου, περιβαλλοντικά ε, θέματα, στα οποία η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ισχυρές αρμοδιότητες και να καταστήσουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση μέρος στη σύμβαση. Ουσιαστικά βοηθάστε να διορθώσουμε μια ανομαλία και φυσικά η προσχώρηση θα βελτιώσει την παρουσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης εντός της δουλειάς σύμβασης, τη λογοδοσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, για θέματα παγκοσμίου εμπορίου και επίσης ε, θα τη βοηθήσει να συμμετάσχει πλήρως στο έργο όλων των ε, φορέων της σύμβασης. Και να πω και κάτι για το ευρύτερο πλαίσιο και να πω ότι αυτή η προσχώρηση γίνεται σε μια πολύ σημαντική στιγμή για την ε, ΣΥΤΕΣ, γιατί ε, δεσμεύεται περισσότερο στο να ρυθμίσει το διεθνέ εμπόριο ε, στα είδη που απειλούνται με εξαφάνιση και σε ό,τι αφορά και την ξυλία και να καταπολεμήσει την παράνομη εμπορία. Επίσης έχει οθετήσει ισχυρά μέτρα πρόσφατα η Σύμβαση για κάποια μέτρα που αφορούν την εμπορία ξυλία, ενό είδου ξυλία και την πορεία ελεφαντόδοντου. Επομένως, ε, η προσχώρηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Σύμβαση θα είναι ένα ορατό βήμα για την Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι ένα βήμα που πρέπει να το κάνουμε για να αυξήσουμε ε, το ρόλο μας στην καταπολέμηση του διεθνούς εμπορίου των ειδών αγρίας χλωρίδας και πανίδας. Θα δώσουμε τώρα το λόγο στην εισηγήτρια, την κυρία Πιλάρ Αγιούσο. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ και την Κομισιόν για την εξήγησή της. Πολύ καλά μας τα εξήγησε, περί την ως πρόκειται, να εγκρίνουμε μια τροπολογία της στην Ευρωπαϊκή Ένωση να ε, γίνει από παρατηρητής ε, μέλος ε, της ΕΣΥΤΕΣ. Το μόνο πρόβλημα που υπήρχε με αυτό και όλοι συμφωνούμε γιατί και τα κράτη-μέλη θα συνεχίσουν να έχουν το καθεστώς που έχουμε μέχρι σήμερα είναι ότι η πρόταση της Κομισιόν για αυτή την ε, τροπολογία μας προτείνει αυτό να γίνει με την ε, νομική βάση δύο άρθρων, το 192 που αφορά το περιβάλλον ε, και το 207 που αφορά την κοινή εμπορική πολιτική. Εγώ πιστεύω ότι πρόκειται για μια ορθή πρόταση, καθώς ένα από τα μεγάλα προβλήματα που έχουν τα ίδια που απειλούνται με εξαφάνιση είναι η παράνομη εμπορία που γίνεται. Επομένως, ε, το να έχουμε υπόψη και το άρθρο 207 ως νομική βάση για την εμπορική πολιτική είναι θεμελιώδες. Παρ' όλα αυτά, η πρόταση του Συμβουλίου είναι μόνο να υπάρχει νομική βάση το άρθρο που αφορά το περιβάλλον. Όμως η θέση μου και η θέση της πολιτικής μου ομάδας είναι ότι πρέπει να έχουμε διπλή νομική βάση, έτσι όπως προτείνει και η Κομισιόν. Δεν ε, χρειάζονται τροπολογίες εδώ, απλώς θα ψηφίσουμε ναι ή όχι. Και αυτή είναι η πρότασή μου και η πρόταση της ομάδας μου. Ευχαριστώ πολύ για την Ομάδα Δημοκρατών και Σοσιαλιστών. Κυρία Μπριάνο. Ευχαριστώ. Και εγώ θα είμαι πολύ σύντομη. Ευχαριστώ την εισηγητρία για τη δουλειά της και ευχαριστώ και την Κομισιόν. Εμείς συμφωνούμε απόλυτα. Επιτέλους η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να προσχωρήσει σε αυτήν την πολύ σημαντική σύμβαση. Θέλουμε λοιπόν να υπερψηφίσουμε για την προσχώρηση και συμφωνούμε και με την άποψη της νομικής Επιτροπή νομικέ υπηρεσίε, δηλαδή να έχουμε διπλή νομική βάση και για το περιβάλλον και για την εμπορική πολιτική. Θέλουμε λοιπόν αυτή η σύμβαση να υπερψηφιστεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ για τους Ευρωπαίου Συντηρητικού Μετεχνιστές. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ επίση και εξ ονόματο ε, της ε, πολιτικής μου ομάδος και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την εισηγήτρια. Η συμφωνία για το διεθνές εμπόριο απειλουμένων ειδών, οι σάιτες, έχει ηλικία πλέον των 40 ετών και σήμερα είναι πλέον απαραίτητο από ποτέ να προστατευτούν ορισμένα είδη. Συζητούμε εδώ την προσχώρηση Ευρωπαϊκής Ενώσεως στην Συμφωνία. Μέχρι πρόσφατα η Ευρωπαϊκή Ένωση είχε το καθεστώς του παρατηρητού Είναι σημαντικό το πλαίσιο ωστόσο και αυτό το πλαίσιο να ε, εξεταστεί μέσα σε μια ιστορική πορεία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση εφαρμόζει την σύμβαση ΣΑΙΤΕΣ με τον κανονισμό 338-97 που έχει όμως μπλοκαριστεί μέσα στον κικαιώνα των εκτελεστικών και κατεξουσιοδότηση πράξεων και ανάμεσα στο Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο ελπίζω ότι οι συζητήσεις για την αναθεώρηση θα μπορέσουν να προχωρήσουν του κανονισμού αυτού. Τώρα, όπως και η κυρία Ιούσο, εμείς υποστηρίζουμε την προσχώρηση Ευρωπαϊκής Ενώσεως στην Σύμβαση ΣΑΙΤΕΣ που θα προσφέρει ασφάλεια δικαίου για τον ρόλο της Ευρωπαϊκής Ενώσεως αλλά και για την ισχύ της ΣΑΙΤΕΣ. Δεν υπάρχει διαφορά από την προσχώρηση σε άλλες διεθνείς συμβάσεις όπως πρωτόκολλο της ε, Καθαγέννης και άλλα που έχουν και αυτές αντικείμενο περιβαλλοντικά θέματα. Υπάρχουν ορισμένα θέματα που θεωρούνται εθνικά θέματα και άλλα, αρμοδιότητες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό όμως δεν τροποποιεί την σχέση μεταξύ των αρμοδιοτήτων αυτών, ούτε τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να αναπτυχθεί η δικαιοδοσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και αυτά τα λέει η συγγήτρια στο επεξηγηματικό μνημόνιο. Σημαντική είναι και η νομική βάση. Η νομική υπηρεσία της Ευρωπαϊκής, ε, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μάλλον συμφωνεί με τη νομική υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τη διπλή βάση για το διεθνές εμπόριο και για το ε, διπλασιό του περιβάλλοντος που εμάς μας βρίσκει σύμφωνος και εν πάση περιπτώσει η συζήτηση αυτή δεν πρόκειται να μας αποτρέψει από το να εγκρίνουμε την προσχώρηση. Ευχαριστώ η ομάδα των φιλελευθέρων τώρα, ο κύριος Γκέρ Μπράντι. Ευχαριστώ και εγώ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ με τη σειρά μου και την ε, εισηγήτρια κυρία Γιούσο καθώ και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που κατέθεσε την πρόταση. Είναι ένα βήμα το οποίο είναι απόλυτα απαραίτητο για να μιλήσουμε μέσα στην ΣΥΤΕΣ με μια φωνή ω Ευρωπαϊκή Ένωση. Κατέστην Μάρτης εγώ ο ίδιο, όταν ήμουν παρόν σε συνδιάσκεψη των μερών το 2010 ότι οι χώρες μέλη της Ένωσης διαπραγματεύονταν πιο πολύ μεταξύ τους παρά με τον υπόλοιπο κόσμο. Και για το λόγο αυτό δεν μπορούσαμε να ασκήσουμε σχεδόν καμιά επιρροή στην ε, σύμβαση ΣΑΙΤΕΣ. Ήταν πραγματικά πολύ απογοητευτικό. Προσπαθήσαμε να περιλάβουμε θαλάσσια είδη, στην συνδιάσκεψη των μερών της ΣΑΙΤΕΣ το 2010, αλλά δεν τα καταφέραμε διότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μιλούσε με μια φωνή και δεν είχε τη σωστή στόχευση. Ένα βήμα λοιπόν που είναι πραγματικά απαραίτητο. Με μια επιφύλαξη. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα μπορεί να μιλεί και να ψηφίζει στο όνομα των 28 χώρων μελών εφόσον φύγεται το ευρωπαϊκό κοινοτικό κεκτημένο. Και αν όχι, τότε ψηφίζουν ξεχωριστά οι χώρες μέλη και μιλούν χωριστά. Βέβαια γι' αυτό δεν μπορούμε να κάνουμε πολλά πράγματα. Νομίζω όμως ότι ήδη με την παρουσία του ο αρμόδιος επίτροπος στη συνδιάσκεψη των μερών και έχοντας μια ισχυρή θέση των χωρών μελών θα μπορεί να μιλήσει παρόλα αυτά όσο είναι δυνατόν αυτό με μια φωνή έτσι ώστε να μην κατακαιρματίζονται οι προσπάθειες των χωρών μελών, στερώντας τους τη δυνατότητα να ασκήσουν οποιαδήποτε επιρροή. Γι' αυτό λοιπόν θα παρακαλέσω και ο αρμόδιος, αρμόδιος Πέτρος Βέλα να παίξει τον ρόλο αυτό και γι' αυτό απευθύνω σχετική έκκληση. Ομάδα FDD Σαφρόντε. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Δεν έχω πολλά να προσθέσω, απλώς να πω ότι και η δική μας ομάδα βλέπει θετικά την ένταξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην σύμβαση της ως σταθερό μέλος. Η Επιτροπή της ούσικτον είναι μία από τις πλέον παλιές σε σχέση με την προστασία του περιβάλλοντος, η έχει συμπληρώσει 30 χρόνια λειτουργίας και είναι και μία από τις πιο αποτελεσματικές και πρόκειται για μία από τις ε, επιτροπές με τα περισσότερα μέλη γιατί 100 από 108 κράτη ε, είναι μέλη και τα εφαρμόζουν, εφαρμόζουν τη σύμβαση στην ομοθεσία τους. Έτσι λοιπόν είναι σημαντικό βήμα για την Ευρωπαϊκή Ένωση να μην είναι πλέον ένας παθητικός παρατηρητή, αλλά να μπορεί να κάνει και τη φωνή τη να ακουστεί ενιαία εντός της σύμβαση αυτή και με αυτόν τον τρόπο να μπορέσει να προωθήσει και πιο αποτελεσματικά την ίδια την πολιτική της ε, για την προστασία του περιβάλλοντος και της πανίδα και τη κλωρίδας. Σα ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Νομίζω ότι για την Κομισιόν δεν φαντάζομαι θέλει να αντιδράσει. Συμφωνείτε? Ίσως σύντομα. Να ευχαριστήσω όσους μίλησαν για τη στήριξη που μας δώσαν. Ο κύριος Γκεμπράντι αναφέρθηκε στο ε, άτυχο επεισόδιο της διαφοράς απόψεων για τον ερυθρό τόνο και σας διαβεβαιώ ότι θα κάνουμε ό,τι μπορούμε και θα ενημερώσουμε και τον Επίτροπο για τα αιτήματα και τις επιθυμίες που εκφράσατε. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Λοιπόν, χρονοδιάγραμμα. Ψηφοφορία στην Επιτροπή μας σήμερα το απόγευμα και στην Ολομέλεια το Δεκέμβριο. Οπότε μπορούμε να κλείσουμε την εξέταση αυτού του θέματος και να περάσουμε στο επόμενο. Ανταλλαγή απόψεων με τον κύριο Φραντς Φίσλερ που είναι πρόεδρος της Διευθύνουσας Επιτροπής του Επιστημονικού Προγράμματος της Ένωσης για την Expo 2015. Η έκθεση, αυτή η Expo αυτή είναι μια παγκόσμια έκθεση που θα λάβει χώρα 1η Μαΐου με 31 Οκτωβρίου 2015 στο Μιλάνο. Θα συμμετάσχουν πάνω από 160 συμμετέχοντες ε, μεταξύ των οποίων η Ένωση και τα κράτη-μέλη της. Περιμένουμε ότι πολλοί άλλοι φορείς θα συμμετάσχουν και αναμένονται πάνω από 20 εκατομμύρια επισκέπτες. Το θέμα είναι ε, πώς θα δρέψουμε τον πλανήτη και ενέργεια για τη ζωή. Και γι' αυτό καλέσαμε εδώ τον πρόεδρο της Διευθύνουσας Επιτροπής για να μας παρουσιάσει τον τρόπο με τον οποίο σκέφτεται να παρουσιάσει αυτό το σημαντικό θέμα και ελπίζουμε να συμμετάσχει επιτυχώς η Ευρωπαϊκή Ένωση σε αυτή τη σημαντική έκθεση. Και να δώσω λοιπόν ε, καταρχάς το λόγο στον κύριο Φίσλερ για την παρουσίασή του. Ευχαριστώ πολύ πρόεδρε. Καλημέρα σας. Ε, κύριοι βουλευτές, κυρίες και κύριοι, σε ακριβώς 177 μέρες θα ανοίξει η Expo Μιλάνο 2015. Θα προσφέρει στην Ευρώπη μια μοναδική ευκαιρία να εστιάσει σε μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις για το κοινό μας μέλλον. Πώς να διασφαλίσουμε ασφαλή, επαρκή και θρεπτική τροφή για όλη την ανθρωπότητα με βιώσιμο τρόπο. Σας ομιλώ ως Πρόεδρος της Διευθύνουσης Επιτροπής, όπως είπε και ο Πρόεδρος, που λειτουργεί ήδη από το Μάρτιο, μαζί με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, συμμετέχουν 11 υψηλού επίπεδο από την Ευρώπη και περαιτέρω και ευρύτερα για να μας δώσουν ε, βοήθεια στην ε, εκπόνηση του επιστημονικού προγράμματος της Ένωσης για αυτήν την Expo 2015. Στόχος μας είναι να συμβάλλουμε στην κληρονομιά της Expo 2015 μέσω ανάπτυξης ενός ε, διαλόγου για την πολιτική και για την ανάπτυξη ενός επιστημονικού προγράμματος για την παγκόσμια επιστηστική ασφάλεια. Θα συμμετάσχουν πολλές οργανώσεις, 147 χώρες, καθώς και οι οργανώσεις του, των Ηνωμένων που έχουν βάσει τη Ρώμη και είναι προς το συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης να αξιοποιήσουμε αυτό το βήμα για να ε, εδρεώσουμε το ρόλο μας ως βασικός ενεχόμενος στη συζήτηση για την επιστηστική ασφάλεια στον πλανήτη μας. Το θέμα της ΕΞΠΟ Πώ θα θρέψουμε τον πλανήτη, η ενέργεια για τη ζωή είναι στο σταυροδρόμι διαφόρων ενωσιακών πολιτικών από την γεωργία στην ανάπτυξη, από την ασφάλεια των τροφίμων στο περιβάλλον, από τη βιομηχανία στην έρευνα και την καινοτομία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να δράξει αυτή τη μοναδική ευκαιρία και να κάνει μια μόνιμη συμβολή στην παγκόσμια συζήτηση για την επιστημιστική ασφάλεια και βιωσιμότητα. Γι' αυτό έχει θεμελιώδη σημασία όχι απλώς να καταδείξουμε τον εξαιρετικό χαρακτήρα το, του τροφιμικού τομέα της Ευρώπης στο Μιλάνο και να καταδείξουμε την ηγετική θέση μας ε, στην έρευνα για την επιστηστική ασφάλεια, αλλά να συνεργαστούμε για να υπάρξει καρποφόρα συνεργασία με όλους τους φορείς και να καλέσουμε τη διεθνή επιστημονική κοινότητα να συμμετάσχει πλήρως σε αυτό το διάλογο. Ένα σημείο έγινε σαφές από την αρχή της συμμετοχής της Ένωσης, η έρευνα και η καινοτομία είναι κεντρικές για να αντιμετωπίσουμε τις πιέσεις στο παγκόσμιο σύστημα τροφίμων και για να μπορέσουμε να θρέψουμε ένα αυξανόμενο πληθυσμό που απαιτεί όλο και περισσότερες ζωικές πρωτεΐνες χωρίς να εξαντλήσουμε τους φυσικούς μας πόρους στις ερχόμενες δεκαετίες. Πρέπει επίσης να αντιμετωπίσουμε τις ελλείψεις που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στη γεωργική παραγωγή. Ωστόσο, οι περιορισμοί και λόγω της κλιματικής αλλαγής ε, έλλειψης ε, υδάτων και, ε, η χρήση, και της χρήσης εδαφών για μη γεωργικούς σκοπούς θέτουν προβλήματα. Χρειαζόμαστε μια βάση καλής γνώσης και καινοτομία που θα μας επιτρέψουν να αξιοποιήσουμε το δυναμικό για να έχουμε υψηλότερες οδιές, περισσότερη ε, αντοχή και πιο αποτελεσματική χρήση της γης. Και ο ρόλος λοιπόν της ε, Επιστημονικής Επιτροπής είναι να διασφαλίσει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα παίξει πολύ ενεργό ρόλο στην Expo 2015 ούτω ώστε να γίνουν γνωστές οι ιδέες μας να περάσουν και να συμβάλλουμε στη διεθνή συζήτηση. Τους τελευταίους μήνες η Διευθύνουσα Επιτροπή έχει αναπτύξει, ε, έχει εκπονήσει ένα έγγραφο για συζήτηση που περιλαμβάνει τις μελλοντικές προτεραιότητες για την έρευνα, την ανάπτυξη και την καινοτομία στον τομέα των τροφίμων. Το έγγραφο αυτό ιδιαίτερα προσπαθεί να εντοπίσει τους τομείς όπου η ευρωπαϊκή έρευνα μπορεί να προσθέσει τη μεγαλύτερη προστιθέμενη αξία. Θα είναι η βάση για τη συζήτηση με τους εμπλεκόμενους φορείς και το κοινό. Κατά την Expo 2015 θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να ληφθούν υπόψη όλες οι πλευρές της επιστημική ασφάλειας μέσω ελκυστικών εκδηλώσεων και θα υπάρξει πολύ περιθώριο για συζήτηση, διαβούλευση και ανταλλαγή εμπειρίας. Με αυτό τον τρόπο θα συμβάλλουμε στην κληρονομιά της Ένωσης μετά την Expo 2015. Επιτρέψτε μου να πω κάπως περισσότερα για τις συστάσεις μας για να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις της ε, παγκόσμιας ε, ασφάλειας τροφίμων, η Επιτροπή μας θεωρεί ότι πρέπει να υπάρξει περισσότερη γνώση στους επόμενους 7 τομείς. Πρώτον, βελτίωση της δημόσιας υγείας μέσω της διατροφής. Πώς μπορούμε να έχουμε υγιεινή και βιώσιμη διατροφή. Δεύτερον, μείωση των απορριμμάτων. Πώς θα έχουμε πιο αποτελεσματική τροφική αλυσίδα πώς θα αυξήσουμε την ε, ποιότητα και την ασφάλεια των τροφίμων, διαχείριση των τροφίμων σε μια όλο και πιο παγκοσμιοποιημένη ε, αγορά τροφίμων, ισότητα στο σύστημα τροφίμων, διαχείριση των εδαφών για όλα τα οικοσυστήματα και για βιώσιμη ανάπτυξη της υπαίθρου και τελευταίο, αύξηση της απόδοσης της γεωργίας, της βιωσιμότητας, δηλαδή θέλουμε μια βιώσιμη μεγαλύτερη παραγωγή. Πολλά από τα θέματα αυτά ε, εμφύτως αφορούν διάφορους επιστημονικούς τομείς. Επίσης, ε, πολλά από αυτά έχουν ε, βαθιές ρίζες στον πολιτισμό των διαφόρων λαών. Η Ένωση μας μπορεί να παίξει έναν κύριο ρόλο για να αντιμετωπίσουμε αυτά τα θέματα που αφορούν διάφορους τομείς μέσω της συμμετοχής της έρευνας, δείχνοντας τον ηγετικό της ρόλο ε, εφαρμόζοντας την έρευνα και την καινοτομία και ενθαρρύνοντας ε, πολυτομιακές προσεγγίσεις. Αλλά μπορεί να μην αρκέσουν αυτά για να βρούμε μια λύση σε αυτό το δύσκολο σύστημα εξισώσεων. Πρέπει να ασχοληθούμε και με την επίπτωση των επιλογών που κάνει ο κάθε πολίτης ε, στην ε, ασφάλεια τροφίμων. Γι' αυτό έχει θεμελιώδη σημασία να βρωθήσουμε μια καλύτερη κατανόηση του συστήματος τροφίμων και να υπάρχει σεβασμός για τα τρόφιμα μέσω της εκπαίδευσης και της επικοινωνίας για να καταλάβουν οι πολίτες καλύτερα τον σφαιρικό αντίκτυπο των δικών τους ατομικών επιλογών και να αλλάξουν λοιπόν τις συνήθειές τους. Κυρίες και κύριοι, το να θρέψουμε τον πλανήτη είναι ένα τεράστιο και περίπλοκο θέμα. Όπως είδαμε πρέπει να το μελετήσουμε και να κατανοήσουμε καλύτερα τις επιπτώσεις και να τις προλάβουμε. Εμείς ως Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να αξιοποιήσουμε πληρέστατα τους έξι μήνες που θα έχουμε κατά τη διάρκεια της Expo 2015 όταν η προσοχή του πλανήτη θα έχει στραφεί σε μας ούτω ώστε να επιτύχουμε αξιοσημείωτα και απτά αποτελέσματα στη διεθνή συνεργασία για να συμβάλλουμε στην πλανητική ασφάλεια των τροφίμων. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ για την ε, εναρκτήρια ομιλία σας και ας αρχίσουμε τώρα με τις ερωτήσεις και σχόλια από τους συναδέλφους μας και ας αρχίσουμε με την κυρία Πιλάρα Γιούσο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστούμε κύριε Φίσλερ. Ε, χαιρόμαστε πολύ που σας ξαναβλέπουμε εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Χάρηκα πολύ που άκουσα ότι η Expo του Μιλάνου στην έξοδο του Μιλάνου θα υπάρχει και μια αφιέρωση, θα υπάρχει ένα τμήμα που θα αφιερώνεται ε, στην έρευνα και στα γεωπιστητικά θέματα. Χαίρομαι πάρα πολύ που το ακούω γιατί έχω ασχοληθεί με τα θέματα αυτά. Εσείς ε, είστε πρόεδρος της Επιστημονικής Επιτροπής ε, και έχετε δημοσιεύσει ένα έγγραφο που θα ήθελα να το λάβω. Εκεί αναφέρατε 7 σημεία. Πολύ ωραία ακούγονται. Εγώ όμως είδα ότι στο τρίτο σημείο μιλάτε για επιστημιστική ασφάλεια. Μιλάτε για την επιστημιστική ασφάλεια που εννοούμε εδώ στην Ευρώπη. Ε, δηλαδή διατροφική ασφάλεια. Μιλάμε για υγιή και ασφαλή τρόφιμα. Θα ήθελα να μπορείτε να μιλήσετε και για την επιστηστική επάρκεια στο τρίτο κόσμο. Εμείς έχουμε τόσο μεγάλη ε, επάρκεια και δεν σκεφτόμαστε ποτέ ότι λείπουν τρόφιμα στον τρίτο κόσμο. Η έρευνα και η καινοτομία πρέπει να προχωρήσουν στο εξής, το να, υπάρχει, να υπάρχουν επαρκή τρόφιμα για όλο τον κόσμο πέρα από το να είναι ασφαλή τα τρόφιμα, ε, να μειωθούν τα απόβλητα κτλ. Λεχθέντων αυτών νομίζω ότι είναι πολύ, σημαντικό, η, πολύ σημαντική η επιτροπή την οποία προεδρεύεται και εγώ φυσικά εύχομαι όλα αυτά να γίνουν και πράξη. Κάτι άλλο, υπάρχει χρηματοδότηση για να ε, υπάρξουν συγκεκριμένα σχέδια, συγκεκριμένα έργα. Δεν μας είπατε τίποτα. Και ναι, από πού θα προέρθουν οι πόροι. Θα είναι μια ευρωπαϊκή χρηματοδότηση, μια παγκόσμια χρηματοδότηση. Μετά από αυτές τις ε, κύριες γραμμές που μας θέσετε, είναι πολύ σημαντικό να μας πείτε τι υπάρχει από πίσω. Δηλαδή πώς θα υλοποιηθούν όλα αυτά και με ποιους πόρους πώς θα χρηματοδοτηθούν όλα αυτά τα project. Σας ευχαριστώ πολύ. Έχετε πάλι το λόγο κύριε, κύριε πρώην Επίτροπε για να απαντήσετε. Μάλιστα, σας ευχαριστώ για τις ερωτήσεις σας. Πρώτα, το επιστημονικό έγγραφο έχει προχωρήσει πολύ αλλά δεν έχει λάβει ακόμη τελική μορφή. Θα διεξαχθεί και άλλη συνεδρίαση αρχές Δεκεμβρίου της Επιστημονικής Επιτροπής στην οποία συνεδρίαση έχουμε σκοπό να επιφέρουμε βελτιώσεις στο κείμενο και θα σας το διαβάσουμε αμέσως βεβαίως και σε εσά εδώ το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Κανένα πρόβλημα. Για τη δεύτερη σας ερώτηση Εδώ ίσως υπάρχει κάποια δυσκολία σχετικά με τη διατύπωση γιατί στην δική μου μητρική γλώσσα δεν κάνουμε διαφορά. Δεν ε, βλέπουμε διαφορά. Food security και food safety βέβαια δεν είναι το ίδιο πράγμα στα αγγλικά. Αναφέρεται μάλιστα ειδικά στο σημείο Γ ή 3 του εγγράφου ότι food safety, ασφάλεια τροφίμων, είναι μία από τις βασικές αρχές και ε, μία από τις προτεραιότητες Θα ζητήσουμε δε από τις επιστήμονες να ασχοληθούν ειδικά για το πώς θα φτιάξουν ασφαλή τρόφιμα. Το άλλο που έχει σχέση με τη food security είναι πιο πολύ η επάρκεια των τροφίμων. Και αυτό είναι βέβαια και το ε, κυρίαρχο θέμα όταν μιλούμε για παγκόσμια ασφάλεια τροφίμων. Διότι υπάρχει μάλιστα και ορισμός του ΦΑΟ, του ε, Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών, για το τι σημαίνει food security. Και εκεί, εκεί περιλαμβάνονται και όλες οι άλλες αυτές τις πτυχές. Τώρα, για τη χρηματοδότηση και τη χρηματοδότηση της έρευνας, η Ένωση έχει διαθέσει έναν προϋπολογισμό για το Ευρωπαϊκό Περίπτερο στο Μιλάνο. Επιπροσθέτως δε αποφασίστηκε ότι στο περίπτωρο αυτό θα διεξάγονται και πολλές εκδηλώσεις στη διάρκεια των μηνών ε, που θα είναι ανοιχτή η έκθεση, αλλά θα δοθεί και μια συνέχεια, ένα follow-up. Και γι' αυτό το λόγο άλλωστε ιδρύθηκε η ε, Διευθύνουσα Επιτροπή, διότι η ιδέα είναι να μην ολοκληρωθεί το πρόγραμμα με το που θα κλείσει τις πόρτες της τον Οκτώβριο η έκθεση. Το follow-up αυτό θα είναι κυρίως έρευνα, πρόγραμμα ερεύνης. Η χρηματοδότηση ιδέα αυτού του προγράμματος ερεύνης θα βασιστεί στις συνήθεις ε, ε, πηγές χρηματοδοτήσεων για τα ευρωπαϊκά προγράμματα ερεύνης που είναι ιδίως ο ορίζον 2020. Όπως ίσως γνωρίζετε, υπάρχει και ένα καθορισμένο ποσό, earmark δηλαδή, στον προπολογισμό για το ορίζοντα 2020 για την έρευνα στη γεωργία και θα εξαρτηθεί από τους ενδιαφερομένους το από ποιο μέρος του διαθεσίμου προϋπολογισμού θα ε, μπορέσουν να ε, λάβουν ποσά. Σας ευχαριστώ πολύ. Να κάνω κι εγώ μια ερώτηση. Είναι γνωστό ότι οι διεθνείς οργανισμοί μιλούν για μια ανάγκη ε, στα τρόφιμα που μέχρι το 2050 θα αυξηθεί 70%. Χρειαζόμαστε λοιπόν ε, ε, να χρειαστούμε, χρειαζόμαστε να παράγουμε περισσότερο και θα πρέπει να συνδυάσουμε ένα μεγαλύτερο επίπεδο παραγωγής με μια υφορία στην παραγωγή. Και από την άλλη πλευρά επίσης έχουμε την ανάγκη να μειώσουμε όπως ε, αναφέρθηκε και στις κατευθυντήριες γραμμές στα 7 σημεία, να μειώσουμε την κατασπατάληση στα τρόφιμα. Σήμερα μιλάμε για μια διαφορετική κατασπατάληση στις αναπτυγμένες χώρες από τις αναπτυσσόμενες χώρες. Στις αναπτυγμένες χώρες έχουμε κυρίως μια κατασπατάληση που είναι στο τελικό τμήμα ε, της αλυσίδας του κλάδου, δηλαδή πιο κοντά στον καταναλωτή. δεν ε, μπορεί να καταλάβει ποιε είναι ακριβώς οι ανάγκες του και αγοράζει περισσότερο από ό,τι του χρειάζονται και κατόπιν τα πετάει, ενώ στις αναπτυσσόμενες χώρες αντίθετα οι απώλειες κυρίως αφορούν το αρχικό στάδιο του τομέα, δηλαδή έχουμε έλλειψη υποδομών και έλλειψη ενός συστήματος να διατηρούνται νοπατατρόφιμα και αυτό σημαίνει ότι έχουμε απώλειε στην αρχή της διαδικασίας. Ε, πιστεύετε ότι θα εστιάσετε την προσοχή σας ε, στο θέμα της ε, κατασπατάλησης των τροφίμων food waste. Είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα στο Κοινοβούλιο και δώσαμε πολύ μεγάλη προσοχή σε αυτό στην προηγούμενη θητεία, αλλά και σίγουρα και σε αυτή τη θητεία θα είναι ένα θέμα στο οποίο θα εμβαθύνουμε, δεδομένου ότι πρόκειται για ένα από τα στοιχεία που θα μπορούν να εγγυηθούν ε, την βιωσιμότητα της γεωργίας. Αυτή είναι η πρώτη ερώτηση. Και δεύτερη ερώτηση. Η Διευθύνουσα Επιτροπή θα αντιμετωπίσει και το θέμα του ανταγωνισμού και της χρήσης των γεωργικών προϊόντων ε, δεδομένου ότι υπάρχει Ε, ουσιαστικά μια αφαίρεση και της γης αλλά και των προϊόντων που προορίζονται για την παραγωγή νέων ε, ειδών ενέργειας και όχι αποκλειστικά για τα τρόφιμα. Δηλαδή μπορούμε να φτάσουμε κάποια στιγμή στην έλλειψη πόρων, σε κάποια στιγμή που δεν θα έχουμε βεβαιότητα και βλέπουμε ότι υπάρχει, καθώς υπάρχει πολύ μεγάλη ανάγκη για τρόφιμα στο μέλλον, είναι ένα στοιχείο που πρέπει και αυτό να ληφθεί υπόψη. για να υπάρξει κάποια ποικιλία θα μιλήσω και εγώ στη μητρική μου γλώσσα κύριε Πρόεδρε να απαντήσω πρώτα ως εξής το καθήκον του Steering Committee δεν είναι, δεν είναι να φτιάξει μια νέα αγροτική πολιτική ή να αναπτύξει μια παγκόσμια αγροτική πολιτική. Διευθύνουσα Επιτροπή που έχει ως πρώτη στο καθήκον να ασχοληθεί με την έρευνα και τα προγράμματα ερεύνης. Ευχαρίστως όμως να εγκύψω λίγο στα επιχειρήματα που καταθέσατε. Ότι στα μέσα του αιώνα θα χρειαστούμε 70% παραπάνω τρόφιμα. Εδώ υπάρχει βέβαια και η δήλωση του Μπαν Κιμούν, Γενικού Γραμματέως του ΟΗΕ, που λέει ότι το 2030 θα χρειαζόμαστε 50% παραπάνω τρόφιμα. Και αυτή είναι η μεγαλύτερη πρόκληση στην πραγματικότητα. Και μάλιστα αυτό συμβαίνει διότι η αύξηση του παγκόσμιου πληθυσμού δεν είναι σταθερή. Έχουμε τώρα τους μεγαλύτερους ρυθμούς αυξήσεων και τις επόμενες δεκαετίες οι ρυθμοί αυτοί θα ε, γίνουν χαμηλότεροι. Οπότε έχουμε αυτή την, τις πρώτες δύο δεκαετίες του 21ου αιώνα την ταχύτερη αύξηση. Μικρό μέρος αυτών τροφίμων που χρειάζονται, που μπορούν να προέλθουν από πρόσθετες γιές. Το μεγαλύτερο μέρος των τροφίμων αυτών θα πρέπει να προέλθει από υψηλότερη απόδοση. Εκεί εντοπίζεται και το πρόβλημα το οποίο έχει σχέση βεβαίως και με τη βιωσιμότητα αλλά και με τα συμφέροντα, στο πω έτσι, της Επιτροπής Περιβάλλοντος. Δηλαδή Εάν κανείς κοιτάξει προς τα πίσω θα δει ότι στη διάρκεια μιας 20 ετίας περίπου κατέστη δυνατό να διπλασιαστεί η παγκόσμια παραγωγή τροφίμων. Αυτή, αυτός ο διπλασιασμός όμως απέβει τελικά σε βάρος του περιβάλλοντος. Η πραγματική πρόκληση είναι αυτή η παραπάνω παραγωγή που χρειαζόμαστε να γίνει εφικτή χωρίς παραπέρα επιβάρυνση του περιβάλλοντος. Ειδικά μάλιστα εδώ στην Ευρώπη όπου έχουμε και τις μεγαλύτερες αποδόσεις σε πολλούς τομείς πρέπει να επιτύχουμε να διορθώσουμε και τα σφάλματα του παρελθόντος και να διαμορφώσουμε μια ε, αγροτική οικονομία που να είναι φιλικότερη προς το περιβάλλον. Αυτή είναι η πραγματική πρόκληση. Το δεύτερο επιχείρημά σας της σπατάλης. Σωστό είναι το επιχείρημα αυτό. Γνωρίζουμε ότι κατά μέσον όρο στις βιομηχανικές χώρες 30 περίπου τις 100 των υφισταμένων τροφίμων πετιούνται τελικά στα σκουπίδια. Γνωρίζουμε επίσης ότι στις αναπτυσσόμενες χώρες ένα μεγάλο ποσοστό των τροφίμων χάνονται από ε, προβλήματα όπως κακές μεταφορές, όπως κακή αποθήκευση και ούτω καθεξής. Και εκεί λοιπόν αν σκεφτούμε αυτό το 30% της παγκόσμιας διατροφής τελικά μας λείπει. Υπάρχει εκεί λοιπόν ένα τεράστιο δυναμικό βελτίωσης και αυτός θα είναι ένας από τους κύριους στόχους της έρευνας. Το τελευταίο σας επιχείρημα, αυτός ο ανταγωνισμός δηλαδή για, ανάμεσα σε χρήση για τρόφιμα και σε χρήσεις, χρήσεις άλλες είναι ένα θέμα όπου τουλάχιστον στην Ευρώπη νομίζω ένα πράγμα πρέπει να είναι απόλυτα σαφές. Δεν χρειάζεται καν να διεξαγαγεί κανείς έρευνα. Είναι ζήτημα πολιτικών αποφάσεων. Ότι δηλαδή ότι το τρόφιμο πρέπει να έχει απόλυτη προτεραιότητα. Εξάλλου, είναι επίσης σωστό ότι στον τομέα της βιοοικονομίας, όπου δηλαδή τίθεται θέμα να χρησιμοποιηθεί βιομάζα για την παραγωγή διαφόρων χημικών ή για την παραγωγή ενέργειας ή και για την παραγωγή ε, θερμότητας. Εδώ πρέπει να ληφθούν υπόψη τα εξή. Πρώτα, πρέπει πρώτα να επικεντρωθεί αυτή η χρήση της βιομάζας ιδίως στα απόβλητα και απορρίμματα. Δεύτερο, θα πρέπει να διδαχθούμε από την δασοπονία. Στη δασοπονία υπάρχουν θεσπισμένες πλέον και παραδοσιακές χρήσεις που λένε ότι πρώτα πρέπει να χρησιμοποιηθεί η βιομάζα της, που προέρχεται από την παραγωγή δασοπονίας κατά τρόπο σταδιακό για το πρώτιστο είδος παραγωγής. Αυτή τη στατική δεν την έχει οθετήσει ακόμα η αγροτική οικονομία και απλώς για να προορίζονται για την καύση Νομίζω τα υλικά της βιομάζας που προέρχονται από την ε, αγροτική οικονομία δηλαδή είναι κρίμα. Μόνο για να χρησιμο... Επίσης, επίσης, ούτε είναι και το καλύτερη, καλύτερη δυνατή χρήση να χρησιμοποιηθούν για την παραγωγή υγρών καυσίμων. Είναι καλύτερα να χρησιμοποιηθούν και να γίνει προσπάθεια να αντικατασταθούν πέτροχημικές ύλες από ε, προϊόντα ή υποπροϊόντα της βιομάζας. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Χάιβη. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να θέσω μια ερώτηση. Εντός ε, του επιστημονικού προγράμματος υπάρχει και μια εμβάθυνση, μια θέση σε σχέση με τη γεωργία με χρήσιμο χιλιόμετρο, με μηδενικό χιλιόμετρο. Δηλαδή, ξέρετε ότι υπάρχουν διάφοροι προβληματισμοί στο θέμα σε επίπεδο παραγωγής και κατανάλωσης σε σχέση με την ανάγκη μιας επικράτησης. Θα ήθελα τη θέση σας για το θέμα αυτό. Also ich äh, habe nicht ganz verstanden, was... Κατάλαβα πολύ καλά την ερώτησή σας. Ε, χιλιόμετρο μηδέν. Υποθέτω ότι πρόκειται αυτό που λέμε σακίδιο διοξίδιο του άνθρακος. Δηλαδή αποτύπωμα μάλλον διοξίδιο του άνθρακος. Δηλαδή δεν έχει έννοια ένα προϊόν να παράγεται σε ένα σημείο και μετά να μεταφέρεται δεκάδες χιλιάδες χιλιόμετρα για να καταναλωθεί. Αυτό είναι θέμα. Είναι πολιτικό θέμα. Αλλά πρέπει να προσέξουμε. Για παράδειγμα. Για παράδειγμα. Η παραγωγή τομάτας. Μπορούμε εδώ κοντά στο Βέλγιο, πολύ κοντά εδώ να παραχθεί ντομάτα. Αλλά γι' αυτό βέβαια πρέπει να έχουμε θερμοκήπια. Και πρέπει να έχουν αναμένο το φως όλη μέρα για να παραταθεί η περίοδος ορίμανσης. Οπότε τελικά είναι χειρότερη επιλογή από το να είχαν παραχθεί αυτές οι ντομάτες στην Αφρική και να είχαν αποσταλεί στο Βέλγιο ή την Ολλανδία. Τι εννοώ λοιπόν. Πάντα πρέπει να έχουμε μια συνολική αντιμετώπιση για να μην κάνουμε λάθη. Πρόεδρος. Η κυρία Τόια. Ευχαριστώ. Καλημέρα κύριε Επίτροπε, κύριε καθηγητά Σίσερ. Εγώ είμαι στην Επιτροπή ΔΕΒ για την αναπτυξιακή συνεργασία και έχει προσκληθεί σε αυτή την συνάντηση. Η ερώτησή μου σχετίζεται περισσότερο με τις δικές μας δραστηριότητες. Θέλω να σας ρωτήσω, Πρόεδρε Φίσερ, αν είναι δυνατόν, όπως προσπαθήσαμε ήδη να προτείνουμε σε κάποιο εμπειρογνώμονα, να εντάξουμε θεματικές που ιδιαίτερα σκόπιμα θέσατε στο στόχαστρο ε, και τα θέματα που σχετίζονται με τους στόχους της χιλιετίας, ε, δηλαδή να μειώσουμε ως έναν βαθμό την πείνα στον κόσμο. Νομίζω ότι πρέπει να επενδύσουμε και σε αυτά τα θέματα, γιατί πρέπει να υπάρχει συρροχή των ευρωπαϊκών πολιτικών με τα θέματα τα παγκόσμια δηλαδή, τα θέματα των στόχων της χιλιετίας και μετά τη χιλιετία και επίσης το θέμα της υφαρπαγής των γεών. Ε, υπάρχουν πάρα πολλά έγγραφα του Κοινοβουλίου. Χθες ε, θέσαμε το θέμα της κλιματικής αλλαγής. Αν εμείς δεν αντιμετωπίσουμε και το θέμα της γης, πώς μπορούμε να μιλήσουμε για τρόφιμα. Και ξέρετε, υπάρχουν πάρα πολύ μεγάλα ενδιαφέροντα και μεγάλες αλλαγές στο θέμα της γης. Ε, land grabbing, φαρπαγή της γης, όπως θέλετε μπορείτε να το βάλετε, αλλά νομίζω ότι σε μια τέτοια διευθύνουσα επιτροπή τόσο σημαντική μπορείτε να εστιάσετε και στο σημείο αυτό. Σας ευχαριστώ. Λοιπόν, όπως ξέρετε, πρώτος στόχος της χιλιετίας είναι ότι μέχρι το 2015 πρέπει να μειωθεί κατά το ίμιση ο αριθμός των ανθρώπων που υποφέρουν από πείνα. Από ό,τι φαίνεται θα επιτευχθεί αυτός ο στόχος. Τώρα για τις συζητήσεις για τους ε, μετα τους στόχους μετά τη χιλιετία θέλουμε να πιστεύουμε ότι ο επόμενος στόχος θα πρέπει να είναι η εξάλληψη της πείνας. Αυτό βέβαια είναι μεγάλη πρόκληση. Συμπεριλαμβάνεται στο πρόγραμμά μας γιατί είναι ουσιώδης αυτός ο στόχος για το μέλλον της ανθρωπότητας. Δεύτερον, ένας άλλος τομέας ε, που μας ενδιαφέρει πάρα πολύ είναι η κλιματική αλλαγή. Είναι σαφές ότι οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής ποικίλουν από περιοχή σε περιοχή, ανάλογα με το κλίμα δηλαδή της κάθε περιοχής. Πρέπει λοιπόν να εξετάσουμε και να αντιμετωπίσουμε σωστά αυτές τις διαφορετικές επιπτώσεις. Και πρέπει να πω ότι για το θέμα αυτό η Ευρώπη θα μπορούσε να τα πηγαίνει και καλύτερα. Ξέρετε ότι υπάρχουν διάφορες ε, κλιματικές ζώνες στον κόσμο. Είναι πολύ πιο εύκολο κάποιες γεωργικές τεχνολογίες να μεταφερθούν από τη Βραζιλία στην Κεντρική Αφρική ή την Νοτιοανατολική Ασία παρά να τις μεταφέρεις από τον βορρά στο νότο. Και αυτό το διαπιστώνουν και τα ερευνητικά προγράμματα. Αλλά συνολικά η κλιματική αλλαγή είναι θεμελιώδες θέμα που μας απασχολεί. Τώρα για την αρπαγή γεών Αν διαβάσετε τις τελευταίες εκθέσεις από τους οργανισμούς, ε, τους αρμόδιους των Ηνωμένων Εθνών, θα δείτε ότι αναφέρονται στο πρόβλημα της έλλειψης δεδομένων. Αλλά φαίνεται, φαίνεται ότι πρώτα απ' όλα αυτό το φαινόμενο δεν έχει τις διαστάσεις ε, ή καλύτερα δεν έχει ως κύριο στόχο να μετατραπούν οι γέες αυτές σε καλλιεργήσιμες, αλλά κυρίως για λόγους επενδύσεων. Γιατί θεωρείται ότι η αξία της γης θα ανέβει, άρα είναι ελκυστική η επένδυση σε γέες. Νομίζω λοιπόν ότι χρειαζόμαστε καλύτερα στοιχεία πρώτα απ' όλα Και επιπλέον μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε μόνο μέσω διεθνής, διεθνούς ρύθμισης. Δεν μπορεί να υπάρξουν απλώς κρατικές ρυθμίσεις. Και πιστεύω ότι πρέπει να υπάρχουν παντού κτηματολόγια. Εάν υπάρχουν σωστά συστήματα καταγραφής των γεών, τότε η αγορά γεών γίνεται πολύ πιο διαφανής. Και η διαφάνεια είναι νομίζω σημείο κλειδί για να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα αυτό. Πρόεδρος. Ωραία, μάλλον η τελευταία ερώτηση από την κυρία Κυρία Μπριάνο, ναι, ένα σχόλιο και μια ερώτηση. Και για το χιλιόμετρο μηδέν συμφωνώ ότι πρέπει να υπάρχει μια παγκόσμια θέση, όμως γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό για μας ε, σε μια ευκαιρία όπως αυτή που μας δίνει η ΕΞΠΟ να αξιολογήσουμε τα θετικά προκύπτουν από το χιλιόμετρο μηδέν. Γιατί αυτό είναι σημαντικό για να δώσουμε ε, μία όθηση και μία ισχύ και στους δικούς μας ε, τοπικούς ε, παραγωγούς ε, και στην ε, δική μου περιοχή είμαστε σε συναγερμό νούμερο 2 και ξέρετε ότι πρέπει να δούμε και το θέμα και της εποχιακότητας των προϊόντων γιατί αυτό συνδέει το θέμα των τροφίμων με την περιβαλλοντική βιωσιμότητα. Θέλω να θέσω μια ερώτηση για την Αλία, γιατί και εγώ είμαι στην Επιτροπή για την Αλία. Μιλήσαμε πολύ για τη γεωργία, για τη βιωσιμότητα σε σχέση με τη γεωργία. Θα ήθελα να ρωτήσω αν προβλέπονται να υπάρχουν συζητήσεις ε, για την ε, βιωσιμότητα και την κατανάλωση προϊόντων αλίας. Ε, φορά και τις δικές μας παραδόσεις, αλλά θα θέλαμε και να δομηθεί μέσα σε μια οπτική βιωσιμότητα. Σας ευχαριστώ. Ναι, ευχαριστώ πολύ για την ερώτηση αυτή. Λοιπόν, σε ό,τι αφορά την περιφερειοποιημένη παραγωγή τροφίμων θα έλεγα ότι κάποιος θα μπορούσε να πάρει πολλά διδάγματα, ειδικά από την Ιταλία. Και από ό,τι βλέπω, αυτή η περιφερειοποιημένη παραγωγή τροφίμων και αυτά τα περιφερειοποιημένα συστήματα θα είναι ε, στην καρδιά του Ιταλικού περιπτέρου στην έξυπο του χρόνου. Νομίζω ότι εδώ η Ιταλία θα καταδείξει όχι μόνο τη σημασία της περιφερειακής παραγωγής, αλλά και τα πλεονεκτήματα και τη σχέση μεταξύ του γεωγραφικού πλαισίου και της ποιότητας. Και τα τελευταία έτη η Ιταλία έχει δώσει αγώνα για την προστασία ε, της, ε, της τοπικής της παραγωγής, ε, ξέρετε ότι έχουμε γεωγραφικές ενδείξεις κτλ. Προστατευμένη ονομασία προέλευσης. Όμως εδώ δεν χρειάζεται πολύ καινούρια έρευνα. Εγώ θα έλεγα απλά κάντε το. Ίσως θα μπορούσαμε να σκεφτούμε πώς μπορούμε να υποστηρίξουμε καλύτερα τέτοια συστήματα παραγωγής. Τώρα για την αλία. Σας, διασφελ... διαβεβαιώ ότι τα θαλάσσια συστήματα και το καλλιεργεία θα είναι τμήμα του προγράμματος της Διευθύνουσας Επιτροπής. Όλοι γνωρίζουν πόσο ευαίσθητα είναι τα θαλάσσια συστήματα αλλά αυτό που είναι λιγότερο γνωστό είναι οι συνέπειες της κλιματικής αλλαγής για αυτά τα συστήματα στο μέλλον. Ίσως θα υπάρχουν πολύ βαριές συνέπειες που δεν τις γνωρίζουμε ακόμα. Έτσι λοιπόν σε αυτό το τομέα θα έλεγα ότι πρέπει να γίνει πολύ περισσότερη και καλύτερη έρευνα και επίσης να χρησιμοποιηθούν και καλύτερες μεθοδολογίες για το πώς μπορούμε να παρατηρήσουμε την εξέλιξη των χθεοποθεμάτων μας. Ε, μου επεσήμανε ότι λαμβάνει η χώρα κάποια έρευνα και από το Κοινοερευνητικό Κέντρο. Χρησιμοποιούνται μέθοδοι γενετικής για να εντοπιστεί η προέλευση των τροφίμων. Έτσι ώστε μπορείτε να πείτε στη συνέχεια αν είναι σωστή η επισήμανση και αν όντω προέρχεται από εκείνη τη συγκεκριμένη περιοχή που αναφέρεται στην ετικέτα. Με τον τρόπο αυτό μπορούμε πολύ καλύτερα να εντοπίσουμε την προέλευση των τροφίμων, αλλά να βρούμε και όσους ε, καταχρώνται τη διαδικασία αυτή της προστασίας προέλευσης. Πρόεδρος, ωραία. Νομίζω ότι δεν έχουμε άλλες ερωτήσεις από τους συναδέλφους. Ε, ευχαριστούμε τον κύριο Φίσλερ για το πολύ χρήσιμο έργο του. και για τη δουλειά που κάνει για την επόμενη Expo. Σας ευχαριστούμε πολύ. Και τώρα θα κάνουμε μια μικρή αλλαγή. We invite here... Λοιπόν, έχουμε προσκαλέσει την Περιφερειακή Διευθύντρια του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για το επόμενο θέμα ringraziamo eh, Σας ευχαριστούμε που δεχτήκατε την πρόσκλησή μας. Την κυρία Σουζάνα Ιακέπ, ε, που είναι Διευθύντρια της Παγκοσμίας Οργάνωσης Υγείας. Και φυσικά περνάμε σε αυτό το σημείο της ημερησίας διάταξης, το σημείο 9, που αφορά μια ανταλλαγή απόψεων με την Περιφερειακή Διευθύντρια του ΠΟΕ για την επιδημία του έμπολα. Πρέπει να πω αντικειμενικά ότι εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, οι Ευρωπαίοι πολίτες παρακολουθούν με πολύ μεγάλη προσοχή τα όσα συμβαίνουν στη Δυτική Αφρική. Όχι μόνο λόγω των αριθμών επί των οποίων θα μας ενημερώσει η Διευθύντρια του ΠΟΗ, αλλά και επειδή υπάρχουν κάποιες ανησυχίες ότι ένα τόσο επικίνδυνος ιός θα μπορούσε να έλθει και εδώ στην δική μας Ήπειρο και να έχει επιπτώσει στην υγεία των πολιτών. Όπως έχει πολλές φορές και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, πρέπει να απομονώσουμε την νόσο και όχι τις χώρες, γιατί μόνο αν απομονώσουμε την νόσο και με πολύ μεγάλες προσπάθειες από την πλευρά όλων, θα μπορέσουν να μειωθούν βραχυπρόθεσμα να συνέπειε στη Δυτική Αφρική και επίσης να περιορίσουμε και τον κίνδυνο να διαδοθεί παγκοσμίως η επιδημία αυτή. Τους τελευταίους μήνες Είδαμε κάποιες ε, μεμονωμένες περιπτώσεις ε, ιατρικού προσωπικού, εθελοντών ε, που είχαν μεταβεί στην περιφέρεια για να αντιμετωπίσουν την όσο. Οι άνθρωποι αυτοί επαντεπατρίστηκαν σε ορισμένες χώρες αφού κόλλησαν την όσο. Ξέρουμε πολύ καλά πως ε, γίνεται η διαδικασία επαναπατρισμού αυτού του προσωπικού. Ξέρουμε ότι αυτό το θέμα είναι ακόμη ανοιχτό, υπάρχει επιτάπητος και σίγουρα μπορούμε να κάνουμε πολύ περισσότερα γι' αυτό. Εγώ πριν να δώσω το λόγο στη Διευθύντρια, θα ήθελα να την καλέσω να μας ε, περιγράψει τι μπορεί και τι πρέπει να κάνει η Ευρώπη κατά τη γνώμη της, έτσι ώστε να αναχαιτήσουμε, να κατεπολεμήσουμε την όσο στη Δυτική Αφρική, αλλά και κυρίως για να οργανωθούμε στην περίπτωση την οποία, που φυσικά δεν το ευχόμαστε, υπάρξει και παρουσία οποιοδήποτε κρούσματο και στην κλίμα και σίγουρα θα πρέπει να προετοιμαστούμε για να μην έχουμε αρνητικέ συνέπειε. Σα δίνω το λόγο για να σα ακούσουμε. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Πρόεδρε, κύριοι βουλευτές, κύριε και κύριοι, καταρχάς σας ευχαριστώ που με καλέσατε σε αυτή τη συνεδρίαση, επειδή είναι η πρώτη φορά που σας βλέπω σε αυτή τη νέα θητεία του Κοινοβουλίου θα ήθελα να σας ευχηθώ κάθε επιτυχία στην πολύ σημαντική και υπεύθυνη εργασία σας και σας διαβεβαιώνω ότι ο ΠΟΗ θα είναι πάντα στο πλευρό σας αν μας χρειαστείτε. Να δούμε πρώτα λοιπόν τα slide για το θέμα του έμπολα. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι έχουμε μια τεράστια πρόκληση ενώπιόν μας για να αντιμετωπίσουμε αυτή την επιδημία έμπολα βράχη πρόθεσμα με αποτελεσματικό τρόπο. Έχουμε μερικά θετικά στοιχεία ότι η επίπτωση δηλαδή των μέτρων που έχουμε λάβει μέχρι τώρα, για παράδειγμα στη Λιβερία, βλέπουμε να μειώνεται ο αριθμός των ε, ασθενών, αλλά πρέπει να τα ερμηνεύσουμε με μεγάλη προσοχή, διότι η επιδημία ακόμη προτρέχει της ε, ανταπόκρισης και μας ε, συνέλαβε χωρίς να είμαστε έτοιμοι ένας συνεργάτης μου που πέρασε 48 ώρες ε, στο κέντρο της περιοχής θεωρεί ότι μπορούμε να νικήσουμε αυτή την επιδημία στους επόμενους 6 με 9 μήνες. Ξέρουμε από τη δεκαετία του 70 τον ιό αυτό. Υπήρξαν επιδημίες στο παρελθόν και σύμβαιναν πάντα σε μικρά χωριά, σε διαφορετικά τμήματα της Αφρικής. Διαφορετικά από, ότι, από εκεί που συμβαίνουν τώρα. Και τις περισσότερες φορές τα ξεσπάσματα αυτά ούτε τα παίρναμε είδηση. Το κύριο στοιχείο αυτού του ξεσπάσματο, αυτής της επιθυμίας, είναι ότι συμβαίνει σε πυκνοκατοικημένε περιοχές, στο σημείο τομή τριών χωρών, κοντά σε μεγάλα αστικά κέντρα και με σημαντική κινητικότητα διαμεθοριακή και στο εσωτερικό των χωρών και αυτό επέτρεψε την ευρεία διάδοση του ιού. Και επιπλέον, καμία από τις τρεις χώρες αυτές δεν είχε τη δυνατότητα να αποτιμήσει και να διαχειριστεί αυτή την επιδημία με αποτελεσματικό τρόπο. Και έχουν αντιμετωπίσει δύσκολες περιόδους ε, μεγάλης φτώχειας, εμφυλίων πολέμων, αστάθειας και τα συστήματα υγείας τους είναι πολύ αδύναμα σε όλη την περιοχή. Και οι βασικές ε, υπηρεσίες υγείας δεν επέτρεψαν, δεν είχαν το επίπεδο που να επιτρέψει να αντιμετωπιστεί το ξέσπασμα. Αλλά Έχουμε και καλά νέα. Είναι δυνατόν να διακοπεί η αλυσίδα μετάδοσης του έμπολα και δεν είναι μόνο αυτή η πρώτη επιτυχία που αντιμετωπίσαμε, επιτυχία που επιτύχαμε, διότι στην Νιγηρία και στη Σενεγάλη μπορέσαμε να σταματήσουμε τη μετάδοση από ε, κρούσματα, που είχαν, ε, που είχαν, κρούσματα πολιτών που είχαν ε, ταξιδέψει σε αυτές τις χώρες. Ξέρουμε τι πρέπει να γίνει και έχουμε τον ε, σφαιρικό μηχανισμό, την παγκόσμια νομοθεσία υγείας για να επιτύχουμε αυτό που θέλουμε. Επειδή δεν έχουμε αυτή τη στιγμή ούτε εμβόλιο ούτε θεραπεία, η ανταπόκριση είναι μια σειρά βασικών μέτρων δημόσιας υγείας. Ε, έγκαιρη διάγνωση, παρατηρώντας τον πληθυσμό για να διαπιστώσουμε τα κρούσματα, να βοηθήσουμε τους ασθενείς, να τους απομονώσουμε και να συνεχίσουμε να παρακολουθούμε την ε, αλυσίδα μετάδοσης για να τη διακόψουμε. Και στο εσωτερικό των κοινοτήτων να ε, ε, διαδώσουμε ασφαλείς πρακτικές, ιδιαίτερα την ασφαλή αλλά και αξιοπρεπή ταφή. Θα ξέρετε όλοι ότι στις 8 Αυγούστου ο Γενικός Διευθυντής του ΠΟΗ δήλωσε ότι αυτή η επιδημία είναι επίγοντος χαρακτήρα διεθνής ε, πρόκληση με βάση τον κανονισμό για τη διεθνή αντιμετώπιση. Αυτό σημαίνει ότι χρειάζεται συντονισμένη διεθνής ανταπόκριση για να σταματήσουμε και να αντιστρέψουμε την πορεία μετάδοσης. Ο Γενικός Διευθυντής επίσης ενέκρινε τις συστάσεις της ε, Επιτροπής Επίγουσας Δράσης για να μπορέσουμε να έχουμε επίγοντα μέτρα για να σταματήσουμε τη διάδοση. Να συμπενθυμίσω Ποιε ποιες είναι αυτές οι προσωρινές συστάσεις που ισχύουν για όλες τις χώρες. Πρώτα απ' όλα τονίζω ότι ο ΠΟΗ δεν προτείνει γενική απαγόρευση διεθνών μετακινήσεων και εμπορίου. Προτείνει, προτείνει να εστιάσουμε, να ενισχύσουμε την ετοιμότητα σε όλες τις χώρες. Προτείνουμε να ελέγχονται οι εξερχόμενοι από τις χώρες και μαζί με τους εταίρους της η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας προσπαθεί να υπάρξει υψηλού επίπεδου εφαρμογή αυτών των ελέγχων. Έχει γίνει ήδη εξωτερική αποτίμηση. μια δεύτερη είναι σε φάση προετοιμασίας που θα γίνει από κοινού με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και χαίρομαι που μπορώ να σε ενημερώσω ότι τα αποτελέσματα της πρώτης αποτίμησης είναι πολύ θετικά. Παρά το ότι η Επιτροπή δεν συστήνει να απαγορεύονται οι συγκεντρώσεις, Καταλαβαίνει ότι αυτά τα θέματα είναι πολύ περίπλοκα και πρέπει να αποφασίζονται κατά περίπτωση. Η Επιτροπή ενθαρρύνει τα κράτη-μέλη να έχουν μια προσέγγιση με βάση την αποτίμηση του κινδύνου όταν αποφασίζουν αν θα απογορεύσουν συγκεντρώσεις. Και φυσικά θα συνεχίσουμε να τους βοηθάμε και να τους στηρίζουμε. Λόγω του μοναδικού χαρακτήρα αυτής της επιδημίας και της επίπτωσης σε όλους τους τομείς, το Συμβούλιο Ασφαλείας δημιούργησε για να αντιμετωπίσει την πρώτη ποτέ αποστολή αντιμετώπισης επίγοντος κινδύνου. Είναι προσωρινή αυτή η αποστολή και εμείς ε, είμαστε υπεύθυνοι για τον τομέα δημόσιας ασφάλειας. Η αποστολή των ΗΠΑ θα αντιμετωπίσει τις άλλες πλευρές, ασφάλεια, οικονομικά και ζητήματα ε, στήριξης. Να σε ενημερώσω τώρα για τη διεθνή προσπάθεια αντιμετώπισης. Ενεργοποιήσαμε τον κανονισμό και λόγω της απόφασης επίσης του Συμβουλίου Ασφαλείας είχαμε μια μεγάλη κλίμακας διεθνή ανταπόκριση. Και ευχαριστούμε πολύ για τη στήριξη που λαμβάνουμε, ιδιαίτερα από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη της. Έχουμε ένα πλήρες σχέδιο 90 ημερών για να ελέγξουμε και να αντιστρέψουμε την ε, εξάπλωση του ιού. Και επί τόπου δημιουργούμε τις αναγκαίες εγκαταστάσεις για την απομόνωση τουλάχιστον 70% των κρουσμάτων και τουλάχιστον 70% ασφαλούς ταφής των θυμάτων. Αυτοί είναι οι δύο στόχοι 60 ημερών. Για να έχουμε αποτελεσματική αντιμετώπιση θέλουμε σημαντικά μέτρα δημόσιας υγείας που ακόμη δεν έχουν υπάρξει. Για παράδειγμα, από τα 750 άτομα προσωπικού που προβλέπει το πλαίσιο για αντιμετώπιση, μόνο 155 άτομα είναι ήδη επιτόπου. Υπάρχουν 15 καταστάσεις αντιμετώπισης του έμπολα λιγότερο από ένα τρίτο από ό,τι θα θέλαμε. Θεωρούμε ότι με βάση τον οδικό χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και του ΠΟΗ χρειαζόμαστε τουλάχιστον ένα δις. Μέχρι στιγμής έχουμε συλλέξει περίπου τα μισά. Άρα επιγόντως χρειαζόμαστε επιπλέον πόρους, εκ των οποίων ο ΠΟΗ χρειάζεται περίπου 260 εκατομμύρια ευέλικτης χρηματοδότηση ε, προς το Ταμείο των Χορηγών. Συνοψίζω λοιπόν ποιε είναι οι ανάγκε για την επόμενη περίοδο, κέντρα αντιμετώπισης, ε, κρεβάτια σε αυτά τα κέντρα, προσωπικό, ιδιαίτερα ιατρικές ομάδες και επίσης ευέλικτη χρηματοδότηση. Πέρα από τα μέτρα δημόσιας υγείας, φυσικά χρειαζόμεθα μέσα θεραπείας και εμβόλια. Τάχιστα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα ασθένεια που θίγει τις ε, φτωχότερε χώρες και τα πτωχότερα τμήματα του πληθυσμού. Άρα τα εμπορικά κίνητρα για έρευνα και ανάπτυξη φαρμάκων δεν υφίστανται. Για τον έμπολα όλα τα μέτρα για την εξέβρεση φαρμάκων και ε, εμβολίων έχουν ήδη ληφθεί, γιατί, ληφθεί για την επίγουσα κατάσταση. Και για μελλοντική ετοιμότητα θα βοηθούσε πολύ να έχουμε ένα μηχανισμό που θα διασφάλιζε την διαθεσιμότητα και εμβολίων και φαρμάκων για αυτές τις παραμελημένες ασθένειες, αλλά και για τις άλλες ασθένειες της φτώχειας. Τώρα για τον έμπολα. Έχουμε ήδη δύο υποψήφια εμβόλια υπό ανάπτυξη, είναι σε προκλινικές φάσεις δοκιμών και έχουμε πέντε ενδεχόμενα εμβόλια που είναι υπό εξέταση. Τα δύο αυτά εμβόλια τώρα ε, είναι αντικείμενα δοκιμής σε ανθρώπους με ιδιαίτερες βέβαια διαδικασίες ασφάλειας. Αν όλα πάνε καλά, μπορεί να μπορέσουμε να αρχίσουμε να χρησιμοποιούμε τα εμβόλια στις χώρες ε, όπου έχουν σημειωθεί κρούσματα τον προσεχή Ιανουάριο. Άλλα προϊόντα επίσης ε, εξετάζονται για να αντιμετωπίσουμε τον ιό. Για παράδειγμα παράγωγα αίματος, όπως ο ιός ε, ανάρρωσης, αντισώματα, αιμογλομπίνη και αντιϊικά φάρμακα που έχουν δείξει ήδη ότι είναι αποτελεσματικά. Τώρα το θέμα που θίξατε κύριε Πρόεδρε. Τι κίνδυνο υπάρχει για την Ευρώπη. Να εστιάσω σε αυτό και να τονίσω ότι ο κίνδυνος για την Ευρώπη επιδημίας, εξάπλωσης του έμπολα είναι πολύ χαμηλός. Ε, άτομα που έχουν ταξιδεύσει στις χώρες όπου έχουν σημειωθεί κρούσματα επίσης ε, είναι πολύ απίθανο να μολυνθούν εάν ακολουθηθούν οι βασικές ε, διαδικασίες. Άτομα που έχουν ήδη μολυνθεί μπορούν να ταξιδέψουν στην Ευρώπη ο κίνδυνος ε, να μολύνουν άτομα του περιβάλλοντος τους ή επαγγελματίες υγείας είναι επίσης χαμηλός εάν εφαρμοστούν τα αναγκαία μέτρα. Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι αυτοί που έρχονται από αυτή τη χώρα και το προσωπικό υγείας καταλαβαίνουν τι είναι ο έμπολα, πώς μεταδίδεται και πώς μπορούν να προστατευτούν. Αυτά είναι ζωτική σημασία για την πρόληψη. Η αντίληψη για το τι κίνδυνος υπάρχει στην Ευρώπη είναι πολύ υπερβολική σε σχέση με, την, ε, με τον πραγματικό κίνδυνο. Οι αρχές δημόσιας υγείας πρέπει να ενημερώσουν λοιπόν την κοινή γνώμη αναλυτικά με διαφανή, έγκαιρο και σωστό τρόπο ούτω ώστε όλοι να κατανοήσουν γιατί θα είναι πλήρως ενημερωμένοι τι συμβαίνει και να θεωρήσουν ότι συμμετέχουν και οι ίδιοι ενεργά στην προσπάθεια πρόληψης. Γιατί λοιπόν λέω ότι είναι χαμηλός ο κίνδυνος, επειδή η Ευρώπη έχει ρωμαλαία συστήματα υγείας, είναι η καλύτερη εγγύηση αυτό ότι μια επιδημία έμπολα δεν θα προκύψει. Έχουμε ρωμαλαία συστήματα υγείας, ε, υπηρεσίες υγείας, αλλά πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Πρέπει να εργαστούμε για να ενδυναμώσουμε τα συστήματα υγείας και όπου υπάρχουν κενά αδυναμίες πρέπει φυσικά να καλυφθούν. Ιδιαίτερα να συνεχίσουμε τη δουλειά μας για να βοηθήσουμε να υπάρχει επαρκής δυνατότητα αντιμετώπισης. Σημεία εισόδου τώρα ταξιδιωτών που προέρχονται και που πηγαίνουν σε χώρες όπου εξακολουθεί να μεταδίδεται ο ιός. Τα σημεία λοιπόν εισόδου και εξόδου πρέπει να είναι τα σωστά σημεία για να δίδεται σωστή πληροφορία που να βασίζεται σε πραγματικά στοιχεία και να γίνεται η σωστή παρέμβαση. Κάποια κράτη-μέλη πρόσφατα έχουν εισάγει μέτρα ελέγχου, οπότε ενθαρρύνει τις χώρες που εφαρμόζουν τέτοια μέτρα να μας ενημερώσουν για την πείρα τους και τα διδάγματά τους. Αυτός ο έλεγχος μπορεί να έχει περιορισμένα αποτελέσματα, αλλά βοηθώντας και η είσοδος και ο έλεγχο κατά την είσοδο και την έξοδο, ο συνδυασμό αυτών των δύο μπορούν να βοηθήσουν. Αλλά πρέπει να αποτιμήσουμε και τι αποτέλεσμα έχουν γιατί είναι και πολύ απαιτητική από πλευρά σπόρων. Η ασφάλεια του προσωπικού υγιές είναι πολύ σημαντικό ούτως ώστε η ευγενή εργασία τους να μπορέσει να έχει την κατάλληλη απόδοση. Γιατί αυτοί υφίστανται τους υψηλότερους κινδύνους. Γι' αυτό το προσωπικό πρέπει να εκπαιδευτεί και να έχει το σωστό εξοπλισμό και να είναι σε πλήρη ετοιμότητα. Εάν κάποιος μολυνθεί πρέπει να του δοθούν όλες οι αναγκαίες φροντίδες. Όλα όσα χρειάζονται. Αυτό μας φέρνει στο θέμα της διακομιδής ασθενών και των κέντρων ε, αντιμετώπισης που πρέπει να υπάρχει και στις χώρες όπου υπάρχει μετάδοση του ιού και θέλω να ευχαριστήσω όλα τα κράτη-μέλη της Ένωσης που βοήθησαν ε, τις διακομιδές ε, προσωπικού από τη Δυτική Αφρική, προσωπικού υγείας. Τους ευχαριστούμε πολύ για αυτό, γιατί είναι ουσιώδης αυτή η προσπάθεια για να ενθαρρύνουμε προσωπικό υγείας να μεταβεί, να βοηθήσει αυτές τις χώρες. Υπάρχει πολύ καλή συντονισμένη αντιμετώπιση μεταξύ της Ένωσης και του ΠΟΗ στον τομέα της διακομιδής λοιπόν επόμενο. Να τονίσω επίση ότι η συνεργασία μεταξύ του ΠΟΗ, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ενός άλλου οργανισμού είναι πολύ ουσιώδης, βοηθάμε τα κράτη-μέλη για να υπάρχει υψηλότερη ε, ετοιμότητα για εμποραγικούς πυρετούς γιατί ο έμπολα είναι μοραϊκός πυρετός και για να έχουμε σε διεθνής, διεθνές επίπεδο το αναγκαίο δυναμικό. Σήμερα είναι ο έμπολα, αύριο μπορεί να είναι κάποιος άλλο ιός. Αυτό το ξέσπασμα έμπολα ήταν καμπανάκι για όλους μας και για πολλά κράτη-μέλη. Πρέπει να ολοκληρώσουμε τις προσπάθειές μας να έχουμε παρκές δυναμικό με βάση του Διεθνή Κανονισμού Υγείας για να αντιμετωπίσουμε τέτοια ξεσπάσματα. Και τέλος, καταλήγω ότι θα ξεπεράσουμε τον έμπολα εφόσον να αντιμετωπίσουμε σωστά στην πηγή αυτή την επιδημία και γι' αυτό πρέπει να επενδύσουμε όλα όσα μπορούμε για να ελέγξουμε αυτή την επιδημία στις χώρες όπου υπάρχει, δηλαδή στη Δυτική Αφρική. Αυτό πρέπει να είναι η αιστεία των προσπαθειών μας, να μην το ξεχνάμε ποτέ. Χάρη στη βοήθειά σας, κύριοι βουλευτές, θα συνεχίσουμε να αυξάνουμε το επίπεδο ανταπόκρισης στη Δυτική Αφρική γιατί κάτι τέτοιο χρειάζεται οπωσδήποτε και εκτιμούμε ιδιαίτερα την βοήθειά σας και ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ για την ενακτήρια τοποθέτησή σας. Έχουμε μακρό κατάλογο μελών που ζητούν να λάβουν τον λόγο για να θέσουν ερωτήσεις. Ας αρχίσουμε πρώτα με τον κύριο Τζον Ράιαν της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που εκτελεί χρέη διευθυντού. Αν θέλετε λοιπόν πέντε λεπτά. Καλημέρα. Μάλιστα κύριε Πρόεδρε πέντε λεπτά. Η Κομισιόν αυξάνει και αυτή τις προσπάθειές της για να συμβάλλει τις χώρες που πλήττονται από το, την επιδημία έμπολα με κάθε δυνατό τρόπο και να υποστηρίξουμε επίσης τις διεθνείς προσπάθειες των οποίων ηγούνται η, ε, των Ηνωμένων Εθνών για να μπορέσει να συγκρατηθεί η επιδημία των δυνατών σύντομότερο. Ταυτόχρονα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνεργάζεται με τις ευρωπαϊκές χώρες μέλη για να ασφαλίσει την ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση απέναντι στον ιό έμπολα. Όπως είπε η κυρία Ιάκαμπ, είναι χαμηλός ο κίνδυνος να ξεσπάσει επιδημία έμπολα στην Ευρώπη. Όμως ακόμα και αυτό το χαμηλό επίπεδο είναι αρκετά σημαντικό. Από την αρχή της επιδημίας η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει συνεργαστεί στενά με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, με το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου των Νόσων, τους άλλους ευρωπαϊκούς οργανισμούς και τις χώρες μέλη μέσω της Health Security Committee που θεσπίστηκε από πέρσι με ειδική απόφαση. Η συνεργασία αυτή επιτρέπει να αυξηθεί η ετοιμότητα, να γίνεται σημαντικότερη επαγρύπνηση, αξιολόγηση και διαχείριση του κινδύνου, κοινοποίηση των κινδύνων και ενημέρωση των πολιτών. Τονίζουμε επίσης ότι οι χώρες μέλη της Ένωσης διαβουλεύονται μεταξύ τους και μέσα στα πλαίσια της ε, Επιτροπής Ασφάλειας της Υγείας και με τους άλλους διεθνείς φορείς. Η Health Security Committee έχει συζητήσει παραπάνω από 20 φορές την επιδημία έμπολα από τον Μάρτιο του 2014 και έχει εκδώσει προφορίες προς ταξιδιώτες σε όλες τις ευρωπαϊκές γλώσσες με ε, τα κέρια μηνύματα Έχουμε κάνει εργασία ενημέρωσης σε αεροδρόμια, λιμένες κλπ. Για τρόπους για να εντοπιστεί το κρούσμα στη διάρκεια της πτήσης και για την αντιμετώπιση των κρουσμάτων έμπολα. Υπάρχει και σύστημα τώρα κοινοποίησης και έγκυρης προειδοποίησης μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το κέντρο της Στοκχόλμης για την αντιμετώπιση των νόσων έχει εκδώσει οδηγό και για την ε, αντιμετώπιση των κρουσμάτων αλλά και για τις διακομιδία στενών. Αυτά συζητήθηκαν και στην ε, άτυπη συνάντηση στο Μιλάνο των Υπουργών Υγείας 21 ε, και 22, 22 και 23 Σεπτεμβρίου και ενημερώνονται και επικαιροποιείται το επίπεδο ετοιμότητας. Ορισμένες χώρες μέλη μας λένε ότι δεν υπάρχουν επαρκείς ε, δυνατότητες αντιμετώπισης των κρουσμάτων και ούτε αρκετά ασφαλή εργαστήρια. Τα μέλη της Health Security ε, Commission έχουν, τώρα committee μάλλον, έχουν θεσπίσει συστήματα για να επιτρέψουν σε όλες τις χώρες μέλη να έχουν πρόσβαση σε ασφαλή εργαστήρια, καθώς επίσης και ασφαλείς κλίνες διεξήχθη εργαστήριο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή με συμμετοχή εμπειρογνωμόνων για να επανεξετάσουν μέτρα τα οποία θα πρέπει να ληφθούν για να μειωθεί στο ελάχιστο ο κίνδυνος να ξεσπάσουν δευτερεύοντα κρούσματα ε, έμπολα, δηλαδή από ε, μόλυνση από μολυσμένους ε, θεραπευτές ή νοσηλευτές και άλλους εργαζόμενους που μπορεί να έρθουν σε επαφή με τον ιό έμπολα για παράδειγμα ε, προσωπικό των αεροπορικών εταιριών. Έχουμε και ένα ε, δίκτυο τώρα κλινικών ιατρών οι οποίοι ανταλλάσσουν απόψεις για την αντιμετώπιση των κρουσμάτων έμπολα μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε ό,τι αφορά τον έλεγχο των εξερχομένων όπως είπε η κυρία Γιάκαμπ για τις αεροπορικές μεταφορές. Γίνεται η σχετική προσπάθεια από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις χώρες της Δυτικής Αφρικής και θα συνεχίσει τις επόμενες ημέρες για να δούμε πώς ε, προχωρεί αυτό το exit screening και ποιες βελτιώσεις μπορούν να επέλθουν σύμφωνα και με τις ε, συστάσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας που είναι πολύ σημαντικές για, και οι επαφές αυτές και με τους ε, νοσηλευτές ή το νοσηλευτικό προσωπικό και με τις ε, χώρες. Για την ενημέρωση του κοινού σύντομα θα διαθέσουμε ένα βίντεο για την ενημέρωση του κοινού και για τρόπους με τους οποίους μπορούν να αντιμετωπιστούν τα κρούσματα έμπολα. Σε ό,τι αφορά τώρα τον επαναπατρισμό ή την ε, ιατρική διακομιδία ασθενών, αναπτύσσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τώρα ίδιο σύστημα για τον επαναπατρισμό ε, νοσηλευτικού προσωπικού από τις ε, πληττόμενες περιοχές προς την Ευρώπη και ήδη ένα τέτοιο κρούσμα υπήρξε και ο ασθενής μεταφέρθηκε στη Γαλλία. Υπάρχει διακοπή του μικροφόνου. Τελειώνω. Ερευνούμε επίσης την δυνατότητα κοινή προμήθειας μέτρων, δηλαδή οι χώρες μέλη να αγοράσουν όλες μαζί προστατευτικό εξοπλισμό καθώς επίσης και εμβόλια. Αυτό ερευνάται. Και ο συνάδελφός μου επικεφαλής της Medicine Agency θα, ε, ε, θα αναφερθεί σε αυτό και γι' αυτό δεν θα επεκταθώ περισσότερο αλλά συζητούμε ήδη με την Επιτροπή Ασφάλειας Υγείας για να θεσπίσουμε διαδικασίες εφόσον φτάσει ένας ασθενής και χρειάζεται αμέσως ε, αντιμετώπιση η περίπτωσή του να υπάρχει σχετικός χάρτης. Σας ευχαριστώ. Μαξ Σπρέγγερ, ο Διευθυντής του Κέντρου Πρόληψης και Παρακολούθησης των Νόσων. Ευχαριστώ, καλημέρα σας. Καταρχήν να πω ότι ε, Δείχνω θέλω να δείξω την αλληλεγγύη μου σε όλα τα θύματα για τι οικογένειε ε, των θυμάτων. Ε, δεν είμαι σίγουρο αν τα αριθμητικά στοιχεία που είδαμε μα δείχνουν τον πραγματικό αντίκτυπο. Φοβάμαι ότι πραγματικά είναι υποτιμημένα τα νούμερα. Υπάρχει πολύ ενδιαφέρον των μέσων μαζικής ενημέρωσης, πολλές ιστορίες για τους ασθενείς ε, και για διάφορες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπου υπάρχουν υποπτά κρούσματα έμπολα και νομίζω ότι το έχουμε τώρα 17 υποπτές περιπτώσεις στην Ευρώπη. Η ευρεία πλειοψηφία αυτών ε, των ύποπτων περιπτώσεων ε, τελικά δεν ισχύουν γιατροί στην Ευρώπη τώρα έχουν ε, συνειδητοποιήσει τον εμπολά και αν κάποιος ε, εμφανιστεί σε ένα νοσοκομείο με πυρετό και προέρχεται από τις πληγήσεις χώρες, ε, υπόκειται σε ιατρικά τεστ. Συνήθως ο πυρετός προκαλείται και από άλλες νόσους και σήμερα έχουν τα νοσοκομεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση αντιμετωπίσει 9 περιπτώσεις έμπολα και οκτώ είδαν ιατρικό προσωπικό που επαναπατρίστηκε μόνο ένα ένα άτομο είχε τον ιό, είχε κολλήσει τον ιό στην Ευρώπη. Έτσι λοιπόν, εγώ θέλω να πω ότι ε, αυτός ο κινδύνος να δούμε περισσότερα κρούσματα στην Ευρώπη δεν θα φύγει αν δεν σταματήσουμε την επιδημία στη Δυτική Αφρική. Υποστηρίζω λοιπόν πλήρως το μήνυμα της κυρίας Γιάκαπ. Σύμφωνα με το ΠΟΗ και την Κομισιόν ότι υπάρχει επίγουσα ανάγκη για ουσιαστική διεθνή στήριξη για να ελέγξουμε την επιδημία. Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Προλήψη και Ελέγχου των Όσων παρέχει τεχνική υποστήριξη για τον έμπολα στην Κομισιόν ε, και στον ε, τομέα τη ασφάλεια τη υγεία. Όπω είπε ο Τζον συμμετέχουμε την εβδομαδιαία στην Επιτροπή για την Ασφάλεια τη Υγεία ε, και φυσικά απαντάμε σε κάποια αιτήματα που τίθεται από την Επιτροπή και έχουμε δώσει πλήρη προτεραιότητα στο θέμα από τον Αύγουστο. Είμαστε έχουμε 40 ε, εμπειρογνώμονες ε, που εργάζονται σε βάρδιες 24 ώρες το 24ωρο. Αυτό σημαίνει ότι γρήγορα μπορούμε να παρέχουμε τις ε, τεχνικές κατευθυντήριες γραμμές, εκθέσεις της κατάστασης και οτιδήποτε άλλο μας έχει ζητηθεί από την Επιτροπή. Και θέλω να σας αναφέρω δύο περιπτώσεις. Σχεδόν όλα τα κρούσματα που έχουν θεραπευτεί στην Ευρώπη είναι άνθρωποι που έχουν διακομιστεί από τη Δυτική Αφρική. Υπάρχουν που έρχονται στην Ευρώπη σε ελεγχόμενες συνθήκες. Και αν ακολουθούν όλες οι ορθές διαδικασίες, δεν υπάρχει κίνδυνος αυτοί να μολύνουν κάποιον άλλο. Όμως, ε, φυσικά στην πραγματική ζωή και στα πραγματικά νοσοκομεία δεν είναι τόσο εύκολο και αν εσείς το κάνετε σωστά είναι αρκετά δύσκολο ε, να βάλει κανείς και να βγάλει όλο το προστατευτικό εξοπλισμό που πρέπει να φοράει. Αν κάνει κανείς ένα μικρό λάθος μπορεί να μολυνθεί και το είδαμε αυτό στον Τάλλας αλλά και στη Μαδρίτη. Έτσι λοιπόν το ECDC έχει υπεράσχει ε, ένα λεπτομερή οδηγό για το ιατρικό προσωπικό για το πώς να χρησιμοποιούν σωστά τον εξοπλισμό πρόκειται για κάποιες κατευθυντήριες γραμμές που είναι διαθέσιμες ε, ελεύθερα στο διαδίκτυο. Επίσης, έχουμε δώσει κατευθυντήριες γραμμές για τα κράτη-μέλη για το πώς ε, να διαχειριστούν αυτές τις υποθέσεις και η Κομισιόν έχει δημιουργήσει ένα δικτύο για να συνδέσει τους γιατρούς ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση που μπορεί να πρέπει να θεραπεύσουν ασθενείς έμπολα εδώ στην Ευρώπη. Επίσης, τους ε, έχουμε μοιραστεί γνώσεις και αποτελέσματα για πειραματικές θεραπείες στο Κέντρο Πρόληψης και Έλεγχου των Νόσων και οι συνάδελφοι από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων συνεισφέρουν σε αυτό. Ε, Χθε μου στην Αφρική συνάντησα συναδέλφους από την Ιγυρία και τους ρώτησα ποιο είναι το θέμα κλειδί για να για την επιτυχία σας κατά του έμπολα και είπαν ε, πρόκειται για θέμα ηγεσίας, δέσμευσης και συντονισμού και νομίζω ότι το ίδιο ισχύει και για την Ευρώπη. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Τώρα να δώσω το λόγο στον κύριο Γκουίντο Ράζι, που είναι διευθυντής του ΕΜΑ, Οργανισμός Φαρμάκων. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Χαίρομαι πολύ που έχω δυνατότητα να σας παρουσιάσω τις δραστηριότητες που κάνει ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων, ΕΜΑ, για να συμβάλλει στην ε, συνολική αντιμετώπιση αυτού του ξεσπάσματος έμπολα. Αυτό το ξέσπασμα είναι μια σφαιρική επίγουσα ανάγκη δημόσια υγείας, γι' αυτό χρειάζεται η διεθνή συνεργασία για την αντιμετώπιση του. Όπως σωστά περιέγραψαν οι τρεις προηγούμενοι ομιλητές, βράχει πρόθεσμα, εξαρτώμεθα για τον έλεγχο της ασθένειας, από την ε, απομόνωση και την παροχή περίθαλψης στους ασθενείς. Αλλά μέσω και μακροπρόθεσμα, αν θέλουμε να εξαλείψουμε την νόσο, πρέπει να έχουμε εμβόλια και φάρμακα. Ο οργανισμός μου έχει συλλέξει τεκμηρίωση που θα επιτρέψει να συμβάλλουμε στην ανάπτυξη βασικών μεθόδων και φαρμάκων θεραπείας του έμπολα και ελπίζουμε και εμβολίων. Θέλουμε λοιπόν να επιταχύνουμε την ε, διαδικασία εξέβρεσης, αποτίμησης και εισαγωγής αυτών των φαρμάκων. Τι έχουμε κάνει μέχρι στιγμής. Ήδη τον Αύγουστο αρχίσαμε να συλλέγουμε την ε, βέλτιστη γνώση για το θέμα αυτό. Συναντηθήκαμε με όλες τις εταιρείες που αυτή τη στιγμή προσπαθούν να παραγάγουν τέτοιους, ε, τέτοια εμβόλια και κάθε φορά που είχαν ε, νέες ερωτήσεις ή νέα στοιχεία να μας δώσουν, αντιδρούσαμε αμέσως για να τους βοηθήσουμε να επιταχύνουν τη διαδικασία. Να υπάρξει, δηλαδή να παραχθούν τάχιστα εμβόλια και να εισαχθούν τάχιστα. Έχουμε ένα πλαίσιο ρυθμιστικό, έχουμε μια ταχεία διαδικασία παροχής επιστημονικών συμβουλών. Την προηγούμενη εβδομάδα χορηγήθηκε το πρώτο πιστοποιητικό για εμβόλιο με πρωτοφανώς ταχύ τρόπο. Και έχουμε και άλλες δυνατότητες υπό εξέταση. Δεν έχουμε προθεσμίες για υποβολή προϊόντων. Συνεχώς δεχόμεθα ενδεχόμενη υποβολή ετοιμάτων για προϊόντα για να ενθαρρύνουμε την ταχύτερη δυνατή παραγωγή εμβολίου. Είναι σημαντικό να έχουμε επίσης και έναν τρόπο για τη συλλογή των καλύτερων στοιχείων. Ξέρουμε ότι σε καταστάσεις ανάγκης, όπως τώρα, πρέπει να αντιδρά κανείς σύντομα και κάνουμε ό,τι μπορούμε για να επιταχύνουμε τη διαδικασία. Αν επιτύχουμε, θα είμαστε επίσης να αντιμετωπίσουμε καλύτερα οποιαδήποτε μελλοντική απευκταία βεβαίως ε, τέτοια ε, επιδημία. Έχουμε πολύ υψηλή επίσης συνέστηση των ευθυνών μας γιατί είμαστε ρυθμιστική αρχή άρα οι, μα πρέπει να βασίζονται σε, οι αποφάσεις μας πρέπει να βασίζονται σε στοιχεία και πρέπει να μπορούμε να δούμε αν ε, τα φάρμακα είναι όντως αποτελεσματικά αλλά και ασφαλή. Φυσικά δεν είναι δυνατόν να αποτύχουμε. Η ανάγκη δημόσιας υγείας μας απαγορεύει την αποτυχία. Μέχρι στιγμή έχουμε πολύ ενθαρρυντικές δηλώσεις από τις εταιρείες που προσπαθούν να αναπτύξουν αυτά τα φάρμακα, αυτά τα εμβόλια και αυτή τη στιγμή είμαστε προετοιμασμένοι να λάβουμε τα στοιχεία και ευελπιστούμε επίσης να χορηγήσουμε και την άδεια για, τα, για ανάπτυξη και ταχεία παραγωγή εμβολίων. Βεβαίω και εγώ και οι συνάδελφοί μου είμαστε απόλυτα αφοσιωμένοι σε αυτή την εργασία και σε στενή συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κέντρο Θεραπείας και Πρόληψη, τη CDC, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ελπίζω να καταφέρουμε να παραγάγουμε αυτό που χρειάζεται. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Και τώρα μπορούν να μιλήσουν οι συνάδελφοι. Πρώτο, ο κύριο Πέτα Λίζε. Σα ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ επίση όλους τους παρεμβάντες. Ε, μου φάνηκε πραγματικά πολύ ενδιαφέρουσα η ενημέρωση. Θα ήθελα να υποστηρίξω όλες και όλους εκείνους που τόνισαν ότι το πρόβλημα εντοπίζεται, η αιστεία του είναι δηλαδή στην Δυτική Αφρική και ότι δεν πρέπει να πανικοβληθούμε σε ό,τι αφορά την ενδεχόμενη κατάσταση που μπορεί να δημορφωθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα όσα συμβαίνουν εκεί στην Δυτική Αφρική πρόκειται βεβαίως για μια ανθρωπιστική καταστροφή και είναι καθήκον μας να δράσουμε εκεί, να βοηθήσουμε το δυνατόν συντομότερα και το δυνατόν περισσότερο αποτελεσματικά. Και όχι μόνο επειδή μπορούν να ξεσπάσουν και μονομένα κρούσματα και στην Ευρώπη, αλλά διότι εκεί κινδυνεύουν οι ζωές των ανθρώπων και διότι πολιτικά δεν μπορούμε να επιτρέψουμε στους εαυτού μας να αφήσουμε τους ανθρώπους αυτούς αβοήθητου. Και υπάρχει και αυτή η παρανοϊκή ιδέα ότι μπορούμε να αποκλείσουμε την περιοχή αυτή και να απαγορεύσουμε οποιαδήποτε ανταλλαγή ώστε να περιμένουμε με την ησυχία μας να πάψει αυτή η, να σταματήσει από μόνη της αυτή η καταστροφή. Φανταστείτε τι μήνυμα θα είναι αυτό για τους επιβιώσαντες εκεί. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να βοηθήσουμε με κάθε δυνατό τρόπο και ιδίως για να προσφέρουμε και μια προοπτική στους ανθρώπους αυτούς εκεί. Και αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο, για τον οποίο υποστηρίζω τον Παγκόσμιο Οργανισμό ε, ε Υγείας για τον ιατρικό επαναπατρισμό. Βεβαίως και ρωτούν πολλοί γιατί φέρνουμε στους ασθενείς αυτούς στην χώρα μας, στη Γερμανία. Έρθε και εκεί στο Αμβούργο ένας ε, από τους συνεργάτες του ΠΟΗ. Και εγώ ο ίδιος ως γιατρός πριν από πολλά χρόνια είχα δουλέψει σε μια αιστεία κρίσος και αναρωτιέται κανείς και τι συμβαίνει αν τελικά κολλήσω εγώ. Έπρεπε να ανεβώ σε ένα τζιπ και να μεταβώ τέσσερις ώρες μακριά για να φτάσω κάπου σε μια ε, πόλη όπου υπήρχαν κάποιες ε, δυνατότητες υποδοχής των ασθενών με κάποιες ευρωπαϊκές ή αμερικανικές προδιαγραφές. Πρέπει να κάνουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να βοηθήσουμε λοιπόν τα πρόσωπα αυτά. Ευχαριστώ ιδιαίτερα τον Μαξ Σπρέγγερ που είπε ότι μονάχα ένας ασθενής μολύνθηκε στην Ευρώπη. Γι' αυτό λοιπόν να αποφύγουμε οποιαδήποτε, οποιοδήποτε πανικό. Παρ' όλα αυτά ρωτώ τους εμπειρογνωμονές μας. Είμαστε, είναι όλες οι χώρες μας πραγματικά καλά προετοιμασμένες. Η Ισπανία απέδειξε ότι αντιμετώπισε το πρόβλημα. Μολύνθηκε μια ε, νοσηλεύτρια και αντιμετωπίστηκε ωστόσο το κρούσμα. Μπορούμε να θεωρήσουμε ότι όλες οι χώρες είναι πραγματικά εξοπλισμένες και προετοιμασμένες εφόσον χρειαστεί να γίνει και ένας ιατρικός επαναπατρισμός. Και τελευταία ερώτηση, κυρίως προς την κυρία Γιάκαμπ. Ακούσαμε πολλά για ενδεχόμενες θεραπείες, για εμβόλια. Η δική μου γνώμη είναι ότι είναι λάθος η στόχευση αυτή. Ενδεχόμενα λοιπόν τον Γενάρη θα μπορούμε να αρχίσουμε ιατρικές εξετάσεις. Αυτό δεν σημαίνει, ε, εμβολιασμούς. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα έχουμε ήδη το εμβόλιο και να είναι αποτελεσματικό. Θα δούμε δηλαδή αν θα λειτουργήσει και πόσα εμβόλια, πόσες δόσεις εμβολίων μπορούμε να αναμένουμε και ποιος θα λάβει τα εμβόλια που θα παραχθούν. Άρα το πρόβλημα δεν το αντιμετωπίζουμε έτσι. Το πρόβλημα θα το αντιμετωπίσουμε εάν ενημερώσουμε τον κόσμο, εάν φροντίσουμε καλά τους ασθενείς, εάν φροντίσουμε να υπάρχουν πραγματικά ισχυρά μέτρα υγιεινής, να ενισχύσουμε δηλαδή τα συστήματα υγείας και εφόσον έχουμε κάποια στιγμή το 2016 σε μεγάλε ποσότητε τα εμβόλια, τότε ίσω όμω υπάρχει κίνδυνο να είναι πολύ αργά πλέον. Γι' αυτό λοιπόν είμαι επιφυλακτικό όταν ρίχνουμε όλο μα το βάρο στην θεραπεία και στο εμβόλιο. Πρέπει να κάνουμε αμέσω και τι επόμενε εβδομάδε κάθε δυνατή προσπάθεια όπω εξήγησα. Ο κύριος Γκρότε, ευχαριστώ. Χαίρομαι πολύ που διεξάγεται η συζήτηση αυτή σήμερα εδώ διότι χρειάζεται πολλή συζήτηση και χρειάζεται πολλή διαφώτιση. Υπήρξαν πολλές περιπτώσεις κινδυνολογίας, πανικού και από τη δική μου μάλιστα εκλογική περιφέρεια όπου ένας απεσταλμένος ε, ιατρικής υπηρεσίας επανέρχεται από την Αφρική και ένας ντόπιο πολιτικός εκεί αρχίζει και φωνάζει προς Θεού θα γεμίσουμε έμπολα. Χρειάζεται λοιπόν πολλή ενημέρωση, πολλή διαφώτιση για να ενισχυθεί και η αποδοχή του κοινού απέναντι στα πρόσωπα αυτά. Νομίζω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση καθυστέρησε πολύ. Είδαμε πότε άρχισε η επιδημία και πότε αντιδράσαμε. Και οι άνθρωποι που πάνε εκεί να βοηθήσουν και στους οποίους προσφέρω τις εγκάρδιες ευχαριστίες μου, αυτούς τους εθελοντές και τις εθελόντριες που δηλώνουν ότι είναι διαθετηθημένοι να πάνε εκεί να βοηθήσουν. Οφείλουν οι άνθρωποι αυτοί να έχουν την ασφάλεια ότι δεν πρόκειται να ε, φέρουν το στίγμα μετά εφόσον επιστρέψουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Χρειαζόμαστε απαντήσει εδώ, ίσως από τον κύριο Σπρέγγερ, ίσως από την Κομισιόν, ίσως από τον ΠΟΗ. Πώς θα βελτιώσουμε την επικοινωνία για το θέμα αυτό. Αυτό είναι σημαντικός ρόλος που πρέπει να παίξουμε. Και επίσης όταν θα έχει κάπως χαλιναγωγηθεί η επιδημία, τι μπορούμε να βελτιώσουμε. Εγώ μαθαίνω ότι λείπουν απλούστατα πράγματα, λαστιχένια γάδια, προσώψια. Είναι αδιανόητο αυτό. Είναι δυνατό να μην υπάρχουν τα πράγματα αυτά. Θα έπρεπε οι προμήθειε αυτέ να είναι πολύ καλύτερε. Θα έπρεπε να γίνει πολύ καλύτερο συντονισμό των ευρωπαϊκών προσπαθειών. Γιατί πρόκειται για λεπτομέρειε. Θα πρέπει να αντιδράσουμε σε αυτά. Και σε ό,τι αφορά τον νοσηλευτικό προσωπικό. Είπε και ο Σπρέγγερ ότι μονάχα ένα πρόσωπο μολύνθηκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ξέρω ότι το προσωπικό των αεροπορικών γραμμών, τα νοσοκομεία έχουν μεγάλη ανάγκη από ενημέρωση, από πληροφόρηση. Πώς μπορούμε να βελτιώσουμε λοιπόν την πληροφόρηση αυτή, ώστε να μην περάσει τόσο πολύ χρόνος. Κοντεύει χρόνος που έχει ξεσπάσει η επιδημία του ιού έμπολα και αφήσαμε να περάσει όλος αυτός ο καιρός και υπάρχει σήμερα τέτοιο έλλειμμα ενημέρωσης. Εκεί πρέπει να στοχεύσουμε στις προσπάθειές μας. Και αφού τα είπα αυτά ευχαριστώ και πάλι όλες και όλους που δραστηριοποιούνται επιτόπου γιατί πρόκειται για πραγματική τραγωδία που παίζεται εκεί και επισκιάζεται βέβαια και από πολλές άλλες κρίσεις σε όλο τον κόσμο αλλά συχνά λησμονήθηκε η Αφρική. Σας ευχαριστώ λοιπόν που έχετε προσέλθει σήμερα εδώ και μας δίνετε την ευκαιρία να συζητήσουμε το θέμα αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Γκέρμπραντι. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ και την κυρία Τζέκα και του υπόλοιπου ομιλητέ που τοποθετήθηκαν για το θέμα αυτό. Ελπίζω να μην ε, είναι ε, πραγματικό για τη στάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ότι έχουμε τους πολλούς ανθρώπους που μιλούν για αυτό το θέμα και είμαστε υπεύθυνοι. Το πρόβλημα θέλω να επικεντρωθώ στην τελευταία διαφάνεια της ε, κυρίας ε, ε, με το ότι πραγματικό αγώνα δεν είναι στην Ευρώπη. Νομίζω ότι αυτό είναι απόλυτα σαφές. Όλοι οι εμπειρογνώμονες μας λένε ότι λειτουργούν πάρα πολύ καλά οι δομές της δημοσίας υγείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και λόγω αυτού είναι εύκολο να καταπολεμηθεί ο έμπολα. Έτσι λοιπόν, η πραγματική μάχη δεν είναι στην Ευρώπη, αλλά στη Δυτική Αφρική. Η ερώτησή μου στην κυρία Τζέικαμπ και θα ήθελα να την παροτρύνω να μην είναι πολύ διπλωματική στην απάντησή της. Είναι η εξή. Είστε ικανοποιημένοι με τον τρόπο που η Ευρωπαϊκή Ένωση συνολικά, ω σύνολο, αντιμετωπίζει αυτή την κρίση, ιδίω απέναντι στην Δυτική Αφρική. Γιατί ακούω ότι είναι ενεργοί η Γαλλοί στη Γουινέα, γιατί είναι γαλλόφωνη χώρα, οι Βρετανοί στη Σιερα Λεόνε, γιατί εκεί μιλούν αγγλικά και έχουν και ιστορικούς δεσμούς ότι στη Λιβερία έχουμε πολλά νοσοκομεία έμπολα κοντά το ένα στον άλλο και υπάρχουν άτομα από τη Σουηδία, τη Γερμανία, τη Δανία, αλλά από ό,τι φαίνεται δεν υπάρχει ένας ισχυρός συντονισμός. Και εγώ χαιρετίζω το ότι τα κράτη-μέλη βοηθούν, προσφέρουν νερογείς σε αυτές τις χώρες στη Δυτική Αφρική, όμως έχω την εντύπωση ότι χρειαζόμαστε μια πολύ περισσότερη ευρωπαϊκή προσέγγιση. Θεωρητικά έχουμε τα συστήματα για να το πράξουμε αυτό, έχουμε την πλατφόρμα για την κρίση, την αντιμετώπιση των κρίσεων που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για κάτι τέτοιο, όμως ακόμη δεν έχει χρησιμοποιηθεί. Και αν δω και ιδιαίτερα δύναμες δηλώσεις πριν δύο εβδομάδες και από το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων αλλά και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο την περασμένη εβδομάδα, δεν ε, έχω την πεποίθηση ότι τα κράτη-μέλη είναι πραγματικά πρόθυμα να επιτρέψουν ένα πιο ισχυρό ευρωπαϊκό συντονισμό. Έτσι λοιπόν θέλω να ρωτήσω την κυρία Τζέικα Είναι γεγονός ότι δεν έχουμε πράγματι μία ισχυρή ευρωπαϊκή προσέγγιση προς το συντονισμό στη Δυτική Αφρική και αυτό επίσης ε, έχει αντίκτυπο στην αποτελεσματικότητα της προσέγγισης της διεθνούς κοινότητας και έχει και αρνητικό αντίκτυπο στην προσέγγιση του Παγκοσμίου Οργανισμού Υγείας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Κυρία Ριβάζη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καλημέρα κύριε Γιάκαμπε. καθώ ε, τώρα είστε εκπρόσωπό του εμείς ε, θεωρήσαμε ότι ε, παλιά ήσασταν διευθύντρια του CDC. Σα γνωρίζουμε λοιπόν όμως ε, δεν ακούμε και πάρα πολύ τον ΠΟΗ, γιατί υπάρχει μια εσωτερική θέση που λέει ότι χρειαστήκατε 6 μήνες για να τη δράσετε. Είπαμε ότι το πρώτο κρούσμα ήταν ε, το Δεκέμβριο του 2013, αυτός ο νεορός ε, που κόλλησε έμπολα και το μετέδωσε στην οικογένειά του. Μετά φτάσαμε στο Μάρτιο, στις 24 Μαρτίου, και έξι μήνες μετά στις 8 Αυγούστου αντιδράσετε και είπατε υπάρχει εκτακτή ανάγκη. Έτσι λοιπόν αφήσατε κι εσείς ε, να διαδοθεί τόσο πολύ νόσος και δεν ε, κρούσατε τον κοδόνα του κινδύνου διεθνώς. Και εγώ νομίζω ότι είναι απίστευτο να μην ε, ακούμε τους γιατρούς χωρίς σύνορα εδώ το όνομά τους να μην αναφέρεται. Έχουν κάνει τεράστια δουλειά και κανένας ε, δεν μιλά για αυτούς τους οργανισμούς, για αυτές τις ενώσεις ε, που σύστησαν τα πρώτα νοσοκομεία για να προσπαθήσουν να κάνουν διάγνωση και να σώσουν τους ανθρώπους. Δεν ε, <laughs> αντέδρασε καθόλου η διεθνής κοινότητα. Δεύτερον, τώρα όλοι μιλούν για εμβόλια, για θεραπείες. Όταν διάβασα ένα άρθρο του 2012 έλεγαν ε, οι επιστήμονες, ο έμπολα δεν ενδιαφέρει κανένα, όμως ε, από το 76 έχουν πεθάνει 2.500 άτομα γιατί τα φαρμακευτικά εργαστήρια λένε δεν υπάρχει ε, επαρκής αγορά για κέρδος, έτσι λοιπόν δεν κάνουμε έρευνα. Εμείς στην Ευρώπη είχαμε ε, πολλές πρωτοβουλίες για τα καινοτόμα φάρμακα. Εγώ ήμουν σκιώδης εισηγήτρια για το θέμα αυτό και είπα πρέπει οπωσδήποτε να ενθαρρύνουμε τα καινοτόμα φάρμακα για τον έμπολο, αλλά έχουμε και το δέγκιο υπηρετό, έχουμε την ενονοσία. Ε, μου είπαν όλα αυτά να ενδιαφέρει τα μεγάλα εργαστήρια. Ε, κύριος Μπερόσο έδωσε 24 εκατομμύρια για αυτό το ταμείο για να ενθαρρύνει την έρευνα και μια ακόμη φορά δίνουμε στα φαρμακευτικά εργαστήρια δημόσια βοήθεια για να ενδιαφερθούν για αυτή την προβληματική. Είναι απίστευτο. Αυτό σημαίνει ότι οπωσδήποτε και στο πλαίσιο του ΕΟΦ ε, και στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψη ε, και Ελέγχου των Νόσων να συμμετέχουν και μη κυβερνητικέ οργανώσει. Γιατί διαφορετικά ε, θα έχουμε φάρμακα μόνο για τη χολυστερίνη, το διαβήτη, την παχυσαρκία. Έτσι λοιπόν, εγώ εδώ θα σα απευθύνω μία έκκληση, γιατί είναι και εδώ και ο Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων και ο Παγκόσμια Οργάνωση Υγεία. Σε, σε ποια πλαίσια κάνουμε αυτές τις κλινικές δοκιμές. Δηλαδή γίνονται στη Σιέρα Λεόνε, γίνονται στη Λιβερία, γίνονται στη Γουινέα και με ποια ηθική. Γιατί αν έχουμε ένα εμβόλιο, πολύ ωραία, αλλά θα είναι πολύ αργά. Πάντως πρέπει να το δημιουργήσουμε, αλλά θα πρέπει να είμαστε σίγουροι γιατί θα εμβολιάσουμε και παιδιά που θα είναι υγιεί και εγγύες γυναίκες κτλ. Θα πρέπει λοιπόν να πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις για να υπάρχει το εμβόλιο και να θεραπεύει. Τώρα, για το κατεπήγον. Εγώ να σας πω ότι έχω μελή της οικογένειας μου ε, που έρχονται από τους γιατρούς χωρίς σύνορα και λένε είμαστε εκτός ελέγχου. Εδώ εκρήγνεται παντού η ασθένεια γιατί εκεί δεν υπάρχουν ε, οι συνθήκες υγειονομικές όπως στην Ευρώπη, αναπτύσσεται δραματικά και 10 με 15.000 άνθρωποι έχουν μολυνθεί και μόνο στα νοσοκομεία έχουμε 300-400 θέσεις και τη νύχτα παίρνουν όλους τους νεκρούς και μετά από 10 λεπτά έχουν καταληφθεί όλα τα κρεβάτια. Περιμένουν άπειροι άνθρωποι στο νοσοκομείο. Υπάρχει λοιπόν τεράστια ανάγκη, είμαστε σε κατάσταση κατεπίγουσα. Θα πρέπει όμως εδώ ε, να σταματήσουμε αυτή το πηγή μόλυνσης και λέτε «Α, στην Ευρώπη είναι μικρός εκείνο περιμένετε αν έρθουν 10-20 περιπτώσεις στη Γαλλία θα έχουμε πάρα πολύ δύσκολες καταστάσεις για να διαχειριστούμε». Πρέπει όλα λοιπόν ε, να τα δούμε στο επίπεδο αυτοχωρών και για δεν είπα Αντέδρασε ο κύριος Ομπάμα, είπε «Θα στείλουμε 3.000 ε, στρατιώτες, πολύ καλά, στρατιωτικούς». Όμως ε, υπάρχουν πάρα πολλοί λίγοι άνθρωποι από τη σκοπιά των ανθρωπίνων πόρων για να καταρτήσουν του ανθρώπου εκεί επί τόπου, γιατί δεν υπάρχει καμία κινητοποίηση στην Ευρώπη για να στείλουμε νοσοκόμου και γιατρού. Γιατί οι άνθρωποι φοβούνται. Και εσεί σε επίπεδο ΠΟΗ περιμένω να έχετε ένα πιο ισχυρό λόγο, ένα πιο στενερό λόγο, είστε πολύ αδύναμοι. Λέτε τι θα γίνει. Όχι και μου είπε, το σταματήσαμε στην Ιγυρία, δείτε την κατάσταση στην να Φάσο. Αν ξεκινήσει ποτέ εκεί, μπορεί να αναπτυχθεί πάρα πολύ δεδομένη και τη ασταθούς κατάσταση στην Αφρική. Τώρα, τι θα κάνει ο ΠΟΗ, τι θα κάνει η Κομισιόν για να εγγυηθεί την ε, πιστιστική βοήθεια και σε επίπεδο προσωπικού, γιατί βρισκόμαστε σχεδόν σε μια κατάσταση πολέμου σε εκείνες τις χώρες. Εμένα πραγματικά ε, με ανησυχεί ο λόγος σας, με ενοχλεί, δεν καταλαβαίνετε τη σοβαρότητα και όλοι οι άνθρωποι που έρχονται από αυτές τις νόσες, από αυτούς τους οργανισμούς έρχονται εδώ τραυματισμένοι. Πώς σας πήρε έξι μήνες για να απαντήσετε, νομίζω ότι θα έπρεπε να έχετε πιο στενερό λόγο για το θέμα αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Και τώρα ο κύριος Ιουαρίστια Μπάουντς. Και σας παρακαλώ ε, να είστε λίγο πιο σύντομοι γιατί όλοι θέλουν να μιλήσουν. Καλημέρα σας. Θα επιμένω λιγάκι σε αυτά που είπε η κυρία Ρίβας. Κυρία Ρίβασή, διότι μας είπατε ορισμένα θετικά, αλλά και εγώ έχω μιλήσει με τους ε, ιατρούς χωρίς σύνορα και λένε ότι επιτόπου η επιδημία συνεχίζει να είναι εκτός ελέγχου. Και είπατε ότι όλα πάνε καλά θα έχουμε εμβόλιο τον επόμενο Γενάρη. Κατά τη γνώμη μου αυτό δεν ε, συμφωνεί με αυτά που είπε την προηγούμενη εβδομάδα η Γκλάξο, η φαρμακευτική εταιρεία. Γιατί είπε ότι το εμβόλιο ούτως ή άλλως θα έρθει καθυστερημένα, πολύ αργά. Δεν ξέρω εάν η Ευρωπαϊκή Ένωση κάνει ό,τι μπορεί για να αποφευχθούν αυτές οι καθυστερήσεις από τις οποίες υποφέρουν οι ασθενείς στην Αφρική. Επίσης οι, αθε... οι, υποσχέσεις που αθετήθηκαν, η βοήθεια που δίνεται σταγόνα σταγόνα, η κατάρρευση των συστημάτων Αφρικής, η κατάρρευση των πάντων. Υπάρχει πολύ υψηλή έμεση θνησιμότητα λόγω αυτής της ασθένειας. Γιατί περιπτώσεις για παράδειγμα ελονοσίας, διάρειας ε, δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν. Ή γιατί δεν υπάρχει βοήθεια για, τις, ε, για τους τοκετούς. Όπως καταλαβαίνετε παρά τότε την τεράστια θνησιμότητα που έχει η έμπολα, ε, σκοτώνει πολύ λιγότερα άτομα από την ελονοσία για παράδειγμα ή την ε, έλλειψη σωστής διατροφής. Στείλαμε μερικά εκατομμύρια, είπαμε ότι θα στείλουμε και περισσότερα μέσω μακροπρόθεσμης αναπτυξιακής βοήθειας. Αυτά είναι ανεπαρκή. Είναι ανεπαρκή. Και δυστυχώς η κοινή γνώμη στην Ευρώπη ανησυχεί πολύ περισσότερο για όσε περιπτώσει ενδεχόμενα μπορεί να υπάρξουν στην Αφρική. Ενώ τα κρούσματα είναι πολύ. Στην Ευρώπη, συγγνώμη, ενώ τα κρούσματα είναι πολύ περισσότερα στην Αφρική. Όπω είπε και ο Τζον Ράιαν, μιλήσαμε πολύ περισσότερο για το τι επίπτωση μπορεί να έχει στην Ευρώπη από το τι κάνουμε για να αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικά στην Αφρική το πρόβλημα. Και εγώ πιστεύω ότι και τα Ενωμένα Έθνη και η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν τήρησαν τις υποχρεώσεις και δεν ανταποκρίθηκαν στις επίγουσες εκκλήσεις που έγιναν επί τόπου από οργανισμούς όπως οι Ιατροί Χωρίς Σύνορα εδώ και πολλούς μήνες. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ λέει ο Πρόεδρος. Ο συνάδελφος Πεντιτσίνη. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ και όλους τους συζήτητες που άνοιξαν αυτή τη συζήτηση. Εγώ θα ήθελα να επανέλθω στο θέμα των εμβολίων, γιατί το είπε η κυρία Τζάκα πριν. Το μήνυμα ήταν κάποιο περισσότερο καθιστικαστικό γιατί μας είπε ότι έχουμε πέντε εμβόλια σε πειραματικό στάδιο και μας είπε ότι αυτό το πειραματικό στάδιο θα υλοποιηθεί με επιταχυμένα πρωτόκολλα. Όμως, ε, όπως ε, είπε ο προηγούμενος ομιλητής, η Glaxo, η φαρμακευτική εταιρεία ε, η οποία έχει αναλάβει να δημιουργήσει αυτό το εμβόλιο σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, είπε πριν ε, λίγο ένα μήνα ότι στις αρχές του Ιανουαρίου 2013 θα ήταν ε, έτοιμες πάνω από 10.000 δόσεις αυτού του εμβολίου χάρη και στην έγκριση της FDA τον είπα που είχε δώσει η FDA για τα εκούσια πειράματα στον άνθρωπο. Τώρα πριν λίγες μέρες ο επικεφαλής του ερευνητικού προγράμματος της Κλάξο είπε ότι δυστυχώς επιστρέφουμε σε ένα παραδοσιακό πρωτόκολλο γιατί χρειάζονται νέες δοκιμές φάσης για την τοξικότητα ε, και νέα τεστ για δεύτερου σταδίου για την αποτελεσματικότητα και νέες δοκιμάσεις για να καθοριστεί η δόση, δηλαδή στα 2-3. Τώρα εμείς αναρωτιόμαστε τι συνέβη και πόσο μπορούμε να εμπιστευτούμε αυτά τα, τα μηνύματα, τα καθιστικαστικά που ακούγονται σήμερα. Γιατί πριν λίγο καιρό είχαμε πει στις αρχές του 2015 θα είναι έτοιμο ένα εμβόλιο, ενώ τώρα ο επικεφαλής του προγράμματος της Γκλάξο μας είπε ότι λόγω όλων αυτών των τελευταίων δοκιμών δεν μπορεί το εμβόλιο να θεωρηθεί ως ε, μία απάντηση στην επιδημία. Έτσι λοιπόν, πώ από ένα τέτοιο επιτυχημένο πρωτόκολλο πήγαμε σε ένα πρότυπο πρωτόκολλο, σε ένα στάνταρ πρωτόκολλο και σε ποιο στάδιο βρίσκεται ο πειρασματισμός για τις άλλες βιομηχανίε και επίσης πώς θα γίνει η εμπορία του φαρμάκου σε αυτές τις δραματικές συνθήκε. Ευχαριστώ. Κυρία Σιλεπερίκ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Το θέμα αυτό το συζητούμε εδώ και καιρό. Και είμαι πολύ ικανοποιημένη που επιμείνατε κύριε Πρόεδρε να μπει το θέμα στην ημερησία διάταξη και να, δεχθούμε, να υποδεχθούμε όλους αυτούς τους εμπειρογνώμονες. Έχω μια ερώτηση τώρα προς το Ευρωπαϊκό Κέντρο Παρακολούθησης Νόσων. Δεν έχει φτάσει ο ιός στην Ευρώπη ακόμη, αλλά μπορεί να φτάσει όμως. Η ερώτησή μου λοιπόν είναι πώς θα το αντιμετωπίσουμε τότε. Νομίζω το να αναμένουμε ότι θα συγκρατηθεί εκεί όπου είναι τώρα είναι η παραπλουστευτική λύση. Τι επαφές έχετε επίσης με την Αφρική, εσείς κυρία Γιακάμπ. Είπατε ότι η Νιγηρία μπόρεσε και αντιμετώπισε καλά τον κίνδυνο. Έχετε επαφέ με αυτού. Ερώτηση που υποβάλλω και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και το πιο σημαντικό ερώτημα που με απασχολεί. Μιλήσαμε για το θέμα αυτό πολύ καιρό. Εκτό από τα 500 εκατομμύρια. Απαιτείται ανθρωπιστική βοήθεια και κόσμο να πάει κόσμο εκεί να βοηθήσει. Πώ μπορούμε να το πετύχουμε αυτό. Είναι σημαντικό αυτό. Δεν θα χρειαστεί κάποιο σχέδιο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να αντιμετωπίσει και το μέγα πρόβλημα των ορφανών. Δεν μπορούν να μείνουν στη μοίρα τους. Όλοι θέλουν να δείξουν ότι κάτι κάνουν, οι Βέλγοι, οι Ολλανδοί, αλλά θα πρέπει να μιλήσουμε όλοι με μια φωνή. Και αυτό ε, αφορά και τους ελέγχους στα αεροδρόμια. Και τώρα την πρόεδρο Σπανιό. Ευχαριστώ πολύ την κυρία Γιακάμπ για την παρέμβασή της, για αυτά που κάνει ως διευθύντρια του ΠΟΗ για την Ευρώπη. Ξέρουμε ότι ήταν επίσης διευθύντρια, η αρχική διευθύντρια του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Πρόληψης ε, και Θεραπείας Νόσων που στις αρχές της δεκαετίας ε, είχε ήδη επαφές μαζί μας για να ε, καθοριστεί μια πολύ σωστή πολιτική θεωρώ για την καταπολέμηση των μολυσματικών ασθενειών. Θα ήθελα να ασχοληθώ με δύο θέματα. Το πρώτον, ήμουν εισηγητής της απόφασης που λάβαμε αρχές του έτους για τις ε, σοβαρές ε, διαμεθοριακές απειλές κατά της υγείας. Και χαιρετίζω την ε, παρέμβαση του κυρίου Ράιαν της Γενικής Διεύθυνσης Υγείας που προσωπεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, διότι η εργασία αυτή μας πήρε δύο χρόνια, θα θυμάστε, ότι υπήρξε τεράστια σύγχυση στην Ευρώπη το 2009 όταν χρειάστηκε να αντιμετωπίσουμε την πανδημία της γρήπης HSN1 και γι' αυτό υπήρξε ανισότιμη αντιμετώπιση των Ευρωπαίων λόγω αυτής της σύγχυσης. Γι' αυτό απευθύνομαι σε εσά, κύριοι συνάδελφοι. Γιατί όπως θα θυμάστε, όταν ε, ξεπεράσαμε αυτή τη γρήπη, διαπιστώσαμε ότι πρέπει να υπάρξουν πρωτοβουλίες από πλευράς του Κοινοβουλίου και της Κομισιόν έναντι των κρατών μελών για να καταλήξουμε σε μια καλύτερη αντιμετώπιση. Τώρα υπάρχει η Επιτροπή Υγειονομικής Ασφάλειας που συνεδριάζει πολύ συχνά στο Λουξεμβούργο και από τότε που ξεκίνησε η επιδημία έμπολα που είναι πολύ σοβαρή απειλή. Θυμάστε τα στοιχεία. Εδώ στην Επιτροπή μας κάναμε μια συζήτηση την 3η Σεπτεμβρίου. Σε δύο μήνες έχουμε 10.067 άτομα που μολύνθηκαν και 3.051 που κατέληξαν στη Δυτική Αφρική λόγω της νόσου. Όπως είπε και η κυρία Διευθύντρια, όπως είπατε και εσείς κύριοι διευθυντές, αντιμετωπίζουμε μια μάστιγα. Πρέπει να διεξαγάγουμε έναν πόλεμο εναντίον της. Εάν λοιπόν το πρώτο που είπα αφορά τι κάναμε και τι επιτύχαμε κατά την προηγούμενη θητεία για να μπορέσουμε να έχουμε σωστές αποφάσεις, καρπός αυτών των εργασιών μας και τις ε, προσπάθειες που κάναμε έναντι των κρατών μελών και δεν ήταν εύκολο να επιτύχουμε αυτό που επιτύχαμε, διότι τα κράτη-μέλη δεν ήθελαν να υπάρξει αυτή η απόφαση. Καρπός λοιπόν είναι αυτή η απόφαση. Αλλά ο συσχετισμό δυνάμεων, ο συσχετισμός δυνάμεων μας επέτρεψε να καταλήξουμε σε αυτή την απόφαση και στα μέτρα που απορρέουν. Βεβαίω ε, λυπάμαι, λυπάμαι βεβαίω, χωρί αυτό να είναι δική μα ευθύνη ούτε του κυρίου Τζον Ράιν, λυπάμαι λοιπόν που όταν αυτές τις ε, τελευταίες εβδομάδε και μήνες λήφθησαν αποφάσεις από τα κράτη-μέλη, δεν έγινε καμία αναφορά στις προσπάθειες που γίνονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Κάθε φορά τα κράτη-μέλη λένε εμείς πήραμε πρωτοβουλίες. Όχι. Εκείνοι βασίστηκαν στις δικές μας ε, πρωτοβουλίες, στις πρωτοβουλίες της Επιτροπής ε, για Υγειονομικά Θέματα που επέτρεψαν να έχουμε αποφάσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο για να προστατεύσουμε τους πολίτες μας, τα 500 εκατομμύρια πολιτών μας, από μια τόσο σημαντική μάστιγα όπως είναι ο ιός έμπολα. Πιστεύω ότι είναι χρήσιμο να το επενθυμίσουμε αυτό, γιατί θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε τόσους αντιπάλους ε, της ευρωπαϊκής οικοδόμησης που χρειάζεται να πούμε ότι να, στον τομέα αυτό μπορέσαμε να προστατεύσουμε τους Ευρωπαίους. Το δεύτερο που θέλω να πω είναι ένα σημείο που προκαλεί πολλές αντιδράσεις. Το είπατε κι εσείς ε, και το υπενθύμησαν και καποιοι παρεβαινοντες παρεμβαίνοντες. Σήμερα ακόμη υπάρχουν κράτη-μέλη και ευρωπαϊκά λοιπόν, κράτη-μέλη της Ένωσης που δεν έχουν αντιληφθεί τις διαστάσεις της οικονομικής συμβολής που πρέπει να υπάρξει. Πρέπει λοιπόν να απαιτήσουμε συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών υψηλότερες χρηματοδότηση και επιτόπου στη Δυτική Αφρική όπως είπατε κύριε Διευθύντρια, ξέρουμε πολύ σωστά ότι αν θέλουμε πραγματικά να έχουμε τα κέντρα αντιμετώπισης και τα κρεβάτια, χρειαζόμαστε ένα δις. Αλλά μέχρι στιγμής έχουμε μόνο τα μισά. Άρα πείτε το, πείτε το ως ευρωβουλευτές, πείτε το στις κυβερνήσεις σας και πείτε το και ευρύτερα. Παρακαλώ να υπάρξει αυτή η χρηματοδότηση για το σύνολο των μέτρων που θα μας επιτρέψουν να εξαλείψουμε αυτή τη μάσκα επί τόπου. Γιατί αν δεν αντιμετωπιστεί επί τόπου, ό,τι και να κάνουμε θα συνεχίσουν οι ανησυχίες και εδώ στην, Αφρική, στην Ευρώπη. σήμερα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Η κυρία Ντορνάν. Ευχαριστώ. Κυρία Διευθύντρια, ο δικό χάρτη ε, που έχει προταθεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μα φαίνεται μη πλήρης. Πρέπει να βρούμε τα πρακτικά και συγκεκριμένα μέτρα να καταπολεμήσουμε τον ιό και θα ήθελα να μου πείτε αν ο ΠΟΗ λαμβάνει υπόψη την ουσιαστική πτυχή ε, που αφορά η διαχείριση των μεταναστευτικών ροών ε, όχι μόνο από του τόπου διέλευση αλλά και στα σύνορα για να προστατεύσουμε την Ευρωπαϊκή Επικράτη από τον έμπολα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Καμπιόν Ρουίς. Ευχαριστώ πρόεδρε. Εγώ θα ήθελα να πω καταρχήν ε, ότι ε, άκουσα πολύ ευχάριστα τις παρεμβάσει, λαμβάνοντας υπόψη ότι τελικά η διεθνής κοινότητα συνειδητοποίησε, αντιλήφθηκε το μέγεθος ε, της επιδημίας το Συμβούλιο μέχρι τις 20 Αυγούστου δεν είχε οθετήσει καθοριστικές αποφάσεις. Ε, ε, τώρα όμως ε, έχει τεθεί σε ισχύ ένα σχεδόν 90 ημερών. Εγώ νομίζω ότι όλα αυτά είναι σημαντικά. Έχω όμως μια αμφιβολία μήπως αυτό αυτό ουσιαστικά τέθηκε σε εφαρμογή επειδή υπήρχαν τα πρώτα κρούσματα του Εύβολα στην Ευρώπη. Και πέρα από αυτέ τι πρόοδου, θεωρείτε ότι αρκούν οι προσπάθειε που έχουν ολοκληρωθεί, που έχουν υλοποιηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή θα χρειαζόταν κάτι περισσότερο. Έχει γίνει πολύ σημαντική προσπάθεια, αλλά εγώ θα ήθελα να μα εξηγήσετε αν όλα αυτά επαρκούν ή αν πιστεύετε ότι χρειαζόμαστε και κάτι παραπάνω για την Ισπανία. Θα ήθελα να κάνω κάποιε συγκεκριμένε ερωτήσει. Η Ισπανία ακολούθησε τον οδικό χάρτη της προστασίας ε, για την προστασία των γιατρών ε, και την ε, πρόληψη του προσωπικού υγείας. Ο ΠΟΗ γνώριζε το ότι γίνονταν αυτές οι μεταφορές σύμφωνα με το πρωτόκολλο και σε δεύτερο επίπεδο αυτή τη στιγμή οι Αμερικανικές αρχές εργάζονται για να θέσουν σε εφαρμογή ε, να στείλουν κάποιο τρικό προσωπικό, ε, όχι ε, μόνο προσωπικό, αλλά και υλικό στις πληγήσεις περιοχές, αλλά και για να μπορέσουν ίσως να εκενώσουν κάποιους ασθενείς. Θα ήθελα να μου πείτε με την Ευρωπαϊκή Ένωση, την κυβέρνηση της Ισπανίας και την ε, Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχει κάποια συνεννόηση για να αντιμετωπίσουμε τα νέα κρούσματα. Σίγουρα οι προσπάθειες πρέπει να επικεντρωθούν στη Δυτική Αφρική, αλλά πρέπει να αποφύγουμε και τέτοια περιστατικά που ε, πραγματικά έχουν μεγάλο αντίκτυπο στην κοινή γνώμη. Υπάρχουν εγγυήσεις ασφαλείας έτσι ώστε ε, να πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις ασφαλείας και να υπάρχουν όλες οι εγγύησεις και για το εμβόλιο που βρίσκεται σε πειραματικό στάδιο. Μας ενημερώσατε πρόσφατα ότι εγκρίθηκε στην Ελβετία. Τι ξέρετε για το εμβόλιο αυτό. Υπάρχουν εγγύησεις ότι θα μπορούσε να αποτελέσει μια διέξοδο. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Κυρία Τσουίκα. Ευχαριστώ. Θέλω να ευχαριστήσω την Επιτροπή μας που οργάνωσε αυτή τη συζήτηση. Όλοι συμφωνούμε, μιλάμε εδώ για μια ανθρωπιστική καταστροφή. Ο κίνδυνος ε, είναι μικρός για την Ευρωπαϊκή Ένωση και θα ήμασταν υποκριτές να απομονώσουμε τη Δυτική Αφρική, την αιστεία της επιδημίας. Έχουμε πάρα πολλά πράγματα να κάνουμε. Ακούσαμε ότι λείπουν ε, τα χρηματοδοτικά μέσα, δεν υπάρχει απαραίτητο, το απαραίτητο προσωπικό, το απαραίτητο ιατρικό προσωπικό. Επίσης, ε, αυτό το ιατρικό προσωπικό πρέπει να καταρτιστεί και δεν υπάρχει και επαρκής ενημέρωση των πολιτών. Ακούστηκε το ποσό του ενός δισεκατομμυρίου, είναι τεράστιο το ποσό. Ταυτόχρονα ακούσαμε και ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει εκταμιεύσει 24 εκατομμύρια ευρώ για την έρευνα στην ιατρική. Βέβαια, μιλάμε εδώ ε, για πολύ μεγάλους χρόνους για την έβρεση ενός εμβολίου. Όμως εγώ θα ήθελα να μου πείτε βραχυπρόθεσμα τι μπορεί να γίνει. Κατά την άποψή μου η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει εδώ να επιδείξει μια ηγετική στάση. Θα πρέπει να δείξουμε ότι δεν θέλουμε να απομονώσουμε καμία χώρα, μόνο θέλουμε να απομονώσουμε τον ιό του έμπολα. Θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι στην ακρόαση του Επιτρόπου Στυλιανίδη ο κ. Στυλιανίδης ε, υπογράμμισε το πρώτο του επίσημο ταξίδι θα είναι ακριβώς στη Δυτική Αφρική. Είναι πολύ σημαντικό να εξαλείψουμε την αιστεία της επιδημίας. Αυτή είναι η σωστή προσέγγιση. Πρέπει να καταπολεμήσουμε τους φόβους μας, γιατί μόνο έτσι θα καταπολεμήσουμε και τον έμπολα. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Κυρία Μέισνερ. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Λέχθηκαν πολλά σχετικά με το τι πρέπει να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση για την υποστήριξη των ε, χωρών που έχουν πληγεί και έτσι δεν θα επεκταθώ περισσότερο. Πράγματι, θαυμάζω τα πρόσωπα που πηγαίνουν εκεί εθελοντικά και γνωρίζουν ότι μπορεί να μολυνθούν. Μήπως χρειάζεται να κάνουμε πολύ περισσότερα από άποψη ευρωπαϊκή, σε αυτό συμφωνώ με άλλους. Επειδή είμαι και στην Επιτροπή Μεταφορών, βρίσκω ότι είναι πολύ σημαντική η πληροφόρηση και είναι σωστό που λέχθηκε προηγουμένως ότι προετοιμάζουν ένα βίντεο για να ενημερώνουν και τους επιβάτες των αερογραμμών. De facto και εμείς όπως ενημερωθήκαμε στην Επιτροπή Μεταφορών είναι όντως χαμηλός ο κίνδυνος για την Ευρώπη, ωστόσο είναι υπαρκτός. Γι' αυτό χρειάζεται προσοχή, όχι ε, πανικός. Έχω μιλήσει εγώ με γιατρούς που εργάζονται σε γερμανικά αεροδρόμια και μου λένε ότι ναι, σκέφτηκαν αν θα πρέπει να κάνουν έλεγχο της θερμοκρασίας των ε, ταξιδιωτών, ιδίως από την Αφρική. Είπαν όμως ότι δεν είναι στην πραγματικότητα το σωστό αυτό. Μπορεί να πάει και να ελέγξει τη θερμοκρασία στο νοσοκομείο και να δουν μετά από ποια νόσο πάσχει. Βέβαια, ο πυρετός και μόνο ε, δεν είναι μεταδοτικός. Μπορεί να καταπιεί και ασπιρίνες ο ασθενής εφόσον έχει πυρετό και μετά δεν είναι μετρήσιμος πλέον. Πολύ καλύτερα είναι να εξεταστεί αν έχουν και άλλα συμπτώματα. Και οι ιατρικές ομάδες είπαν όχι μόνο πυρετός αλλά και διάρκεια και εμετή. Διότι η μετάδοση του ιού γίνεται μέσα από τα υγρά του οργανισμού. Εφόσον κάποιος είναι πραγματικά άρρωστος ή εφόσον υπάρχει μια αιτιολογημένη υποψία θα πρέπει να κινητοποιείται ένας όγκος μηχανισμός. Αυτό το θέλουμε βεβαίως, αλλά όχι αν δεν υπάρχει η απόλυτη αναγκαιότητα. Στα αεροδρόμια λοιπόν γίνεται νομίζω λογική, λογικά η διαχείριση. Τώρα για τα καράβια. Και χθε είχαμε παρουσία εκπροσώπου της ΕΜΣΑ στην Επιτροπή Μεταφορών και μας είπε ότι είχαν φτιάξει και μια ειδική ομάδα task force για να δουν ποια πλοία έρχονται με το ραντάρ μάλιστα από τη Δυτική Αφρική και μπορούν να μεταφέρουν την ασθένεια. Διαπίστωσαν όμως μετά ότι δεν είναι καν απαραίτητο διότι πρόκειται συνήθως για φορτηγά καράβια. Εξακολουθούν βέβαια να τα μελετούν τα πράγματα αυτά, ώστε να μην μεταφέρουν ούτε και αυτά κρούσματα στην Ευρώπη. Πάντως είναι πολύ χαμηλή η βαθμολόγηση που δίνουν στον κίνδυνο από την πλευρά αυτή. Βεβαίως πρέπει να δώσουμε, κυρίως αυτό είναι το σημαντικό, πολύ περισσότερη βοήθεια επιτόπου. Μπάλζο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε που μου δίνετε το λόγο. Ευχαριστώ την κυρία Διευθύντρια για τις πληροφορίες που απήντησε και σε δύο σημαντικά ερωτήματα που έχει θέσει η Κομισιόν, τι μπορεί να γίνει δηλαδή για να αντιμετωπιστεί ο κίνδυνος διάδοσης και τι μπορεί να γίνει για την ε, φροντίδα των ασθενών. Εγώ έχω και μια ακόμα ερώτηση. Τι μπορεί να κάνει ο Οργανισμός Ενωμένων Εθνών για να μην προκύψουν νέες τέτοιες επιδημίες. Απευθύνομαι δε σε εσάς, όχι μόνο υπό την ιδιότητά σας ως υπεύθυνη διευθύντρια ε, του ΠΟΗ. Τα Ενωμένα Έθνη θέλουν να δραστηριοποιηθούν παγκοσμίω υπέρ μιας ποιότητας ζωής. Πρόκειται όμως εδώ για φτωχές χώρες. Και χώρες φτωχές που έχουν μεγάλες διαφορές μεταξύ τους, δεν είναι οι ίδιες. Οι παγκόσμιοι φορείς, σε ολόκληρο τον κόσμο δηλαδή, χρησιμοποιούν με διαφορετικό τρόπο τις, ε, τους ανθρώπινους πόρους. Ακούμε ότι υπάρχουν, ε, υπάρχουν χώρες όπου ο αριθμός των γιατρών είναι ένας ανά 100.000 κατοίκους. Ένας. Θεωρεί ότι φέρει κάποια ευθύνη ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ώστε να λάβει κάποια μέτρα για να βελτιώσει την κατάσταση σε τόσο φτωχές χώρες. Να υπάρχουν περισσότεροι γιατροί και γενικότερα ε, ιατρικό προσωπικό και θεραπευτικό προσωπικό ε, σε τέτοιες χώρες. Υπάρχει δυνατότητα, υπάρχει μάλλον η δυνατότητα τα επόμενα χρόνια ξεσπάσουν και άλλες, και άλλες επιδημίες και εκεί είναι πολύ σημαντική η πρόληψη. Έχετε σχέδια σχετικά. Κυρία Γιούτλαντ. Ευχαριστώ πολύ που είχαμε τη δυνατότητα να κάνουμε αυτή την τόσο σημαντική συζήτηση. Ευχαριστώ και την κυρία Γιάκαμπ. Ήταν πολύ καλή η εισαγωγή της και μας περιέγραψε την κατάσταση με σαφήνεια. Τώρα, Όποιος όμως βλέπει την κατάσταση διαπιστώνει ότι οι πόροι είναι ανεπαρκείς. Χρειάζεται ευέλικτη χρηματοδότηση, κρεβάτια, νοσηλευτικό προσωπικό και φυσικά συμμερίζομαι την ανησυχία και απογοήτευση και άλλων συναδέλφων ότι δεν δίνουμε αρκετή βοήθεια ως Ένωση, αρκετή στήριξη. Δεν κάνουμε αρκετά όλοι από κοινού ως Ένωση. Οπότε θα ήθελα η κυρία Γιάκαμπ να μου πει τι αλλαγές πιστεύει ότι μπορούν να, να γίνουν ως προς τα εξής τρία. Πρώτον, πώς θα σταματήσουμε την αλυσίδα μετάδοσης. Είπατε ότι χρειάζονται περισσότεροι πόροι. Εντάξει, αλλά τι μπορούμε να κάνουμε εμείς για να ασκήσουμε πίεση στα κράτη-μέλη για να σταματήσει η μετάδοση της νόσου. Δεύτερον, Επίσης πολύ προωθημένη βοήθεια γενικότερα για τις κοινωνίες που πλήττονται. Και άλλοι συνάδελφοι ε, εξήγησαν τις ευρύτερες επιπτώσεις που έχει για τα ευάλωτα άτομα, για τις εγγύους, για τους ασθενείς από άλλες ασθένειες όπως η ελονοσία που δεν ε, λαμβάνουν ε, την φροντίδα που χρειάζονται. Τι μπορεί να κάνει η Ένωση γι' αυτό γιατί είναι καταστροφή η οποία θα χτίσει πάνω ε, σε αυτά που έχει ήδη προκαλέσει η προηγούμενη καταστροφή. Επίσης, αυτό το εμβόλιο, η ελπίδα για εμβόλιο που μπορεί να το έχουμε διαθέσιμο τον επόμενο Ιανουάριο. Αλλά νομίζω ότι πρέπει να ε, βγάλουμε διδάγματα από τα λάθη που έχουμε κάνει στο παρελθόν, σε προηγούμενες περιπτώσεις. Όταν υπάρχει αυτή η έντονη πίεση των ε, μέσων μαζικής ενημέρωσης, προσπαθούμε να κάνουμε κάτι, μετά που απομακρύνεται σταματάμε. Θέλουμε να μας πείτε εσείς τι πιστεύετε ότι πρέπει να κάνουμε, ώστε να μην ξεχαστούν τα θέματα αυτά, να συνεχίσουμε να ασχολούμεθα και όταν θα σταματήσουν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Πίερκα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ που έχω δυνατότητα και από πλευρά της ε, ομάδας μου να σας πω ε, την άποψή μας. Κοιτάξτε, κάθε επιδημία έχει μία πορεία. Ξεκινάει, κάποια στιγμή φτάνει σε ένα μέγιστο και μετά σιγά σιγά ε, αδυναμ μειώνεται η έντασή της και σταματάει. Θα ήθελα να μας πει κυρία Γιάκομπ σε ποια φάση είμαστε τώρα. Είμαστε τώρα στο μέγιστο ή είμαστε ήδη στην καθοδική καμπύλη. Είμαστε ήδη σε φάση μείωσης της ε, επιδημίας. Υπάρχουν πολύ ακραίες ε, απόψεις για το τι ε, σημασία έχει αυτή η επιδημία. Υπάρχει και πολύ πανικός. Ίσως όμως ε, να μην αντιμετωπίζουμε σωστά αυτή την επιδημία. Διότι ξέρετε ότι πολλές φορές υπάρχει λαϊκιστική αντιμετώπιση και γι' αυτό θέλω να κάνω μία ερώτηση προς τους εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Οργανισμού Φαρμάκων. Η έρευνα ε, για τα εμβόλια γίνεται με το σωστό ρυθμό. Παρακολουθούμε τις δυνατότητες μεταλλαγής του ιού ή είναι πολύ αυξημένες. Γιατί η έρευνα πρέπει να παρακολουθεί και αυτές τις δυνατότητες, αλλιώς δεν έχει έννοια. Οπότε η ερώτηση. Υπάρχει συντονισμένη προσπάθεια του Οργανισμού Φαρμάκων και του Αμερικανικού Ομοσπονδιακού Οργανισμού Φαρμάκων FDA για να καταλήξουμε σε ένα σωστό εμβόλιο. Ξέρω πολύ καλά ότι είναι πάντα δύσκολο να αντιμετωπιστούν. Οπότε είναι πολύ σημαντικό να είναι και η έρευνα στο αντίστοιχο επίπεδο και επίπεδο συντονισμού. Και κάτι άλλο για τον πανικό που έχει προκύψει. Μήπως κάναμε τα λάθη που κάναμε και κατά τον, ε, την γρήπη των χείρων, όπου καταλήξαμε σε παραγωγή πολλών εμβολίων, τα οποία μετά χρειάστηκε να καταστρέψουμε με μεγάλο κόστος όλα αυτά. Επαναλαμβάνω λοιπόν. Σε ποιο σημείο είναι η επιδημία, έχει φτάσει στο μέγιστο, έχει αρχίσει να μειώνεται η έντασή της. Και δεύτερη ερώτηση, η έρευνα για να βρούμε ε, ε, εμβόλιο γίνονται με σωστή συνεργασία. Άλλους δύο μιλητές έχουμε. Η κυρία Εύη είναι η πρώτη. Ευχαριστώ διάδοση του διευκολύνεται από κάποιους παράγοντες όπως η μαζίκωση των δασών. Ε, εδώ λοιπόν πρέπει να σκεφτούμε την εκμετάλλευση των φυσικών πόρων και πώς πρέπει να γίνεται. Όμως υπάρχει και άλλη μια πτυχή, η κατανάλωση του μπουσμιτ, δηλαδή του θυράματος, Έχουμε κάποια ζώα που μπορεί να έχουν μολυνθεί ε, είτε ε, αν έχουν, ε, έχουν καταναλωθεί κάποια φρούτα που έχουν δαγκώσει νυχτερίδες και είναι δυνατό στη θεραπεία να σκεφτούμε κάποιους τρόπους πρόληψης, δηλαδή να χρησιμοποιήσουμε και κάποια προγράμματα ενημέρωσης για τους πληθυσμούς που εκτίθενται σε αυτή την όσο. Σας ευχαριστώ. Και τέλος, ο κύριος Τούρμπες. Ευχαριστώ. Επανέρχομαι σε κάτι που είπε η κυρία Ριβασί. Χρειαζόμαστε περισσότερη οργή και περισσότερη δράση. Μάλιστα, το πρόβλημα λοιπόν εντοπίζεται εκεί επί τόπου. Όσοι από εμάς έχουμε σχέση με επαφές με τους γιατρούς του κόσμου ή τους γιατρούς χωρίς σύνορα, γνωρίζουμε ότι τα πράγματα είναι πολύ χειρότερα. Γι' αυτό παρακαλώ κύριε Πρόεδρε σε κάποια επόμενη συνεδρίαση θα υποβάλουμε και επίσημα το αίτημα να προσκληθούν και ε, ε, εκπρόσωποι των γιατρών χωρίς σύνορα. Άνθρωποι που δηλαδή είναι πολύ πιο κοντά στην αιστεία και όχι άνθρωποι που προσπαθούν να συγκαλύψουν λάθη που έχουν κάνει από την αρχή. Προεβδομάδος με ρώτησε ένας δημοσιογράφος. Τι γίνεται, εάν Δεκέμβρη, Γενάρη, Φεβρουάριο, Μάρτι ξεσπάσει επιδημία γρήπης στην Ευρώπη. Βρισκόμαστε στην εποχή, ζούμε στην εποχή της πλήρης, πλήρους κυριαρχίας του διαδικτύου. Οι, οι ειδήσει διαδίδονται μέσα από το διαδίκτυο με αστραπία ταχύτητα. Πώς είστε προετοιμασμένοι, πώς είμαστε προετοιμασμένοι για ένα οποιοδήποτε γεγονός το οποίο μπορεί να ξεσπάσει την Ευρώπη και να διαχυθεί μέσω ίντερνετ με τεράστια ταχύτητα. Δεν πρέπει να έχουμε κάποια προετοιμασία για ένα τέτοιο ξέσπασμα ενός κύματος πανικού διότι οι εφημερίδες πλέον και οι ειδήσει της τηλεόρασης που ε, βγαίνουν στις 8 το βράδυ είναι πλέον για τους γέροντες. Οι ενημέρωση σήμερα γίνεται μέσα από το διαδίκτυο. Πώς έχετε προετοιμαστεί για ενδεχόμενο ξέσπασμα κύματος πανικού από, την, από το διαδίκτυο. Ο κύριος Γραμματικάκης έχει ζητήσει ακόμη το λόγο. Είμαι τελευταίος, ελπίζω θα είμαι πολύ σύντομος. Εξάλλου λέει το βιβλικό ρητό «Η έσχατη έσονται πρώτοι». Εγώ πολύ ευχαριστήθηκα κύριε Πρόεδρε και σας συγχαίρω από την ε, εμπεριστατωμένη τα έλεγα σημερινή παρουσία. Καλό θα ήταν να είναι και μερικοί γιατροί χωρίς σύνορα. Δεν μπορούμε να τα έχουμε όλα και ιδιαίτερα από την παρουσία της Προέδρου της ΠΟΗ. Και θα είμαι πάρα πολύ σύντομος. Θέλω αν γίνεται να διαβεβαιωθώ ακόμα μια φορά γιατί είναι πολύ ωραία η διαπίστωση ότι είμαστε σε καλή φάση ότι οι ευρωπαϊκές χώρες, οι 28, έχουν την απαραίτητη τεχνογνωσία για να αντιμετωπίσουν τον ιό και ιδίω οι χώρες που υφίστανται αυτή τη στιγμή μια άδικη κατά τη γνώμη μου οικονομική κρίση όπως για παράδειγμα η Ελλάδα που έχει ισοπεδώσει ένα μεγάλο μέρος από το σύστημα υγείας. Η δεύτερη παρατήρησή μου γιατί δεν άκουσα τίποτα πάνω σε αυτό είναι ότι ενδεχομένως αυτός ο ιός, αυτή η φοβερή επιδημία να δημιουργήσει και δευτερευόντως κύματα ή φαινόμενα ρατσισμού απέναντι στις αφρικανικές ή στις φτωχές χώρες και γι' αυτό πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Και θέλω να τονίσω κι εγώ, υπόθηκε και από άλλους συναδέλφους, ότι πρέπει να βγάλουμε διδάγματα για το μέλλον από αυτή την κρίση. Διδάγματα από την αργοπορία μας, διδάγματα ίσως από την έλλειψη αλληλεγγύης προς τις φτωχές χώρες, διδάγματα για τους εαυτούς μας και τους άλλους. Ευχαριστώ πολύ. Thank you very much. And now... Ευχαριστώ πολύ. Και τώρα θα δώσω το λόγο στην ε, κυρία Γιάκαπ για να απαντήσει. Σίγουρα δεν ε, είναι πολύ εύκολο να απαντήσετε σε όλες αυτές τις ερωτήσεις. Παρακαλώ. Πρώτα, ευχαριστώ για τη θαυμάσια συζήτηση. Βεβαίως οι ανησυχίες σας είναι δικαιολογημένες. Ας αρχίσω με το τελευταίο. Η ανησυχία σας είναι 28 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η δική μου ανησυχία είναι οι 53 της περιφέρειάς μας που περιλαμβάνει και την ε, Ρωσία και τη Ρωσία και άλλες χώρες. Ε, και εγώ βέβαια ηγούμε της ευρωπαϊκής περιφέρειας του ΠΟΗ με έδρα στην Κοπενχάγη. Πολλοί από το προσωπικό μου όμως βρίσκονται στη Δυτική Αφρική, όπως και το δεξί μου χέρι που είναι επικεφαλής του τμήματος μολυντικών νόσων μολυσματικών συγγνώμη, νόσων που είναι στην Ουινέα τώρα. Και έχουμε από πρώτο χέρι λοιπόν πληροφορίες. Άρα αυτά που σας λέω δεν προέρχονται από τον ελεφάντινο πύργο μας στην Κοπενχάγη αλλά από επιτόπου παρατήρηση. Για την Ευρωπαϊκή Ένωση εξακολουθώ να πιστεύω ότι ο κίνδυνος ε, διάδοσης της ε, επιδημίας είναι χαμηλός. Πρέπει όμως να διδαχθούμε από κάθε περίπτωση και από την ισπανική περίπτωση και να δούμε τι πρέπει να γίνει. Γιατί όπως είπα και πριν και σε πολλές άλλες δηλώσεις που έχω κάνει, αυτό που με απασχολεί και με ανησυχεί πάντοτε είναι ότι κάθε φορά που εφαρμόζεται ένα πακέτο λιτότητας, οι πρώτες που πέφτουν θύματα είναι οι υπηρεσίες υγείας. Εξετάζοντας μόνο τις ευρωπαϊκές χώρες, διαπιστώνουμε ότι για πρόληψη από όλο τον προϋπολογισμό της υγείας, για την πρόληψη καταβάλουμε μονάχα το 3%. Ένας από τους τομείς λοιπόν όπου το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ιδίω η Επιτροπή σας μπορεί να βοηθήσετε είναι να διασφαλίσετε ότι θα υπάρξει μεγαλύτερη επένδυση δημοσίων πόρων στην πρόληψη, ότι θα εντοπιστούν τα κενά στην ετοιμότητα των χωρών μελών της Ευρώπης και ότι θα καλυφθούν. Σήμερα είναι ο ιός της έμπολα. Αύριο μπορεί να είναι ο ιός κορώνα από την Μέση Ανατολή και ούτω καθεξής. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι, πρέπει να έχουμε τις απαραίτητες δυνατότητες που προβλέπονται και στη διεθνή νομοθεσία. Και ασφαλώς δεν έχουμε φτάσει ακόμη στο επίπεδο αυτό. Αυτό είναι από τα πράγματα που πρέπει να έχουμε υπόψη μας, κύριε Πρόεδρε. Συνολικά συμφωνώ μαζί σας και νομίζω αυτό είπατε άλλωστε και εσείς, ότι οφείλουμε να ελέγξουμε στην πηγή την κρίση. Ακόμα μας ξεφεύγει. Προηγείται η επιδημία και ερχόμαστε εμείς από πίσω και προσπαθούμε. Γι' αυτό και κάνουμε μεγάλη προσπάθεια να επιταχύνουμε τη διεθνή αντιμετώπιση και να εξασφαλίσουμε ώστε να αντιμετωπιστούν όλες οι ανάγκες που προβλέπουν οι σχετικοί οδικοί χάρτες. Έχουμε μόνο 15 κέντρα, όπως είδατε και ε, στο ε, πίνακα. Χρειαζόμαστε διεθνές προσωπικό. Έχουμε μόνο 150 από τους 750 που χρειαζόμαστε. Χρειαζόμαστε και πολύ περισσότερους στις χώρες μέλη, εθνικό προσωπικό δηλαδή. Και πρόκειται πραγματικά για ανθρωπιστική κρίση άνευ προηγουμένου, έχει ένα καταβήγοντα χαρακτήρα άνευ προηγουμένου και γι' αυτό ο ΠΟΗ ηγείται βεβαίω, αλλά ολόκληρη η οικογένεια των οργανισμών του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών δηλαδή συμμετέχουν. Αντιμετωπίζουν βεβαίω και πολιτιστικά θέματα όπως τις κηδείε και ταφή που είναι πολύ σημαντικό η αξιοπρεπή ταφή. Κινούμεθα προς σωστή κατεύθυνση αλλά δεν έχουμε φτάσει ακόμα του στόχου μα. Δύο πράγματα που είναι πολύ σημαντικά. Το ένα είναι να απομονώσουμε τις ε, νόσους και το άλλο είναι να προσφέρουμε θεραπεία, φροντίδα για αυτούς που έχουν μολυνθεί. Εκεί όμως χρειαζόμαστε την πλήρη συμμετοχή των τοπικών κοινοτήτων αλλά και ε, διεθνές προσωπικό. Χαίρομαι που η κυρία Ριβασί έθεσε το θέμα που εμφανίζεται συχνά άλλωστε και στα μέσα μαζικής ε, ενημέρωσης. Υπήρξε καθυστέρηση στην ανταπόκριση των ΗΠΑ και του ΠΟΗ. Η απάντησή μου είναι όχι. Ανακοινώσαμε στις 8 Αυγούστου ότι υπάρχει κατεπίγουσα κατάσταση σύμφωνα με τους κανονισμούς, αλλά τους προηγούμενους μήνες ήμασταν ήδη επιτόπου. Τον Μάρτι είχαμε ε, αναγάγει σε επίπεδο ε, υπερθμών 2 και Μάιο, όχι, Απρίλιο-Μάιο και Απρίλιο-Μάιο στείλαμε 110 δικούς μας από το προσωπικό μας επιτόπου, κυρίως από την Αφρικανική περιφέρεια, η οποία επίσης πολύ έχει επικριθεί, αλλά χωρίς να υπάρχει πραγματικός λόγος. Είναι αλήθεια ότι η επικοινωνία μας ήταν ελληματική και δέχομαι την κριτική αυτή, αλλά δεν νομίζω ότι κάναμε κάποιο σοβαρό λάθος και ότι καθυστερήσαμε να ανακοινώσουμε το ξέσπασμα της επιδημίας. Στις 8 Αυγούστου αυτό απαιτούν άλλωστε οι διεθνείς κανονισμοί, τα είπαμε. Αυτό έκανε και η Emergency Committee που ε, το σύστησε στον Γενικό μας Διευθυντή. Βεβαίως χρειάζεται να κάνουμε κάποια αξιολόγηση για τα διαβήματά μας αυτά. Και όταν θα μπορέσουμε να συγκρατήσουμε την επιδημία θα κάνουμε και την αξιολόγηση αυτή. Υπάρχουν όμως ε, μηχανισμοί υπάρχουν ρυθμίσεις. Θα θυμάστε ίσως κυρία Ρίβαζη ότι και με την άλλη επιδημία Α1 ή τα 1 που ε, είχαμε κάνει πολύ μεγάλη προσπάθεια και μετά εμείς βιαστήκαμε πάρα πολύ και χρειάστηκε πάλι τότε να υπερασπιστούμε την ε, στάση μας. Είχαμε και την Επιτροπή για τον ιό αυτό, είχαμε και συζητήσει με όλες τις χώρες μέλη, το ίδιο θα πράξουμε και τώρα, σας βεβαιώνω. Αλλά Τώρα κυρίως θέλουμε να στοχεύσουμε και να συγκεντρώσουμε όλες μας τις προσπάθειες στην προσπάθεια αντιμετώπισης δηλαδή της κρίσης αυτής. Ορισμένα από τα θέματα τώρα που θέσατε και σας ευχαριστώ και πάλι συμφωνούμε νομίζω όλοι ότι χρειάζεται να δώσουμε όλη την έμφαση στις χώρες της Δυτικής Αφρικής και αυτό κάνουμε. Κατά την άποψή μου η λιτότητα δεν θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί ως πρόφαση για να αποδυναμωθούν οι υπηρεσίες δημόσιας υγείας. Το ίδιο πρέπει να κινητοποιηθούν οι δωρητέ για τη βοήθεια από δυτικές αφρικανικές χώρες. Δεν αρκεί μονάχα η επένδυση σε ειδικά προγράμματα και εμβολιασμού κλπ. Χρειάζεται και άλλα στοιχεία. Για τη Δυτική Αφρική ένα πρόβλημα ήταν και ο εμφύλιος πόλεμος ένας βαρύτατος εμφύλιος πόλεμος ο οποίος αποδυνάμωσε τις χώρες αυτές, τις υποδομές τους, τα συστήματα υγείας τους. Πολλοί γιατροί έφυγαν από τις χώρες αυτέ αυτές και τώρα μόλις έχουμε αρχίσει να ε, ενδυναμώνουμε τα συστήματά τους, αλλά όταν άρχισε ο, ε, η επιδημία έμπολα. προχωρούμε λοιπόν σε αποκατάσταση των συστημάτων υγείας τους για το ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νομίζω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έπαιξε πολύ θετικό και επικοδομητικό ρόλο. Με δύο τρόπους. Αφενός για να προστατεύσει βεβαίως τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά επίσης για να συνεισφέρει στις προσπάθειες στη Δυτική Αφρική. Σε ό,τι αφορά την προστασία των Ευρωπαίων πολιτών, συμφωνώ με τα όσα είπε ο Τζον Ράιν, ότι οι τακτικές συνεδριάσεις της Health Security Committee και σε επαφή με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας είναι πολύ σημαντικές. Το ίδιο βεβαίως η Ιταλική Προεδρία που έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο όχι μόνο για τη συζήτηση των θεμάτων στο Συμβούλιο Υπουργών αλλά μάλιστα συγκάλεσε και έκτακτη συνεδρία των Υπουργών Υγείας για να συζητήσουν αν χρειάζονται exit screening, δηλαδή ε, έλεγχος των, των ε, ταξιδιωτών που φεύγουν και μάλιστα και Συμβούλιο, Επιτροπή και ε, με μένα συμμετοχή και δική μου συζητήσαμε τα θέματα αυτά. Και για το βίντεο. Επίσης οι χώρες μέλη της Ένωσης έπαιξαν σημαντικό ρόλο στην προσφορά πόρων και στήριξης στους δικούς χάρτες του ΠΟΗ και των Ηνωμένων Εθνών και σας ευχαριστώ και πάλι. Στην τελευταία συνεδρίαση, αν θυμούμε καλά, ανακοινώθηκαν 180 εκατομμύρια ευρώ που θα χρηματοδοτήσουν τον οδικό αυτό χάρτη από πλευρά ευρωπαϊκών χωρών μελών. Χρειαζόμαστε ακόμα περισσότερο. Ακόμα περισσότερα και χρήματα και προσωπικό. Το προσωπικό είναι το κλειδί. Αλλά τα κέντρα θεραπείας τώρα σιγά σιγά στείνονται. Θα είδατε και πέραν των 15 που ήδη έχουν ε, δημιουργηθεί, στείνονται τώρα σιγά σιγά άλλα 20 και ελπίζουμε ότι θα μπορέσουν να είναι λειτουργικά σύντομα που θα προσφέρουν 5.000 κλίνες παραπάνω από αυτές που ήδη υπάρχουν. Εκεί που χρειάζεται να κάνουμε μεγαλύτερη προσπάθεια είναι να στείλουμε περισσότερο διεθνές προσωπικό στις χώρες αυτές, επιτόπου. Για να γίνει αυτό όμως πρέπει να προσφέρουμε και την ασφάλεια στο προσωπικό αυτό, ότι εάν αντιμετωπίσουν πρόβλημα, αν μολυνθούν δηλαδή, θα μπορέσουν να τύχουν τη φροντίδα που είναι απαραίτητη και επιτόπου και ενδεχομένως να επαναπατριστούν. Ισπανία. Νομίζω ότι θα είναι ευκολότερο για όλους αν μπορούν τα πρόσωπα αυτά να ε, λάβουν την απαραίτητη φροντίδα υψηλής ποιότητας επιτόπου που αυτή τη στιγμή δεν είναι δυνατόν. Αλλά με την ενίσχυση των υποδομών εκεί στις δυτικοαφρικανικές χώρες πιστεύουμε ότι θα υπάρξει περαιτέρω ικανότητα αντιμετώπισης των κρουσμάτων αυτών. Και βεβαίως και ο ιατρικός επαναβατρισμός που είναι πάρα πολύ σημαντικός μέχρι τώρα στην περίπτωση αυτή βέβαια θα, μειωθούν, ε, ε, θα μειωθεί ανάγκη να, να γίνεται προσφυγή σε αυτόν έρθω και σε μερικά άλλα θέματα. Ένα άλλο θέμα ήταν τα εμβόλια. Πολλοί από εσά αναφερθήκατε σε αυτό. Όπως είπα, προς στιγμή βασιζόμαστε στα μέτρα δημόσιας υγείας, απουσία εμβολίων και άλλη θεραπεία. Όμως ε, το καλό με τη σημερινή κατάσταση είναι ότι συνεχίζεται η έρευνα και η ανάπτυξη για την ανάπτυξη αυτού του εμβολίου. Αυτό δεν ίσχυε στο παρελθόν, γιατί όπως γνωρίζετε μέχρι τώρα τα εμπορικά κινήτρα δεν υπήρχαν. Και αυτό είναι το δεύτερο θέμα κύριε Πρόεδρε. να ξέρω ότι πρέπει να είμαι σύντομη. Αυτό είναι το δεύτερο θέμα λοιπόν ε, που θέλω να σας ε, ε, ζητήσω να με υποστηρίξετε. Δηλαδή για όλες τις ε, ασθένειες που είναι παραμελημένες, για όλες τις ασθένειες της φτώχειας, να βρούμε κάποιο μηχανισμό όπου μπορεί να προχωρήσει η έρευνα και η ανάπτυξη. Γιατί αυτό ε, ήλθε στο προσκήνιο μόνο όταν η ΕΠΑ, η Ευρώπη και άλλες ε, προηγμένες χώρες επλήγησαν. Οι προκλήνικες δοκιμές του εμβολίου είναι στο πρώτο στάδιο, ολοκληρώνεται τώρα το πρώτο στάδιο για την ασφάλεια του εμβολίου. Η ασφάλεια είναι το κύριο θέμα. Στο δεύτερο στάδιο εξετάζουμε την αποτελεσματικότητα του εμβολίου και κάποιοι ε, που έχουν μολυνθεί με την ε, σύμφωνη γνώμη τους ε, θα δοκιμάσουν ε, το εμβόλιο αυτό και αν όλα πάνε καλά φυσικά θα μπορέσει να διαδοθεί στη συνέχεια το εμβόλιο. Φυσικά αυτό είναι ένα θέμα που παραμένει να το δούμε. Και κατόπιν πρέπει να συμφωνήσουμε επί των κριτηρίων για το ποιος θα εμβολιαστεί. Όταν θα είναι διαθέσιμα τα εμβόλια βέβαια. Να αναφερθώ και σε κάποια άλλα ζητήματα όπως η μετανάστευση. Θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό το μεταναστευτικό κίνημα, ε, έχουμε μεγάλη συνεργασία με τις χώρες του Ευρωπαϊκού Νότου, πολλοί μετανάστες προέρχονται από όλες χώρες, όχι από τις τρεις πληγικές χώρες και περισσότεροι είναι υγιείς μετανάστες. Αυτό είναι ένα θέμα επί το οποίο πρέπει να συνεργαστούμε για να βρούμε πώς θα αντιμετωπίσουμε τις υγειονομικές ανάγκες των μεταναστών, αλλά από τη σκοπιά του έμπολα δεν θα συνέστηνα εγώ κάποια συγκεκριμένα μέτρα για τους μετανάστευς και σίγουρα όχι να ελέγξουμε τις κινήσεις του. Τα μέτρα που είδατε στις διαφάνειες ισχύουν για όλους όσους μπαίνουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κύριε Αντιπρόεδρε, σας ευχαριστώ που θίξατε το θέμα των διδαγμάτων. Ναι, φυσικά πρέπει να μάθουμε από όλα αυτά. Θα τα ξελογίσουμε. Δύο θέματα εδώ είναι σημαντικά. Καταρχήν, πρέπει να ενδυναμώσουμε τα συστήματα υγείας στην Αφρική, το είπατε, και όλα τα ειδικά προγράμματα νόσων πρέπει να είναι ολοκληρωμένα και επίσης θα πρέπει να οικοδομήσουμε όλες τις ε, ικανότητες που δεν υπάρχουν στις ευρωπαϊκές χώρες αλλά στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα έλεγα ότι ισχύουν αυτές οι κύριες ε, ικανότητες Ενισχύω κυρίως για τις χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα έλεγα ότι οι προσπάθειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης επαρκούν. Αυτό ανέκυψε πολλές φορές. Φυσικά πάντοτε μπορεί να γίνει κάτι παραπάνω, αλλά νομίζω ότι για την προστασία των Ευρωπαίων πολιτών βεβαίω και υπάρχουν μέτρα. Τώρα, ω προ τη Δυτική Αφρική, θα ήθελα να ενθαρρύνω τι ευρωπαϊκέ χώρε ε, και τι χώρε τη Ευρωπαϊκή Ένωση να παράσχουν περισσότερη υποστηρίξη στον οδικό χάρτη. Ναι, ναι, τελειώνω. Απλώ ήταν πολλέ οι ερωτήσει και φυσικά να απαντήσω συνολικά θετικά. Τώρα για το θέμα του θυράματος που θεωρήσα ότι είναι πολύ σημαντικό. Αυτό είναι ένα κύριο ζήτημα. Πρέπει να γνωρίζετε ότι αυτές οι χώρες είναι πολύ φτωχές ε, και όταν ε, οι άνθρωποι μπαίνουν στην απομόνωση πολλές φορές ε, δεν έχουν τροφή. Έτσι λοιπόν ένα θέμα που πρέπει να λύσουμε είναι και το στοιχείο της επιστηστικής ασφάλειας. Χρειαζόμαστε πρόσθετους πόρους όπως ευέλικτη χρηματοδότηση. Το είχα και αυτό κατά νου, γιατί πρέπει να δώσουμε και τρόφιμα στους ανθρώπους αυτούς. Και ένα ακόμη θέμα, και θα σταματήσω, για τη γρήπη. Ε, υπάρχουν ε, πάρα πολλοί λανθασμένοι συνεγερμοί. Είχαμε μια παγκόσμια συνάντηση στο Τζιμπετζάν πρόσφατα. Ήθελα να, να την ακυρώσουν, αλλά είπαμε όχι, ας προχωρήσουμε και είχαμε ε, ε μια, ένα κρούσμα που τελικά ήταν ελαιονοσίας. Και τώρα βλέπετε ε, είναι πολύ σημαντικό να έχουμε και τα εμβόλια κατά της γρήπης για να προστατεύσουμε τους αυτούς μας αλλά και για να ε, μειώσουμε αυτές τις δυνατότητες των λαθασμένων ε, συναγερμών και φυσικά και οι άλλες νόσοι που αφορούν τη Δυτική Αφρική αφορούν τη Δυτική Αφρική γιατί τώρα Δίνουμε όλοι μας την προσοχή στον εμπολά, αλλά πολύ λίγη προσοχή προς τις άλλες νόσους. Όπως το χάρη την ασφαλή εγκυμοσύνη, του ασφαλείς ε, τοκετούς, ε, χρόνες νόσους, τη φροντίδα μητέρας και παιδιού. Πολύ λίγη προσοχή δίνεται και είναι πάρα πολύ μικρή η ικανότητα των χωρών αυτών. Ζητώ συγγνώμη που μακρηγόρησα, Πρόεδρε, και ζητώ συγγνώμη αν δεν απαντήσα σε όλες τις ερωτήσεις, αλλά ολοκληρώνω εδώ. Πρόεδρος, θέλω να ευχαριστήσω την ε, διευθύντρια του ΠΟΗ για την περιοχή της Ευρώπης. Και να σας πω ότι εδώ ολοκληρώνονται υπηρεσίες διερμηνίας και αν ε, χρειάζεται πράγματι θα δώσω το λόγο στην Κομισιόν στους εκπροσώπους των δύο οργανισμών τηλεγραφικά. Η Κομισιόν λέει όχι. Αν πούν όχι και οι εκπρόσωποι των οργανισμών, α, μάλιστα από το Κέντρο Πρόληψη και Ελέγχου Θέλετε να νόσων τηλεγραφικά, αν μπορείτε να μα απαντήσετε στην ερώτηση που τέθηκε. Ναι, θα ήθελα να αναφέρω ότι μπορούμε να μειώσουμε τον κίνδυνο στην Ευρώπη στο μηδέν, ε, μόνο απομονώντα τη Δυτική Αφρική. Όμω εκεί χρειάζεται, ε, χρειάζεται ιατρικό προσωπικό και πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι. Καταρχήν πρέπει να εγγυθούμε ότι μπορούν να επιστρέψουν στην Ευρώπη, ότι τα νοσοκομεία είναι έτοιμα. Και εκεί εγώ θα εστίαζα τι προσπαθίε μου. Ευχαριστώ. Πρόεδρος, θέλω να ευχαριστήσω ε, όλους τους ε, βουλευτές ε, και τη Γραμματεία. Πρόεδρος, ευχαριστώ και τους διερμηνείς. Ευχαριστούμε και εμείς και θα τα πούμε σήμερα το απόγευμα για την επόμενη συνεδρία της Επιτροπής μας.